Το πρώτο μας θέμα είναι η προετοιμασία της ε, Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17-18 Μαρτίου και η συζήτηση για τη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και για πολύ καιρό συνάδελφο, την κυρία Χένις Πλασάρτ. Καλώς ήλθατε κυρία Υπουργέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Λυπάμαι κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ως ε, παλαιό μέλο έχετε την ε, δυνατότητα να μιλάτε από το αναλόγιο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να αναφερθώ σε εσά εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 17η-18η Μαρτίου, που θα ασχοληθεί με οικονομικά θέματα, αλλά κυρίω με τα θέματα μετανάστευση. Φυσικά, θα ήθελα να αναφερθώ και στα αποτελέσματα τη συνάντηση τη Δευτέρα των αρχηγών κρατών και κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα για τη μετανάστευση. Στις συνεχείς προσπάθειές μας να σταματήσουμε τι προσφυγικέ προσφυγικές η Δευτέρα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Έγινε πρόοδο. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε ευρωπαϊκές λύσεις στην κρίση. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως τονίστηκε και από τον πρόεδρο Τάσκ όταν μίλησε ενώπιον τη Ολομέλεια. Η μόνη λύση είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Η συνάντηση της Δευτέρας ήταν μια πολύ επίκαιρη ευκαιρία να κάνουμε μια ανασκόπηση της, ε, του θεματολογίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και να δούμε μέχρι πού έχουμε φτάσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σαφείς ότι η πρόοδο στην εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης. Αν θέλουμε όμως να σταματήσουμε την μεταναστευτική ροή, πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες και από τι δύο πλευρές να κλείσουν οι δρόμοι μετανάστευσης και να κατασταθεί το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών. Μέσα στα πλαίσιο, στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσει Τουρκίας είναι καλόδεκτες. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε επί τη βάση ορισμένων αρχών. Πρώτον, η επιστροφή όλων των νέων παράτυπων μεταναστών που διασχίζουν την, το Αιγαίο προς τα ελληνικά νησιά από την Τουρκία. Δεύτερον, επιτάχυνση της διαδικασίας για τη χορήγηση ε, εξαίρεσης από την ανάγκη προξενικής θεώρησης. Τρίτον, την ταχύ εκταμείευση των 3 δισεκατομμυρίων και πρόσθετα χρήματα για τους, μετανάστε, για τους πρόσφυγες στη Συρία. Τέταρτον, προετοιμασία για το άνοιγμα νέων κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέμπτον, τη δυνατότητα να δημιουργηθούν στη Συρία περιοχές οι οποίες θα είναι ασφαλείς. Έκτο και τελευταίο, το να επαναγκατασταθούν οι πρόσφυγες από τη Συρία με τη βάση του ένας για ένα. Προφανώς κύριε Πρόεδρε χρειάζονται περισσότερα πράγματα να συμφωνήσουμε με την Τουρκία επί τη βάση των προτάσεών τους και ο πρόεδρος Τούσκ θα εξασφαλίσει ότι θα συνεχιστούν αυτές τις προσπάθειες μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην 17η και 18η Μαρτίου. Αν τηρήσει τα υπεσχημένα η και 18 η μαρτιου αν τη τα υπεσχημενα η τουρκια να πάρει όλους τους μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στις ελληνικές ακτές, έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε το έργο των διακινητών και να σταματήσουμε μια ανθρώπινη τραγωδία η οποία λαμβάνει χώρα στο Αιγαίο. Θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε την τωρινή άτακτη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση με ένα ε, οργανωμένο μηχανισμό ε, προσφύγων. Είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι έχουμε επιτύχει όπως και για πολλά άλλα θέματα, όλα εξαρτώνται από την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Αν μπορέσουμε όμως το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να περατώσουμε τη συμφωνία με την Τουρκία, αυτό θα είναι μια δυνατή, μια δυνητική μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι μονάχα ένα στοιχείο τη κοινή μα στρατηγική. Πέραν των σχεδίων μα με την Τουρκία, έχουμε και τη συνεργασία με τρίτε χώρε που είναι κομβική και θα πρέπει να, είναι, να συνεχίσει να είναι κομβική για να εμποδίσει του ε, μετανάστε οι οποίοι κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προ την Ευρώπη. Προφανώ το να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών μα συνόρων παραμένει μια προτεραιότητα για μα. Το έργο του Συμβουλίου για μια πρόταση για μια δύναμη η οποία θα ελέγχει τα σύνορα τη Ευρώπη και ακτοφυλακή για, τις, ε, για τα θαλάσσια σύνορα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχετε εσείς ήδη να συζητάτε αυτή την πρόταση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και εμείς προσβλέπουμε στην συνεργασία μαζί σας ώστε αυτό το σύστημα να γίνει το ταχύτερο δυνατό λειτουργικό. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε μια πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου μέχρι τον Ιούνιο. <clears throat> Χθε είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον συζητή σας τον κύριο Παύλη και βλέπω ότι υπάρχει πραγματικά θέληση και από τις δύο πλευρές για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κύριε Πρόεδρε, να στραφώ τώρα στην κατάσταση κατά την... στο μήκος του δρόμου των Δυτικών Βαλκανίων έχουμε συμφωνήσει στο, στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει εν καιρό όλοι να επανέλθουν στον κώδικα του Σέγγεν. Έχει σταματήσει η ροή στα Δυτικά Βαλκάνια, δεν υπάρχει πια αυτή η διαδικασία που περνούν ελεύθερα, αλλά είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην εφαρμογή των κανόνων του Σέγγεν. Αυτό είναι δύσκολο, υπάρχουν ε, συνέπειες που έχουν προκύψει οι οποίες απαιτούν ταχεία δράση. Αν θέλουμε να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική δράση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα δώσουμε βοήθεια σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτό το μέτρο, ιδίω στην Ελλάδα. Μετά από την έκκληση του Φεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα διατύπωσε μια πρόταση για έκτακτη βοήθεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί υποστηρίζουμε ιδιαίτερα αυτή την πρωτοβουλία. Το έργο εφαρμογή αυτή τη πρόταση έχει ξεκινήσει ήδη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα, θα εγκριθεί πριν από το Συμβούλιο τη 17η-18η Μαρτίου. Φυσικά αυτό περι... προϋποθέτει το Συμβούλιο θα εγκρίνει ένα διορθωτικό προπολογισμό για το 2016 για να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια και εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Πρέπει να δράσουμε επίση με συντονισμένο τρόπο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα επανέλθει η λογική, η φυσιολογική ε, λειτουργία του χώρου του Σέγγεν. Η συζήτησή μα χθε τόνισε ποια ήταν τα μέτρα τα οποία αναπαραίτητα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε στου επόμενου μήνε, κύριε Πρόεδρε. <clears throat> τα πράγματα προχωρούν γρήγορα. Νομίζω ότι είναι φανερό για όλου. ότι η κατάσταση ζητά από μας μια ταχεία δράση και μια κοινή δράση. Το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα πρέπει να καταλήξει σε πλήρη λύσει σε όλα αυτά τα θέματα για να καταλήξει και στι κατευθύνσει για του επερχόμενου μήνε. Όλε αυτέ λοιπόν οι εξέλιξει έχουν την πλήρη προσοχή μα. Συγχρόνω δεν πρέπει να ξεχάσουμε και άλλε προκλήσει που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο του Μαρτίου θα αντιμετωπίσει το θέμα τη απασχόληση, τη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα όπως γίνεται κάθε, σε κάθε αρινή σύνοδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν θετικά μηνύματα. Υπάρχει ανάκαμψη ε, στην Ευρώπη παρά το γεγονός ότι η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αλλά έχει μειωθεί η ανεργία σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση Τίποτα όμω δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο. Είναι εύθραυστη ακόμα η ανάκαμψη και θα πρέπει να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τι προσπαθίε μα. Η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη ξεκινά και το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο του 2016. Η αναχώραση τάσει βρισκόνται στην καρδιά αυτού του εξαμήνου. Γι' αυτό η Προεδρία έχει τονίσει ιδιαίτερα την εφαρμογή αυτών των συστάσεων στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η κοινή συζήτηση λοιπόν που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες στη μήνυ ολομέλεια του το Βρυξελών ήταν πάρα πολύ σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δώσει κατευθύνσεις για τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες που θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπαθίες μας εφέτος. Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις θέσεις απασχόλησης, η εσωτερική αγορά είναι το πιο σημαντικό μας ατού για να μπορέσουμε να έχουμε μόνιμα οικονομικά ωφέλη. Χαιρόμαστε που γίνονται πολλά προσπάθεια για την στρατηγική της εσωτερικής αγοράς και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την ψηφιακή ατζέντα μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα και η Προεδρία μας χαίρεται για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπογραμμίσει και πάλι τη σημασία της εσωτερικής αγοράς για να μπορέσει ακόμα περισσότερο να εφαρμοστεί το θεματολόγιο της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση του κεκτημένου. Ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο Κορυφής του Ιουνίου θα μπορέσει να δώσει συνέχεια σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έννης Πλάσα Λεοπρόδος. Δίνω το λόγο τώρα εξ ονόματο της Κομισιόν στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μιλώ εξ ονόματο του Πρόεδρου Γιούγκερ σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποια μηνύματα τα οποία έχει στείλει πάρα πολύ συχνά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπαθεί να δώσει πολιτικέ απαντήσει στι μεγάλε προκλήσει τη εποχή μα. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά το ζήτημα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Το ευρώ αποτελεί ένα πολιτικό εγχείρημα, άρα χρειάζεται πολιτική διακυβέρνηση και δημοκρατική λογοδοσία. Έτσι λοιπόν η οικονομική μα στρατηγική απαιτεί οικονομικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα, εθνικά και ευρωπαϊκό επίπεδο ουσιαστικά θα εξολογηθούμε βάσει τη ικανότητά μα να μπορούμε να αποκριθούμε στι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα και αύριο. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν είναι μια τεχνοκρατική άσκηση, ένα τεχνοκρατικό εγχείρημα, αλλά μια πολιτική διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια δραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο ζήτημα νομιμοποίηση, αλλά μπορείτε πραγματικά κι εσεί να λογοδοτείτε ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Έχουμε μια ήπια ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις. Έχουμε βασικά μια μείωση της οικονομικής ανάπτυξης σε χώρες όπως η Κίνα και μείωση θέσεων απασχόληση, καθώ επίση και μειωτικέ τάσει στι παγκόσμιε αγορέ. Το 2016 θα είναι ένα έτος οικονομικής ανάκαμψης για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε ανάπτυξη τη τάση του 0,9%. Επιστρέφει η εμπιστοσύνη και δεν μπορούμε να ανησυχούμε πλέον ιδιαίτερα για την ε, Ευρωζώνη. Ήδη από το 2008 και μετά έχουμε δει μια ανάκαμψη και στις θέσεις απασχόλησης. Αυτό όμως δεν αρκεί. 22 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν εργασία και το ίμιση αυτών βρίσκονται κάτω της ηλικίας των 25 ετών. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη θητεία της, θεσπίσαμε μια ξεκάθαρη στρατηγική για τις θέσεις απασχόλησης. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε επενδύσεις, διαφορετικέ αλλαγές, καθώς επίσης και υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές. Ακολουθούμε λοιπόν την στρατηγική αυτή και στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής έχουμε μια έντονη αιμονία, θέλετε, στο ζήτημα της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς έχουν τα πράγματα γενικότερα στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, από το 2,2% του ΑΕΠ θα περάσουμε στο 1,9% φέτος. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά μας, να μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στους εαυτούς μας, αλλά και στις επόμενες γενναίες. Για πρώτη φορά σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, τα επίπεδα του χρέους έχουν αρχίσει να μειώνονται. Ας συνεχίσουμε σε αυτό το θετικό δρόμο. Όσον αφορά τώρα τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, αυτέ εναπόκεινται από τη βούληση των κρατών μελών. Από τι εκθέσει που έχουμε από τα κράτη-μέλη όμω έχουμε και συγκεκριμένα πλέον μηνύματα. Υπάρχουν πολλέ χώρε που σημειώνουν πρόοδο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τι οικονομίε μα. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέλαβε την θητεία τη, η πρώτη βασική πρωτοβουλία μα ήταν να ανταποκριθούμε πάρα πολύ γρήγορα σε μία από τι μεγαλύτερε αδυναμίε τη ευρωπαϊκή οικονομία, όταν υπήρχαν αρκετέ επενδύσει. Με τη βοήθεια όμω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να τονώσουμε τι επενδύσει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα τη προσπάθεια αυτή. Κατά, κατά τους πρώτους έξι μήνες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων κινητοποίησε πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε 22 από τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 8% περίπου των νέων αυτών επενδύσεων παίρνουν τη μορφή νιωτικών κεφαλαίων. Ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Ουσιαστικά σημειώνουμε πρόοδο, αλλά ακριβώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας και να συνεχίσουμε την, τον αγώνα που ξεκινήσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουν δράση αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη. Έρχομαι κατά αυτόν τον τρόπο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, καθώ επίση και στον πολιτικό ρόλο που διδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το εξάμεινο μα βοηθά να καταφέρουμε να εντοπίσουμε νέου κινδύνου, νέε προκλήσει και να καταφέρουμε να πετύχουμε νέα αποτελέσματα. Επικεντρωνόμαστε στι πιο επίγουσε προτεραιότητε. Κάθε κράτο μέλο συμβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο στο σύνολο, στην ενδυνάμωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις ε, εκθέσεις ε, των κρατών μελών που μας βοηθούν πάρα πολύ να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές και πολιτικές ε, εξελίξεις στα κράτη-μέλη και να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά προγράμματα συζητώνται και εφαρμόζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τις δημοσιονομικές ανισορροπίες τους. Έχουμε πρόοδο σε σχέση με τις συστάσει που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι και υπάρχουν διαφορέ βέβαια από τη μία χώρα στην άλλη. Οι προσπάθειε αυτέ θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βοηθήσουν και στη σύγκληση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Χθε ε, αποφασίσαμε επίση τι πρέπει να κάνουμε και με το ζήτημα των ε, δημοσιονομικών ανισορροπιών. Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι είναι λιγότερα πλέον τα κράτη-μέλη τα οποία παρουσιάζονται δημοσιονομικέ ανισορροπίε σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι θερετικό γιατί σημαίνει ότι τελικά καταφέρνουμε να μεταρρυθμίσουμε τις οικονομίες μας και καταφέρνουμε να συγκλίνουμε περισσότερο τις οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις 18 χώρες που εξετάσαμε, οι 6 δεν έχουν καθόλου ανισορροπίες, οι 7 παρουσίασαν κάποιες ανισορροπίες και 5 αντιμετωπίζουν υπερβολικές δημοσιονομικές ανισορροπίες. Υπάρχουν διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η βασικότερη ανησυχία είναι ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα χρέους, ιδιωτικού εξωτερικού, ότι πολλές φορές μειώνεται η αγωνιστικότητα και σαφώς θα πρέπει να λάβουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Καταλαβαίνετε ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργία ουσιαστικά βάλουν κατά της ε, κατά των οικονομιών και θα πρέπει να μειωθούν. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και τι μακροπρόθεσμε αδυναμίε μα. Δεν είναι εύκολο αυτό βέβαια γιατί κάθε φορά υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό κόστο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο όμω μπορούμε πραγματικά να τονώσουμε τι οικονομίε μα, να τι κάνουμε πιο ανταγωνιστικέ και να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει απασχόληση και μια πιο έντονη κοινωνική πτυχή στι πολιτικέ αυτέ. Απαιτείται όμω ένα πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό συντονισμό και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο τις προσπάθειάς μας. Την αξιολόγηση αυτή θα τη συζητήσουμε αυτό το μήνα και τον επόμενο μήνα με τα κράτη-μέλη. Το εξάμεινο βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του χρόνια μπορούμε να πούμε, αλλά έχουμε ήδη επιφέρει κάποιες αλλαγές προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο υπεύθυνο και κάποιες μικρές ενδεχομένως αλλαγές θα επιφέρουν πολύ σημαντικές τροποποιήσεις. Μπορούμε να καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα και να συντονίσουμε καλύτερα την όλη αυτή διαδικασία και να προβλέψουμε περισσότερο διάλογο και να καταφέρουμε τελικά να προωθήσουμε τι προτεραιότητε εκείνε οι οποίε θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη. Δημοσιεύοντα τι αιτήσει εκθέσει νωρίτερα, μπορούμε να κάνουμε και καλύτερε συζητήσει. Οι συστάσει μα πλέον είναι καλύτερα στοχευμένε. Επικεντρωνόμαστε συγκεκριμένε προτεραιότητε που απαιτούν την προσοχή των κυβερνήσεων των κρατών μελών για του επόμενου μήνε. Και δημοσιεύουμε τι συστάσει για την Ευρωζώνη στην αρχή πλέον του εξαμήνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί καταφέρνουμε και έχουμε σφαιρική εικόνα της κατάστασης και μπορούμε να έχουμε όλοι μια κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και για τις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Η αξιοπιστία του όμω δεν έχει να κάνει μόνο με τι καλέ οικονομικέ αναλύσει, αλλά και με τη διαφάνειά του και με τη λογοδοσία τη όλη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο εμεί αναφερόμαστε με κάθε δυνατή ευκαιρία στο εξάμεινο αυτό και επιφέραμε τι απαραίτητε αλλαγέ προκειμένου να έχουμε πολιτικό διάλογο και πολιτική συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε διαφορέ που υπάρχουν και να φέρουμε στη συζήτηση όλου του σημαντικού εταίρου όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε τη λογοδοσία εξουσία τη οικονομική διακυβέρνηση και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική μα στρατηγική οδηγεί στι θέσει απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Όσον αφορά τώρα την συζήτηση που έλαβε χώρα στι 7 Μαρτίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Βλέπετε ότι και οι δύο πλευρέ αποφάσισαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα παράτυπη μετανάστευση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητώντας με τον κύριο Νταβούτογλου είπαμε ότι όλους τους παράτυπους μετανάστες θα πρέπει να δεχθεί πίσω η Τουρκία, όλους αυτούς που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αυτούς που φτάνουν δηλαδή στην Ελλάδα. Τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι θα αρχίσει να ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να καταφέρουμε να επιστρέψουμε πίσω στην Τουρκία σύρους μετανάστες οι οποίοι θα μπορούν πλέον από την Τουρκία να κάνουν αίτηση για χορήγηση ασύλου. Η συμφωνία δηλαδή που έγινε στην βάση ένας προς έναν. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη λοιπόν. Με το νέο αυτό σχέδιο θα καταφέρουμε να σταματήσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη απόγνωση. Δεν θα υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα κίνητρο προκειμένου να πληρώσει κανεί του διακινητέ αυτού για να περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γνωρίζουν πλέον οι μετανάστε ότι μόνο μέσω νομίμων διόδων μπορούν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, προκειμένου οι Σύριοι πρόσφυγοι να έχουν τι καλύτερε ε, συνθήκε στην Τουρκία, θα δημιουργηθούν κάποιε νέε δομέ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην Τουρκία. Τα αρχικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε προβλέψει και το αρχικό ταμείο θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά το 2018. Όσον αφορά την πρόταση απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες, να σας πω τι είπε ο Επίτροπος Γιούνκερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις της και η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει και όταν θα συζητάμε για το άνοιγμα των νέων ενταξιακών κεφαλαίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι το επόμενο Συμβούλιο να επεξεργαστούμε περισσότερο τις λεπτομέρειες συμφωνίας αυτής οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τάχθηκαν υπέρ του νέου οδικού χάρτη προκειμένου να λειτουργεί πλήρως το Σέγγεν μέχρι τα τέλη του έτους. Ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, να σταματήσει η διέλευση των συνόρων χωρίς να γίνονται καθόλου διατυπώσεις και καλύτερο έλεγχο των συνόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ο δικό λοιπόν χάρτη για την αποκατάσταση του Σέγγεν απαιτεί περισσότερε προσπάθειε στι χώρε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη κρίση, όπω η Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα με επίση ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα νέο μέσο έκτακτη ανάγκη. Η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Θα πρέπει πάλι από αυτού να ληφθούν συγκεκριμένε αποφάσει πριν το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίση να δραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να εγκριθεί η απόφαση αυτή, είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του προπολογισμού 2016 να προβλεφθούν τα νέα αυτά κονδύλια. Για το 2016 προβλέπονται 300 εκατομμύρια και ακόμα επίση 200 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το 2017 και το 2018. Η χρηματοδότηση αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί από τεφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστική συμβολή Ευρωπαϊκή Ένωση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προκειμένου να έχουμε μια συντονισμένη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτόν το λόγο περιμένουμε και τη βοήθεια και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ομάδας του ΕΛΚΟ, κύριος Βέμπερ. Κύριε πρόεδρε, κύριε αντιπρόεδρε. Είναι πολύ καλό να έχουμε μια πρώην συνάδελφο ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου εδώ. Ε, δεν ξέρω τώρα τι κάνετε με αυτό το ε, αναλόγιο. Εκεί μπροστά έχετε και χώρο για να σας σερβίρουν καφέ. <clears throat> Είσαστε σε πολύ πιο άνετη θέση από τους υπόλοιπους βουλευτές εδώ που βρισκόμαστε. Στη συνέχεια όμως θα ήθελα να εκφράσω τη θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι πολύ καλό που έγινε αυτή η διάσκεψη κορυφής τη Δευτέρα <clears throat> και για πρώτη φορά έχουμε το διάγραμμα μιας πλήρους και αποτελεσματικής λύσης η Ευρώπη μαζί με την Τουρκία μπορούν να βρουν μια κοινή λύση η οποία θα μπορεί να έχει μόνιμο και αηφόρο χαρακτήρα. Θα πρέπει να σταματήσουμε την ελεύθερη διέλευση από το δρόμο των Βαλκανίων, πρέπει να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Αυτές είναι σωστές απαντήσεις και θέλω να τονίσω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και να την υποστηρίξουμε γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών που έχει συγκεντρωθεί στην Ιδωμένη και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Είναι θετικό στοιχείο από τη διάσκεψη της Δευτέρας. Θα πρέπει να τονίσω ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε και μια θέση σεβασμού προς την Τουρκία. Η Τουρκία έχει υποδεχτεί 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και έχει δαπανίσει 9 δισεκατομμύρια ευρώ για να τους περιθάλψει. Και η Ευρώπη μέχρι τώρα δεν έχει δώσει αρκετή σημασία στην προσπάθεια αυτά που έχει γίνει. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο ενεργοί στο μέλλον. Και αυτά είναι τα δύο σημεία λοιπόν τα οποία είναι πολύ σημαντικά να τα εξετάσουμε διεξοδικά. Τώρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια εταιρική σχέση με την Τουρκία, όχι μια σχέση εξάρτησης δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι στο μέλλον θα αποφασίσει η Τουρκία πόσους πρόσφυγες θα φέρνει στην Ευρώπη ή δεν θα φέρνει στην Ευρώπη και έτσι να ασκεί πίεση. Μετά μπορεί το Μαρόκο να πει αν δεν μας δώσετε τις ίδιες συνθήκες τότε θα ανοίξουμε και εμείς τα σύνορα προς την Ισπανία. Όχι, πρέπει να έχουμε μια εταιρική σχέση με αμοιβέ υποχρεώσεις και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα εξωτερικά της σύνορα και αυτό σημαίνει και τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προάσπιση των σύνορων της. Ένα δεύτερο το οποίο πρέπει να γίνει σαφές σε όλους είναι ότι αν εμείς δούμε το θέμα της ε, απελευθέρωσης <clears throat> στις προξενικές θεωρήσεις θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το ΕΛΚ είναι θετικό στο να εξεταστούν τα θέματα αυτά, αλλά υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Η Τουρκία θα πρέπει να τηρήσει τα απαραίτητα πρότυπα. Και αν δω την ε, προστασία δεδομένων στην Τουρκία, ξέρουμε ότι στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη αρχή δεδομένων στην Τουρκία και η Τουρκία θα πρέπει να το εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατό, όπως προβλέπετε. Επομένως δεν πρέπει να δώσουμε καμία επιταγή εν λευκό προς την Τουρκία και το ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο θα πρέπει να είναι κάπως πιο προσεκτικό για τα θέματα αυτά. Το πώς θα γίνει η φιλελευθερωποίηση αυτή για τις ε, προξενικέ θεωρήσει δεν είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά των Υπουργών Εσωτερικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επίσης όταν μιλάμε για εταιρική σχέση και όχι για εξάρτηση, τα οικονομικά μέσα τα οποία θα δώσουμε στην Τουρκία θα πρέπει να καταλήξουν στους πραγματικού δικαιούχου και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα επενδυθούν πράγματι στους καταβλισμού των προσφύγων και θα δοθούν άμεσα στην τουρκική κυβέρνηση. Λοιπόν, εταιρική σχέση αλλά όχι εξάρτηση. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μια τελευταία σκέψη θέλω να σας αναφέρω. Θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια διάκριση. Θέλουμε όλοι να λύσουμε το θέμα της μετανάστευση αλλά το θέμα της διεύρυνσης και τη ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. <clears throat> Για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία, η ομάδα μου είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστική σε σχέση με τη δυνατότητα πλήρους ένταξη στην Τουρκία. Θεωρούμε ότι δεν έχει θετικό χαρακτήρα μια τέτοια προοπτική. Πρέπει να πούμε όμω στην Τουρκία με σαφή τρόπο ότι Εάν θέλετε να είσαστε εταίρος μας δεν πρέπει να απομακρυνθείτε περισσότερο από την Ευρώπη. Οι επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία είναι πραγματικά απαράδεκτες. Η θέση, η υποκειδαιμονία της Ζαμάν <clears throat> είναι και η ανάληψή της από το κράτος είναι κάτι το οποίο είναι ε, απαράδεκτο. Δεν μπορεί να βγαίνει <clears throat> την επόμενη μέρα η Ζαμάν με μια γιγαντιά φωτογραφία του Ερντογάν, γιατί αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά η εφημερίδα αυτή τίθεται στην υπηρεσία τη κυβέρνηση. Κάνουμε λοιπόν μια έκκληση προ όλου. Έχετε να κάνουμε έκκληση προς την Τουρκία. Έχετε την ευκαιρία να έχετε μια εταιρική σχέση με την Ευρώπη. Γι' αυτό σταματήστε να <clears throat> επιτίθεστε κατά των μέσων ενημέρωσης. Σταματήστε να δημιουργείτε ένα αυταρχικό κράτο Αλλιώς δεν θα μπορέσετε ποτέ να προσεγγίσετε περισσότερο την Ευρώπη. <coughs> Και τώρα το θέμα το οποίο θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, που είναι το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Ευρώ. Το ανέφερε ο κ. Ντομπρός και αυτό κανονικά θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού του Ετησιανής Συνόδου του Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις στις χώρες όπου κυβερνά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βλέπουμε ότι υπάρχει οικονομική αύξηση, αμεγέθυνση και μείωση της ανεργίας Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην αλλάξει αυτή την πορεία και οι υπόλοιπε χώρε θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι η δική μα είναι η σωστή οδό και να την ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Για την Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα, ο πρόεδρος Πιτέλα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Τζανίν. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην συμφωνία. Συμφωνία που ακόμα βέβαια δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια Ευρώπη κυβερνήσεων η οποία δεν μπορεί πλέον ούτε καν να αποφασίσει. Για να σώσουμε την Ευρώπη και κυρίως για να σώσουμε τους χιλιάδες Σύρους που φεύγουν από τον πόλεμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία, αρκεί να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφισημία σε αυτή τη συμφωνία. Τα άτομα αυτά, και σκέφτομαι κυρίως τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αλλά και τους άντρες και τις γυναίκες. Είναι άνθρωποι, είναι ανθρώπινα όντα, δεν είναι νούμερα, δεν είναι εμπορεύματα. Η συμφωνία λοιπόν αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει παζάρι, παζάρεμα εις βάρος των ίδιων των μεταναστών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παζαρέψουμε για ζητήματα όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα όσα συνέβησαν αυτή τη στιγμή με την εφημερίδα Τζαμάν στην Τουρκία πρέπει πραγματικά να μας απασχολήσουν και θα πρέπει να στιγματίσουμε σωστικά τη συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας. Επίσης ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει τον κορδικό πληθυσμό. Όλα αυτά βαρύνουν αυτή τη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μην μπερδεύουμε το προσφυγικό ζήτημα με το ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας ή το ζήτημα της απελευθέρωσης των προξενικών θεωρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε και εμείς να εξετάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτάσεις αυτές της Τουρκίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους Σύρους δίνοντας χρήματα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν δίνουμε λευκό επιταγή αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε μία διεθνή συνεργασία, η οποία όμω να σέβεται το διεθνέ δίκαιο, να σέβεται τη σύμβαση τη Γενέβη, να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουμε μία αξιοπρεπή λύση για όλους αυτούς τους ε, μετανάστες. Και ας μην ξεχνάμε και την περίπτωση της Ελλάδας, που αυτή τη στιγμή μοιάζει να γίνεται ένα κλουβί μπορούμε να πούμε για τους μετανάστες, οι οποίοι φτάνουν εκεί, συσσωρεύονται εκεί και δεν μπορούν να πάνε πουθενά άλλου. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε λοιπόν και τη χώρα αυτή μέσω μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες, μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως άλλωστε έχει αποφασιστεί. Όταν θα γίνει η πρώτη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν όλε αυτέ οι παράνομε διελεύσει προ την πρώην Κρουσταδική Δημοκρατία τη Μακεδονία και προ άλλε χώρε. Και μην ξεχνάμε και την περίπτωση τη Συρία. Η Συρία που βρίσκεται πραγματικά στη γειτονιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή πραγματικά επηρεάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν και για τη Συρία μια πολιτική συμφωνία, όπου ηγετική θέση μέσω τη κυρία Μογκερίνη θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε ειρήνευση στην περιοχή. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε επιτέλους πάλι μια ομαλότητα και μια σταθερότητα στη Βόρεια Αφρική και στη Μεσόγειο και δεν θα ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο σε κατάσταση συνεχή αναστάτωση. Είτε μιλάμε για την Τουρκία πάντω, είτε μιλάμε για τη Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εξωτερικεύουμε τα ευρωπαϊκά προβλήματα σε άλλε χώρε. Δεν θα λύσουν τα δικά μα τα προβλήματα άλλε χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη μέσω δεσμευτικών αποφάσεων. Α μην περιμένουν οι άλλοι να κάνουν για μα αυτό το οποίο πρέπει εμεί να κάνουμε η πτώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σταματήσει μόνο αν καταφέρουμε να κτίσουμε την ηθική μας δύναμη, αν καταφέρουμε να ανακτήσουμε πραγματικά την αξιοπιστία μας, αυτή πραγματικά μας προωθούσε και μας πρόβαλε περισσότερο σε όλο τον κόσμο. E Ο το λόγο από την του ECR. Την περασμένη εβδομάδα μας δόθηκε μια σαφή, ένα σαφής μήνυμα ε, για τους παράτυπους μετανάστες. Είπε να μην έρχεστε στην Ευρώπη, να μην πιστεύετε τους διακινητές. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να σπάσουν αυτήν την διέλευση με τις βάρκες. Για να αναχαιτήσει κανείς την ροή θα μπορούμε να εστιαστούμε στο να βοηθήσουμε τους μετανάστες, τους πρόσφυγες που χρειάζονται προστασία. Αλλά είμαστε σαφείς, οι εχθροί μας δεν είναι οι πρόσφυγες που φεύγουν από τις διώξεις και τον πόλεμο. Οι εχθροί μας δεν είναι οι παράτυποι που έρχονται από άλλες χώρες και που χρησιμοποιούν ε, την κατάσταση για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Οι εχθροί μας είναι οι διακίνητες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτούς ε, τους ε, που βρίσκονται σε απόγνωση την Δευτέρα οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν το πλαίσιο με την τουρκική κυβέρνηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία, αλλά πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω και επιφυλάξεις και ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα η διαδικασία. Βλέπουμε ένα ή δύο ηγότες, ηγέτες ε, που ε, συνεργάζονται με την Τουρκία χωρίς να έχουν συμβουλευτεί τις άλλες χώρες. Δεύτερον, δεν βλέπω πώς αυτό, όλα αυτά είναι νόμιμα ή πρακτικά πώς θα πρέπει ε, να παραβιάσουμε τις διεθνείς συμβάσεις και μετά ε, με ανησυχεί το γεγονός ότι ε, αντικαθιστούμε τους μετανάστες, ανταλλάσσουμε τους μετανάστες οικονομικούς με το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων χωρίς να βλέπουμε τις συνέπειες πώς τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν. Θα έχουμε σαφείς στόχους ή είδα δεν θα ήταν καλύτερα να ξοδέψουμε αυτό το μεγάλο ποσό εδώ με, ε, για τις επιστροφές. Και η Τουρκία η ίδια αυτοί που πιστεύουν στην ελευθερία του τύπου θα πρέπει να ανησυχούν για τη δράση κατά της, εταιρεία, της εφημερίδας Ζαμάν. Αλλά αν θέλουμε να εργαστούμε την Τουρκία για τη μετανάστευση ως φίλοι, ως φίλοι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί για το πώς είναι ρεαλιστικό να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν καταπατούνται οι ελευθερίες στη χώρα τους. Όποια και αν είναι η γνώμη μας θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι δεν θα αρχίσουμε να ελέγχουμε αυτή την κρίση αν δεν κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει ένας μόνος τρόπος για να επιληθεί αυτή η κρίση. Κάναμε με το πρόγραμμα με την κατάσταση σε αυτό το λάθος πέρσι, μην το επαναλάβουμε. Ενώ δεν μπορούμε να σταματήσουμε όλη τη ροή, μπορούμε να δείξουμε ότι ε, δεν είναι ανοιχτά όλα τα σύνορά μας και θα πρέπει να δούμε την συμφωνία των επανεισδοχών ε, και της επιστροφής και να βρούμε πόρους για να επιτυχύνουμε την ε, διαδικασία αυτή. Μπορούμε να βάλουμε πλοία ε, στο Αιγαίο για να καταπολεμήσουμε τους διακινητές. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Αλλά μήπως θα πρέπει να ξαναεπινοήσουμε το Δουβλίνο ή να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ένα, ένα σύστημα αποτελεσματικό για να βοηθήσουμε αυτούς που υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση ε, το Δουβλίνο ε, έχει, δεν έχει καμία αξία διότι δεν εφαρμόζεται. Μπορούμε να, να βοηθήσουμε στην ανθρωπιστική κρίση, αλλά μην κάνουμε το λάθος ε, να έχουμε μια κακή αντιμετώπιση της Ελλάδος, διότι αυτό που προτείνουν μερικοί πολιτικοί και σας βλέπω ότι με κοιτάτε. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές φορές που αναφέρετε τον κύριο Καμάλ στις παρεμβάσεις σας, αλλά Ελπίζω να μην αναφέρετε το όνομά μου στον ύπνο σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω εσάς και άλλους σήμερα να μην ε, με κατακρίνετε, αλλά να εργαστούμε όλοι μαζί για να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Όχι ορισμένες λύσεις που δεν είναι πρακτικές αλλά πρακτικές λύσεις ε, για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, διότι το οφείλουμε στους πολίτες μας και στους πρόσφυγες ε, να αναχαιτήσουμε την ροή αυτών που δεν είναι πρόσφυγες ε, και να αναλάβουν χώρες την ευθύνη τους και να δώσουν καταφύγιο σε αυτούς των οποίων η ζωή διακυβεύεται. Ευχαριστώ. Ο κύριο Έθριτς θέλει να σα θέσει ένα ερώτημα. Το δέχεστε? Äh, um ένα ερώτημα το οποίο ε, θα θέσει ο κύριος ε, Εθερίτς. Έχετε ζητήσει όλοι σχεδόν από το UKIP να λάβετε το λόγο, αλλά θα δώσω το λόγο στον Εθερίτς, κύριο Εθερίτς μονάχα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Καμάλ. Εγώ σας είχα θέσει την τελευταία φορά ένα ερώτημα προς, για την Τουρκία και έχετε ε, ακολουθήσει αντίθετη θέση από αυτή που είχε ακολουθήσει ο αρχηγός σας, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας σε σχέση με την ε, Τουρκία. Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα να καταδικάσετε αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει με την Τουρκία ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση οικέτευσε την Τουρκία να σώσει το πρόβλημά της και της έδωσε χρήματα προστασίας ουσιαστικά. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό. Κύριε Εύριτζ, δεν είστε ούτε αφελής, ούτε πραγματικός αισιόδοξο. Αν θέλετε εδώ να κατακρίνω τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό της χώρας μου, θα έλεγα ξυπνήστε πρωτού να έρχεστε εδώ. Αλλά αυτό το οποίο Αυτό που θα σας έλεγα είναι επίσης τον κατακρίνεται στις διαπραγματεύσεις και κανένας ο Πρωθυπουργό δεν έκανε περισσότερο για να διαπραγματευτεί μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτόν και γι' αυτό θα πρέπει να τον επενέσετε. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Δίνω τώρα το λόγο για την φιλελεύθερη ομάδα στον κύριο Φερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι ε, κατάλαβα δεν πρέπει κανείς ούτε να κοιτάζει τον κύριο Καμάλ ε, και πάντως δεν θα ε, εξεπλήξω τον κύριο Καμάλ διότι σύμφωνο μάλλον με τις κριτικές που εκφέρατε σχετικά με την πρόταση που είναι επιτάπητος. Χρειαζόμαστε πρακτικές και τεχνικές ρυθμίσεις ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης. Αλλά αυτή δεν είναι ρυθμισή πρακτική και τεχνική. Είναι μια συμφωνία με την Τουρκία όπου εμείς ε, θα εξάγουμε τα προβλήματά μας σε μια συμφωνία όπου θα δώσουμε το κλειδί εισόδου, τα κλειδιά για τις πύλες της Ευρώπης στην Τουρκία για την επιτυχία του Ερντοάν, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα αποφασίζουν για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι τι είναι η συμφωνία. Η συμφωνία είναι ότι εμείς θα μπλοκάρουμε συλλογικά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Σύρους και για άλλα άτομα και είναι η Τουρκία ατομικά που θα αποφασίσει ποιος είναι πρόσφυγας που θα μπορεί να μπει σε, μια, σε έναν διανταλλαγή, έναν προς έναν. Παραδείγματος χάρη οι, οι Αυγανοί οι οποίοι καταπολεμούν ε, το Ισλαμικό κράτος και οι Κούρδοι που θέλουν να φύγουν από το Ιράκ και από άλλη χώρα δεν θα γίνουν δεκτοί ίσως, μάλλον, να ε, περιληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καμάλ για μία φορά και βρίσκω ότι αυτή η συμφωνία είναι προβληματική. Προβληματική επειδή ένας ε, τύπος ε, ενός ροφουλμό συλλογικού και μια απόθεσης συλλογικής και αυτό απαγορεύεται από την Σύμβαση της Γενέβης. Επιπλέον πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να ξέρουμε ότι η ε, Τουρκία είναι πλήρες μέλος αλλά δεν έχει ε, επικυρώσει ορισμένα πρωτόκολλα. Ένα παράδειγμα, η Τουρκία δεν δίνει πολιτικό άσυλο στους Σύρους, μόνο πολιτικό άσυλο σε πρόσφυγες που έρχονται από χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και δεύτερον, δεν παρέχει άσυλο σε θύματα εσωτερικών σειράξεων, όπως την σύραξη που υπάρχει στην νοτιοανατολική Τουρκία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη διένεξη είναι λοιπόν προβληματικό να ζητούς, από μια χώρα η οποία δεν έχει πλήρως δεχθεί τα πρωτόκολλα της Σύμβασης της Γενέβης, να τους πούμε εσείς θα κάνετε τη δουλειά. Είναι σαν να λέγανε οι Αμερικανοί στους Μεξικανούς, εσείς θα ορίζετε τα σύνορα στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ προβληματική αυτή η συμφωνία. Και δεύτερον, όλα αυτά και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω αυτό το συλλογισμό του κυρίου Ντομπρόφσκι ε, που έχει επαναληφθεί σήμερα το πρωί. Ναι, είναι ένας τρόπος να σταματήσουμε τους διακινητές. Είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε την παράνομη διακίνηση. Εγώ δεν είμαι καθόλου αυτή τη γνώμη. Νομίζω ότι θα συμβεί το αντίθετο, μειώνοντα την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο ε, τρόπο όπως το κάνουμε τώρα, δίνοντας μόνο στην Τουρκία την δυνατότητα μόνη της ε, να παρέχει δικαίωμα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι αυτοί οι πεγνωσμένοι πρόσφυγες θα ψάξουν άλλες εναλλακτικές οδούς και πάλι σας λέω ότι είχαμε μια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο ε, για την, ανα, για την, ε, την οδό της Λαμπεντούζα, από τη Μάλτα, από την Αλβανία, από την Βουλγαρία και δεν θα επιλύσουμε το πρόβλημα, διότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί από άλλους, από τρίτες χώρες, θα πρέπει να λυθεί από μάσα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λείπει τώρα. Η έκκλησή μου σε εσά κύριε Ντομπρόφσκι και στην κυρία Πλασχάρτ είναι να κάνουμε αυτό το οποίο είναι αναγκαίο στο επόμενο Συμβούλιο να λάβουμε μια απόφαση για την στρατηγική για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μα μας λέτε ότι κάνουμε πρόοδο. Μα είναι μήνες που κάνουμε πρόοδο γιατί δεν χρησιμοποιούμε το άρθρο 78 παράγραφο 3 της συνθήκης το άρθρο 78 σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε έκτακτα μέτρα σε, περί... σε περίπτωση ε, εισρωής μεταναστών και προσφύγων. Δεν χρειάζεστε άλλη νομοθεσία. Μπορείτε βάσει ε, της συνθήκης να κάνετε κάτι, να αρχίσετε με αυτό, με τους φύλακες ε, στα σύνορα της Ελλάδας, με την Τουρκία. Και αυτά τα τρία δισεκατομμύρια. Γιατί να πληρώσουν τα κράτη-μέλη 3 δισεκατομμύρια να μην τα πληρώσουν στις, στις ε, τουρκικές αρχές και στις ΜΚΟ, αλλά απευθεία στα στρατόπεδα για να μην ζουν με 7 δολάρια το μήνα, διότι αυτός είναι ο λόγος που έρχονται σε εμά διότι πρέπει να επιβιώσουν με 7 δολάρια το μήνα και αυτά τα 3 δισεκατομμύρια πρέπει να είναι άμεση βοήθεια στους πρόσφυγες. Και πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο ε, για το σύστημα ασύλου. Να αλλάξουμε το Δουβλίνο. Τι κάνουμε στην πράξη. Δεν αλλάζουμε το Δουβλίνο. Βάλαμε και την Τουρκία μέσα στο σύστημα του Δουβλίνου. Αυτό αποφασίσαμε. Αντί να αλλάξουμε το σύστημα του Δουβλίνου και να έχουμε μια καλή ε, δίκαια κατανομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εγώ από την αρχή ήμουνα της γνώμης ότι ίσως αυτή η συμφωνία θα μπορούσε ε, να βοηθήσει. Αλλά όσο περισσότερο την εξετάζω, τόσο περισσότερο βρίσκω ότι είναι αρνητική ε, και θα ήθελα να ζητήσουμε από τον κύριο Τούσκ να, να, να, να φτιάξει μια πραγματική ευρωπαϊκή συμφωνία. Η κυρία Γκραπίνη θέλω να σας θέσει ένα ερώτημα κύριε αν συμφωνείτε. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σαφέ ότι είστε δυσαρεστημένο. Αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά από την παρέμβασή σα. Ωστόσο, να σα ρωτήσω το ακόλουθο. Μετά τον λόγο του κυρίου Αντιπροέδρου, θεωρείτε εδώ πέρα ότι έχουμε πραγματικά ένα σαφέ συνεπέ πρόγραμμα γιατί ε, ο Αντιπρόεδρος μας έλεγε ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε αποκατάσταση του Σέγγεν. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε μια συμφωνία πολύ γρήγορα για τους επόμενους τρει ή έξι μήνε ή μια ολοκληρωμένη συμφωνία μόνιμη την οποία θα μπορούσαμε πραγματικά να εξηγήσουμε στου Ευρωπαίου πολίτες Και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να έχουμε δύο κατηγορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες Σέγγεν και χώρες εκτός Σέγγεν. Πρωτού απαντήσετε κύριε Φερχόφστατ. Κύριε Γκραπίνη, αν μιλάτε πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να σας ακούσουν οι διερμηνείς, τότε αυτά που λέτε δεν πρόκειται να διερμηνευτούν. Παρακαλώ και εσάς και όλους τους συναδέλφους μιλάτε με ένα ρυθμό ο οποίος να μπορεί ανθρωπίνως να ερμηνευτεί. Ο κύριος Φερχόφστατ. Και εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω πολύ καλά το ερώτημα, λέει ο κύριος Φερχόφστατ. Κάτι ρωτήσατε για το Σέγγεν. Είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή λύση και δεν είναι μοναχά θέμα Σέγγεν αλλά είναι και το ίδιο θέμα με το ευρώ. Κάναμε τα ίδια ασφάλματα, ξεκινήσαμε και μετά είπαμε «Α, ξαφνικά δεν έχουμε τρόπο να προστατεύσουμε την, ε, τη, τα σύνορα του Σέγγεν, όπως δεν έχουμε ένα κοινό σύστημα για να προστατεύσουμε το ευρώ». Πρέπει να πάρουμε λοιπόν κάποια μαθήματα και όχι να λέμε «Οι Τούρκοι θα λύσουν το πρόβλημα». Όχι, εμείς πρέπει να επομιστούμε τις ευθύνες μας μέσα και έξω από το Σέγγεν. Πολύ καλή απάντηση κύριε Φερχόφστα, δεδομένου δεν καταλάβατε το ερώτημα, λέει ο πρόεδρος. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Τσίμερ για την Ενωτική Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια ικτρή εικόνα που δημιουργούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της κοινή γνώμης. Την Δευτέρα Έχουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτή το δηλητηριασμένο δώρο των τουρκικών αρχών, της τουρκικής πλευράς. Και κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν θέλανε να το λάβουν υπόψη. Έχουμε εδώ πέρα μία κατάσταση που είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να παζαρεύουμε για τις ανθρώπινες ζωές και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο προτείνεται τώρα θυμά, μας θυμίζει μια κατάσταση όπου θα κατηγοριοποιήσουμε τους ε, πρόσφυγες επί τη βάση της εθνικής ή ακόμα και τοπικής προέλευσής τους. Και αυτό είναι μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σκεφτείτε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Ιδωμένη και περιμένουν να τους επιτραπεί να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν το ταξί τους και τους οποίους έχει αρνηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το δικαίωμα. Και το λέω σαφώς σε όλους οι οποίοι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Αυτό το οποίο επετευχθεί δεν είναι ευρωπαϊκή λύση. Αυτό το οποίο είδατε τη Δευτέρα δεν ήταν καθόλου ευρωπαϊκό. Οι προσπάθειες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αφορούσαν μονάχα τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντά τους ως εκπροσώπο των χωρών τους. Δεν κάνανε κανένα βήμα παραπάνω για μια κοινή λύση. Η προηγούμενη διάσκεψη κορυφής είχε αποφασίσει ότι δεν θα κλείσουν τα σύνορα και τώρα έχουν κλείσει τα σύνορα. Και αυτή τη στιγμή τη Δευτέρα ή την Τρίτη το πρωί λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τι θα γίνει, ας κλείσουμε και τα υπόλοιπα σύνορα. Και βλέπω τώρα την Ελλάδα. Πολύ ωραίο ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια πρόταση να υπάρξει ένα νέο εργαλείο ανθρωπιστικής βοήθειας και να βοηθήσει τους φορείς οι οποίοι εργάζονται εκεί για τους πρόσφυγες. Αυτό δεν αλλάζει όμως τη φύση του προβλήματος. Τίποτα δεν αλλάζει ό,τι αφορά το βάρος που πρέπει να φέρει η Ελλάδα και την έλλειψη αλληλεγγύης μας με ένα κράτος μέλος. Εγώ ξέρω πολύ καλά από τη δική μου εμπειρία, το ξέρω από το πετσί μου τι σημαίνει να κτίζει κανείς τείχη και φράχτες. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να θεωρεί ότι μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα ένα ακυβέρνητο κράτος. Ο κ. Τεμεζιέρ είχε πει την ε, Δευτέρα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει απλώς ένας χώρος συσσόρευσης προσφύγων. Αυτά είναι απλώς κοιν, κοινικά όμως. Δεν υποστηρίζουν την κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα για την Τουρκία. Εμείς έχουμε παραδώσει τον εαυτό μας στην Τουρκία, στα χέρια της Τουρκίας. Μια Τουρκία που εμείς δεν θέλουμε να δεχτούμε με την αυταρχική αυτή κυβέρνηση της. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι όλα αυτά τα οποία είχαν συζητηθεί για την Τουρκία να τα στείλουμε στο περιθώριο. Είμαστε έτοιμοι να συνδιαλλαγούμε και να διαπραγματευτούμε με μια χώρα η οποία σκοτώνει τον ίδιο πληθυσμό της που βομβαρδίζει την Συρία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με τον Ερδογάν. Αυτό δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γι' αυτό ζητώ την δική σας, κάνω μια κλίση εσάς να μην, να πείτε όχι σε αυτό. Ευχαριστώ λέω ο, ο πρόεδρος για την ομάδα των Πρασίνων ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πτώχευση ηθική. Αυτές είναι λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό μετά τη Δευτέρα. ηθική αποτυχία, διότι αντί να τον τιμωρήσουμε, ανοίγουμε την αγκάλι μας σε ένα καθεστώς ενός ανθρώπου που ε, καταπνίγει κάθε δημοκρατική αντιπολίτευση και για να κερδίσει τις εκλογές βομβαρδίζει τον πληθυσμό και αναζωπυρώνει τον εμφύλιο πόλεμο. Οι Σύροι μόνο να βοηθηθούν, λένε, ε, ε, για αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν με παράτυπους τρόπους, μειώνοντας βεβαίως αυτούς που πεθαίνουν στον δρόμο. Ε, θεωρήσεις, ε, ενταξιακή ε, διαδικασία, όλα αυτά επειδή μια πλειοψηφία της Ένωσης και στην Γερμανία έχει υιοθετήσει αυτήν την γνώμη και ορισμένη υπέρ μιας λευκής και χριστιανής Ευρώπης δαπανώντα χρήματα για να μην μιλήσουμε για όσους κρύβονται δειλά πίσω από όλα αυτά. Είναι σημαντικό κυρίες και κύριοι, ε, οι αρχηγοί κρατών να υιοθετήσουν μέτρα που θα θέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ύψος των ηθικών και νομικών υποχρεώσεων της. Έχετε δίκιο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ασφαλή οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η οδός δεν μπορεί να προορίζεται μόνο για τους Σύρου. Υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν ε, που είναι θύματα πολέμου. Ε, δεν μπορεί ε, να ξανασταλούν στην ε, Τουρκία και ε, για την σύμβαση της Γενέβης κάθε ετών άσυλο δικαιούται εξέταση ατομική της αίτησή του και αν μπορείτε να βρείτε ξέρω πόσα δισεκατομμύρια για να βοηθήσετε στην υποδοχή εκεί νομίζω ότι εμείς η πλούσιοι Ευρώπη θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο για την υποδοχή εδώ αλλά υπενθυμίζω ότι πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε 0,25% του πληθύσματός μου. Είναι 100 φορές λιγότερο από μια χώρα όπως ο Λίβανος και η Ορδανία ε, που ε, δέχονται περισσότερους και χρειάζονται τη βοήθεια μας. Για αυτήν την πολιτική θα πρέπει να μιλήσουμε για την Τουρκία, αλλά όσο πιο ισχυρή θα είναι η αποφασιστικότητά μας τόσο θα μπορέσουμε να πιέσουμε τον Ερντογάν, διότι γεωπολιτικά είναι βάλωτη η Τουρκία, οικονομικά επίσης και χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ευρώπη την Τουρκία. Η πρώτος όρος επιτυχίας προϋποθέτει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα δράσουμε μαζί. Και θα ήθελα να απευθυνθώ σε δύο χώρες κυρίως. Ε, κύρια ε, ε, Χένις Πλεσάτ έρχεστε από τις κάτω χώρες και προεδρεύετε και η χώρα σας είναι χώρα του πολιτικού φιλελευθερισμού όταν η Ευρώπη είχε να κάνει με τους θρησκευτικού πολέμους και τα πολιτερχικά καθεστώτα η χώρα σας δεχόταν όλους τους πρόσφυγες του Ευρωπαίους ως προς την Γαλλία αντί να επιδείξει μια αλληλεγγύη επιφανειακή και αντί να κάνει ο πρόεδρος μάθημα στην καγκελάριο και δίνοντας παράσημο στον, στον ε, κληρονόμο, στον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας θα πρέπει η Γαλλία να αναλάβει τις ευθύνες της για να μπορεί να είναι πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κάνει μερισσότερη προσπάθεια και να ε, είναι περισσότερο ηγετική. Και απέναντι στον Κατσίνσκι, στον Ορμπάν, στον Πεγκιντά, στον Φίτσο, πρέπει να, για την Ευρώπη, την χριστιανή για να γίνει Ευρώπη φρούριο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εδώ και 18 ε, μήνες τι είπε ο Πάπας Φραγκίπτος. Είπε ότι θα πρέπει μαζί να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μεταναστών. Δεν πρέπει να γίνει ακροταφείο η Μεσόγειος. Μας έλεγε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα εάν με σαφήνεια μπορούσε ε, να επιδείξει την ταυτότητά της στην πολιτιστική και να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και να εγγυηθεί την υποδοχή, την υποδοχή ε, των μεταναστών, να έχει δίκες πολιτικές συγκεκριμένες που να βοηθούν τις χώρες προέλευσης να επιλύσουν τις εσωτερικές διενέξεις αντί για πολιτικές συμφερόντων που τροφοδοτούν αυτές τις διενέξεις. Θα πρέπει να δράσουμε στις αιτίε και στις συνέπειες. Ο Πάπας έλεγε ότι όσοι ορθώνουν ε, τύχη και όχι ε, γέφυρες δεν είναι χριστιανοί. Ε, πρόκειται γέφυρες και όχι τύχη αυτά που βάλαμε στα χαρτονομίσματά μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μία ακόμη φορά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες πλέον γίνονται μόνιμες και απασχολούν τις συζητήσεις μας. με την αστευτική κρίση και η οικονομική κρίση. Τα δύο αυτά ζητήματα διαφορετικά μεταξύ τους ως προς τη φύση τους. Παρόλα αυτά όμως καλούμεθα ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε με τρόπο ιδιαίτερα επίγοντα. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε αυτή τη στιγμή ότι χρειαζόμαστε λύσεις οι οποίες να είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές που υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα. Περισσότερες προσπάθειες για την οικονομική κρίση. Μόλον ότι κάναμε προσπάθειες δεν καταφέραμε τελικά να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, δεν καταφέραμε να τους καθησυχάσουμε, να τους προστατεύσουμε. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει απαραίτητη αλληλεγγύη, ούτε καν αλληλεγγύη στη μέθοδο που ακολουθούμε. Και αυτό το βλέπουμε στην αντιμετώπιση που διαφυλάξαμε για την Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτε μα βρίσκονται σε ιδιαίτερη αδύναμη θέση. Η μεταναστευτική κρίση στη συνέχεια μα βρίσκει για άλλη μια φορά έκθετου σε μηχανισμού οι οποίοι επηρεάζονται και αυτοί με τη σειρά του από την οικονομική κρίση. Είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ κυβερνήσει ε, οι οποίε προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την έλευση αυτή των μεταναστών θεωρώντας ότι θα πρέπει να καταργηθούν όλοι αυτοί οι κανόνες που θεωρούσαμε δεδομένους όλα αυτά τα χρόνια και ουσιαστικά στρέφονται κατά της ίδιας ενοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδεικνύουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια ουσιαστική παράλυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τι βασικέ αυτέ δηλώσει που γίνουν ότι δίθεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη ή πρόοδο, ουσιαστικά λέμε ότι θα τι συζητήσουμε όλα στην επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Εξακολουθούν λοιπόν και υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πώ θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε με μια χώρα όπω η Τουρκία, που πριν από λίγε μέρε έλαβε αποφάσει οι οποίε στρέφονται κατά τη ελευθερία του λόγου και τη ελευθερία τη έκφραση. Πώ ακριβώ θα πραγματευτούμε με αυτού του ανθρώπου. Είναι σαφέ ότι αν πραγματικά θέλουμε να δούμε τα πράγματα κατάματα, κατάματα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν αναλαμβάνουν την απαραίτητη δράση οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, πιο αποτελεσματική προσέγγιση που θα οδηγήσει σε λύση των κρίσεων αυτών. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Α μην ξεχνάμε τι βασικέ μα αξίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι θα έπρεπε να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ελευθερία λοιπόν, πολύ ωραία. Βλέπουμε, αυτή τη στιγμή ζητάμε από την Τουρκία να κάνει μια προσπάθεια για να δεχθεί περισσότερους πρόσφυγες και θα δώσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν μπορούμε όμω να ανταλλάξουμε την υποχρέωση αυτή υποδοχή που έχει η αλλω η Τουρκία με το ζήτημα τη καταστολή ελευθερία του λόγου. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στι δράσει και τι βασικέ τη αρχές ως προς τη δικαιοσύνη. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια κατοίκου. Το 2015 δεχθήκαμε χιλιάδες πρόσφυγες. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραλύει και γονατίζει εξαιτία των χιλιάδων αυτών προσφύγων σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση που έχουμε στα σύνορα μεταξύ Ελλάδο και Μακεδονία, λέει ο μιλητή. Ω προ τη δικαιοσύνη επίση, πρέπει πάλι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε δράσει προκειμένου να εξηγήσουμε στου συμπολίτε μα ποιο θα γίνει αποδεκτό, με ποιο τρόπο, πώ θα γίνει υποδεκτό και ποιο θα πρέπει να επαναπροωθηθεί. Χρειάζονται δηλαδή ουσιαστικέ αποτελεσματικές λύσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Άνεμανς θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Κύριε Μπορέλη, το δέχεστε? Άνεμανς. Έχω ένα ερώτημα για σας κύριε Μπορέλη για να διευκρινιστεί η συζήτηση που γίνεται ακούγοντάς σας ξέρω ποια είναι η άποψη του UKIP για την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση αυτά που λέτε εσείς τώρα σήμερα αλλά εκπροσωπείτε το σύνολο της ομάδος του EFTD ή μόναχα του δικού σας κόμματος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είχε επιληθεί και πριν από κάποιους μήνες στην Ολομέλεια όταν σας είχαμε πει ότι εμείς ως Ιταλική συνιστός είχαμε μια άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν το είχατε παρατηρήσει αυτό τότε. Για την ομάδα η κυρία Λεπέν έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι σκληρή η αλήθεια. Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντοχάν ε, μας επέβαλε κάτι σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ε, αδύνατη και είναι η μεγάλη ε, μαλακή μέδουσα, έτσι την είχα ονομάσει και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Αφού δώσαμε 3 δισεκατομμύρια για να μειωθεί η ροή των μεταναστών και δεν απέδωσε τίποτα, ζητάει σήμερα 6 δισεκατομμύρια. Ε, βεβαίως οι υποσχέσεις δεν τηρούνται τον ε, Ιανουάριο. Ε, περισσότεροι μετανάστες από την Τουρκία έφτασαν στην Ελλάδα σε σχέση με το 2015. Σας εξαπατά ο Ερντογάν, σας εκβιάζει ο Ερντογάν ακόμη και απαιτεί σήμερα την κατάργηση των θεωρήσεων για τους Τούρκους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας ως ανταμοιβή για τη μη συνεργασία του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθιστά κάποιον πιο δυνατόν, αλλά έχει μια αδυναμία, μια αδυναμία ε, σημαντική την οποία εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν. Μα σας δείχνει πώς τα ηθικά σας μαθήματα τα αγνοεί διότι με τις επιλογές σας τις ανεύθυνες τον κάνατε υπερισχυρό. Ένα, μια εφημερίδα τη αντιπολίτευση. Ε, έκλεισε από τους αστυνομικούς που με δακρυγόνα απεμάκρυναν τις πολίτες, βομβαρδίζονται οι Κούρδοι στη Συρία. Οι Κούρδοι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Νταέσ και της Αλκάιντα έχει ε, καταρρύψει ένα ρωσικό αεροπλάνο, η Τουρκία συμμετέχει στο λαθρεμπόριο πετρελαίου της ΑΕΣ και εσεί το αγνοείτε. Αποσταθεροποιείται από πάρα πολλά θέματα λόγω των μεγάλων λαθών εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του Ερογάν. Αυτή την χώρα θέλετε να εντάξετε στην Ευρώπη. Ας υπενθυμίσουμε ότι μια χώρα βρήκε αποτελεσματική λύση για την μετανάστευση είναι η Αυστραλία. Μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια καμπάνια έγινε σε όλες τις χώρες για να προειδοποιήσει ότι οι παράτυποι και τα πλοία θα επαναπατρίζονται στις χώρες προέλευσης και από την πολιτική ε, ε, απέφερε καρπούς. Ας είμαστε ρεαλιστικοί, ας υιοθετήσουμε την ίδια πολιτική. Ας έχουμε εθνικά σύνορα στερεά Ας έχουμε στρατόπεδα στη Συρία και στις γειτονικές χώρες για να εγκατασταθούν ευπρεπώς οι μετανάστες με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι θα κερδίσουν εμείς οι Ευρωπαίοι ε, όπου οι χώρες μας δεν θα κατακλειστούν από αυτούς τους μετανάστες διότι αυτοί δεν θα μπορούν πια ε, να έλκονται από υποσχέσεις απατηλές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη που δεν είναι εγγεγραμμένη έχει το λόγο. Κυρία Υπουργέ, εξ ονόματος ε, του Συμβουλίου και κύριε Επίτροπε ε, που εκπροσωπείτε τον κύριο Γιούγκερ, θα σας παρακαλούσα να διευκρινίσετε με τρόπο ευθύ για τους πολίτες της Ευρώπης τι ακριβώς είναι η μεγάλη αλλαγή για την οποία ε, κάνετε λόγο. Ίσως ε, εμείς δεν ξέρω αν καταλάβαμε καλά. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι εφ' εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει σε κανέναν από καμία δυστυχισμένη χώρα να έρθει και να εγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνον πρόσφυγες από εμπόλεμες χώρες. Μπορείτε να απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Πάρα πολύ σύντομα για το ποια είναι η κατάσταση. Η δεύτερη μου ερώτηση, οι Ευρωπαίοι οι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Μιλάτε καμιά φορά για την ε, μετανάστευση, την μεταναστευτική πολιτική. Έχω 1,5 λεπτό, Έχω 1,5 λεπτό κύριε Πρόεδρε. Ναι, μπορείτε να μου το δώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ. Το, η δεύτερη ερώτηση είναι καμιά φορά μιλάτε για μετανάστευση, για μεταναστευτική πολιτική εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το άσυλο ή ε, την πολιτική των προσφύγων. Δεν ε, είναι μια, ένα θέμα γνώμης, αλλά παρόλα αυτά για τους Ευρωπαίους πολίτες θα ήθελα να διευκρινίσετε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τίποτα να κάνει με την μεταναστευτική πολιτική των κρατών μελών. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι σαφές αυτό, είναι γεγονός. Συμφωνείτε ότι αυτό είναι γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μορβά. Για δύο λεπτά η κυρία Νίβλα. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Όλα εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες. Μετά από τη συμφωνία η οποία σε γενικές και αδρές γραμμές συμφωνήθηκε θα πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας κατά των διακινητών. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους μας ότι χθε την ημέρα των γυναικών μιλήσαμε για την κατάσταση των γυναικών που είναι μετανάστριες, που έχουν εκθέσει τον εαυτό τους και τα παιδιά τους σε μεγάλο κίνδυνο πολλές φορές στα χέρια των διακινητών. Τώρα έχουμε μια συμφωνία με την Τουρκία η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και εγώ θέλω να πω ότι Χαίρομαι και χαιρετίζω αυτήν την διαπραγμάτευση και την πρόοδο που επετεύχθη. Δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα ακόμα, δεν υπήρξε κάποια τομή όπως ελέγχθη, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο εάν συνεργαστούμε με την Τουρκία. Πρέπει να υποστηρίξουμε την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους διακινητές και γι' αυτό είναι απαραίτητη και απαραγράπτη μια συμφωνία με την Τουρκία. Θέλω να τονίσω ότι η σχέση μας με την Τουρκία δεν έχει να κάνει με την ένταξη. Είναι μια συμφωνία που θα πρέπει να υπόκειται σε σαφείς κανόνες, ιδίως σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των τριών δισεκατομμύριων. Για τα θέματα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να εμπλέξουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πιθανή ή ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας, στη, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τα θέματα της διευκόλυνσης της προξερικές θεωρήσεις και εγώ έχω μια πολύ κριτική στάση για το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο και στο παρελθόν και δεν καταλαβαίνω πώς το Συμβούλιο μπορεί να παίρνει θέση για τα θέματα αυτά χωρίς την άποψη του Κοινοβουλίου Επομένως, εγώ βλέπω με πολύ επικριτικό και σκεπτικιστικό τρόπο μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νίμπλερ. Για δύο λεπτά ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και δύο μήνες ο κύριος Ρούτε και ο κύριος Τούσκ είπαν ότι είχαμε δύο μήνες για να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Πέρασαν δύο μήνες. Μάλλον περνάνε, τελειώνουν την επόμενη εβδομάδα. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ε, επόμενης εβδομάδος θα πρέπει να κάνει κάτι και θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πούμε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τι περιμένουμε από αυτούς. Εμάς μας απασχολεί αυτό που συμφωνούν με άλλους, αλλά μας δημιουργεί και ντροπή αυτό το οποίο γίνεται εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνδρες, οι γυναίκες, τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι χαμένοι μέσα στον ευρωπαϊκό χειμώνα έχουν την ίδια αξιοπρέπεια με τους ε, πολίτες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον Ισπανικό εμφύλιο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τις φασιστικές και κομμουνιστικές δικτατορίες, από τους πολέμους των Βαλκανίων. Θα πρέπει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να μην υποκύψουν στον πειρασμό του λαϊκισμού, να μην παραδοθούν στο φόβο, να πούνε καθαρά στην κοινή γνώμη των χωρών τους ότι οι βασικές αξίες και αρχές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πριτανεύσουν και σε αυτή την κατάσταση. Και επίση θα πρέπει να τους ζητήσουμε όλα αυτά που συμφωνούν με τρίτε χώρε να σέβονται τις αξίες της ανθρωπιστικής δράσης και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Πάνω απ' όλα όμω, δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σιωπηλοί ενώπιον αυτής της επιδημίας απανθρωπιάς που βλέπουμε <clears throat> σε τόσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή της απανθρωπιάς που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρία πλειοψηφία την καταδικάζει. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό στο όνομα του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι στο όνομα του Κοινοβουλίου, όχι στο όνομα το δικό μας και φυσικά και εγώ ο ίδιος το απέφχομαι τελείως και δεν το αποδέχομαι. Ευχαριστώ κύριε Αγγερέο Σαλόμ. Ενάμιση λεπτό κύριε Φωτίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω μιλώντας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Συντοποιούμε όλοι ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, η υπό το φως του επερχόμενου δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο το ζήτημα αυτό της ανταγωνιστικότητας γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Και πραγματικά εκτιμώ όλα αυτά τα οποία κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Τώρα όσον αφορά την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι μετά από πάρα πολλούς μήνες, μην πω χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά συντοπεί ότι είναι πολύ σημαντικό στρατηγικό εταίρος η Τουρκία. Βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο μιας τεράστιας ε, μεταναστευτικής κρίσης. Και βέβαια αυτή ε, η ε, στάση παζαρέματος που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που θα είχε πριν από κάποια χρόνια. Είχε γίνει τότε η συζήτηση αυτή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να φοβόμαστε αυτό το οποίο ορισμένοι συνάδελφοι ονόμασαν εξωτερήκευση των προβλημάτων μας προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι να αποθέτουμε όλα μας τα προβλήματα ή την έβρεση όλων των λύσεων στην Τουρκία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια εταιρική σχέση με την Τουρκία και βάσει μια εταιρική σχέση θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Προφανώς ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ντιβέλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη χαρά είναι για μας να μπορέσουμε να σας έχουμε και πάλι μαζί μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια παράθεση στα αγγλικά. Χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση στα θέματα αυτά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάθε συμβούλιο που παίρνει μια απόφαση ξαφνικά ανάγει τον μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή σε μικρότερο κοινό παρονομαστή αυτά είναι αυτά που είπε η βουλευτής Χένις ε, Πλάσαρ το 2009 όταν ήταν η για την πολιτική ασύλου. Τότε εξετάζεται το θέμα ενός υποχρεωτικού μηχανισμού κατανομής των προσφύγων. Η συμφωνία αυτή με την Τουρκία καταδεικνύει και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή είναι αμφισβητήσιμη νομικά και ανάξια σε ηθικό επίπεδο. Και κοιτάξτε και τα θέματα της, ευρωπαϊκής, της οικονομικής ανάπτυξης. Κύριε Ντομπρόφσκης, ποιος θέλει να επενδύσει σε μια Ευρώπη η οποία πάει για διάλυση. Κάνω μια έκκληση σε εσά και στην Ολλανδική Προεδρία. Εργαστείτε για μια αξιοπρεπή και μόνιμη και βιώσιμη πολιτική μετανάστευση. Ευχαριστώ κύριε Ίνφελτ. Ακολουθεί κύριε Βερζιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι από την Τουρκία και ε, με καταπλήσουν αυτά περί συμφωνίες, αυτά τα οποία είδα οι δικαστές, οι πανεπιστημιακοί που κατηγορούνται για τρομοκρατική δραστηριότητα, παρετούνται πάνω από 760 άμαχοι δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 100 παιδιά. Και η Σύρσε ε, δείχνει εικόνες ε, της Συρίας, μάλλον παρά δημοκρατικής χώρας. Η πόλη έχει καταστραφεί. Ε, το δίκαιο του πολέμου δεν τηρείται και οι σωροί εξαφανίζονται σε αυτό το ΠΕΗ, σε αυτή τη χώρα θα αναθέσουμε τη μεταναστευτική πολιτική. Οι τουρκικές αρχές δημιούργησαν την κρίση των ε, προσφύγων στην Ευρώπη, εκβιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτυγχάνουν. Πρέπει να αποφύγουμε ένα νέο σύρσε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την ψυχή της. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και θα πρέπει μια επίσημη αποστολή της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάει επί τόπου. Πάρα πολλές ομάδες το ζητούν αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βερισιά. Ο κύριος ε, Τέρι Κάμπρας έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Έχουν αναφερθεί πολλά επιχειρήματα. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα μονάχα. Πρώτον, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υπόχρεη παροχής βοήθειας στους μετανάστες. Ακόμα και αν αναθέσουμε κάτι στην Τουρκία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε το τι κάνει η Τουρκία και να έχουμε πάντα εγγύησεις που θα δοθούν. Και επίσης θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για τις χιλιάδες Ιρακινών Αφγανών και τα λοιπά που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία που έχει γίνει με την Τουρκία. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα. Η βοήθεια που μπορεί να δοθεί από την Τουρκία είναι μια ανθρωπιστική βοήθεια, βοήθεια ευκαιρίας. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να την ξεπληρώσουμε με διευκολύνσεις για να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεχάσουμε τις ε, προδιαγραφές μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, θα πρέπει να επομιστούμε τις πολιτικές και ηθικέ υποχρεώσει μα. Το να βοηθήσουμε τους ε, πρόσφυγες δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γονατίσουμε μπροστά σε ένα αυταρχικό κράτο το οποίο δεν τηρεί τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τέρη Κάμπρα, Ακολουθεί για τρία λεπτά ο κύριο Φάρατσου. Αυτή τη στιγμή πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη ανοησία. Η κυρία Μέρκελ μα είχε πει πριν από μερικού μήνε: Ελάτε όλοι, ελάτε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίστε πού βρισκόμαστε τώρα. Και τώρα μα εκβιάζει και η Τουρκία. Ήρθαν στην αρχή και μα ζήτησαν 3 δισεκατομμύρια και μα υποσχέθηκαν τότε ότι θα μειώσουν τον αριθμό των προσφύγων προ την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμω αυξήθηκαν οι αριθμοί αυτοί, επέστρεψαν οι Τούρκοι και λένε άλλα 3 δισεκατομμύρια θέλουμε τώρα και θα συνεχίσουν να επιστρέφουν και να ζητούν περισσότερα χρήματα, σα το λέω. Όπω είπε ο Κίπλινγκ όσον αφορά την εισβολή των Δανών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό είναι το τίμημα το οποίο πρέπει να καταβάλει κανείς. Όταν όμως καταβάλει κανείς το τίμημα, ουσιαστικά ουδέποτε καταφέρνει να διώξει τον εκβιαστή του και αναγκάζεται να καταβάλει νέα αντιτήματα. Και τώρα μας λένε ότι ε, η αποδοχή ενός σύρου πρόσφυγα θα προσβλέπεται για κάθε σύρο που επαναπροωθείται. Τους έχουμε πληρώσει ουσιαστικά μια ολόκληρη περιουσία και παράλληλα λέμε ότι θα πρέπει ε, τα 75 εκατομμύρια Τούρκων από τον Ιούνιο του 2016 να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να μείνουν θεωρητικά 90 μέρε, στην πρακτική βέβαια μπορούν βέβαια να μείνουν πολύ περισσότερο και να ζητήσουν οικογενειακή επανένωση και να αυξηθεί ο ρυθμό του τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως αντάλλαγμα τι λαμβάνουμε εμείς, τι απόφαση να επιταχύνουμε την προοπτική, την ευρωπαϊκή της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι ο Ντέβιτ Κάμαρον να ήταν τόσο καλός και πραγματεύσω όσο είναι οι Τούρκοι. Αυτό θα ευχόμουν, ευχόμουν μόνο. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θα μπούμε σε πολιτική ένωση με μια χώρα που έχει σύνορα με το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία. Ουσιαστικά θα έχουμε πολιτική ένωση με μια χώρα η οποία είναι φτωχότερη από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσβλέψουμε ελεύθερη κυκλοφορία για 75 εκατομμύρια Τούρκους υπήκοους. Σε μια κυβέρνηση επίσης η οποία είναι όλο και περισσότερο Ισλαμιστική και νομίζω και αυτα, αυταρχική. Είπαν ότι πραγματικά η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει σημείο καμπής, μα έχουν απόλυτο δίκιο σε το λένε αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μολονότι πέρασαν δέκα χρόνια και δεν έχει ενταχθεί ακόμα η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταλήξουμε τελικά να δώσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Το δημοψήφισμα πάντω στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει να κάνει με την πιο ασφαλή λύση. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρομοκράτε Ισλαμιστέ που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντα του δρόμου τη προσφυγιά. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε την Τουρκία, αν πραγματικά θέλουμε να επιτρέψουμε την αύξηση των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουμε να καταστήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα πιο ευάλωτο στην τρομοκρατία. Νομίζω το καλύτερο είναι να βγούμε ω Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακτήσουμε την κυριαρχία και τον έλεγχο των συνόρων μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φάρατς. 1,5 λεπτά το, ο Δεν υπάρχει θάρρος στους Ευρωπαίους ε, ηγέτες. Ντροπή σα έχετε συνθηκολογήσει ενώπιον του δικτάτορα Ερντογάν. Έχετε θέσει τα συμφέροντα των κρατών πάνω από την Ευρωπαϊκή Ενότητα και έχετε υποθηκεύσει την ελευθερία μας. Με τη συμφωνία αυτή. Έχετε όλο και περισσότερο μια κατάσταση πανικού σε αυτήν την Ευρώπη που μοιάζει πια σαν Σοβιετική Ένωση. Αφήσατε τους Τούρκους να έλθουν στην Ευρώπη, να πάρει ο Σουλτάνος της Άγκυρας 6 δισεκατομμύρια ευρώ και να είναι ο επιδιαιτητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ε, θέτεται κάτω από το Ισλάμ και φαίνεται την μουσουλμανική Ευρώπη πια στο προσκήνιο. Αυτό το σχέδιο λοιπόν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Αμέσως θα πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε χρήματα στην Τουρκία, θα πρέπει να σταματήσουμε τη μετανάστευση, θα πρέπει να σταματήσουμε να υποβάλουμε τον ευρωπαϊκό πληθυσμό σε όλα αυτά. Μόναχα μια λύση υπάρχει, μόνο ένας τρόπος για να βγούμε από την κρίση, μόνο μια αποτελεσματική απάντηση υπάρχει στην ροή των μεταναστών που θέλουν μια καλύτερη λύση. Ας κλείσουμε και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά σύνορα και ας τα ελέγχουμε σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκράφ. Ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία Ντότς. Κύριε Πρόεδρε, σε μια εβδομάδα το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στα λεπτομεριακά θέματα που έχουν μείνει εκκρεμή με το σχέδιο συμφωνίας με την Τουρκία. Παρά τις θαραλές προσπάθειες του κυρίου Βέμπε να παρουσιάσει το θέμα αυτό ως μια εταιρική σχέση και όχι σχέση εξάρτησης με την Τουρκία. Η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτική μεταναστευσή μας είναι χαοτική, πολυδάπανη και ουσιαστικά ε, υποχωρεί ενώπιον της Τουρκίας για τα θέματα φιλελευθεροποίησης προξενικών θεωρήσεων και ένταξης. Και συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς θεωρούμε όμως ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από το να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο από μια κακή συμφωνία. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, όπως έλεγε ο πρόεδρος του Αγγλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερο δρόμο και ο δρόμος αυτός μας οδηγεί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Ντότς. Δύο λεπτά κύριε Γκζιμπ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή η συμφωνία με την Τουρκία κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, κάποιοι την κατακρίνουν λέγοντας ότι θα έχουμε εξάρτηση από την Τουρκία. Αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση χωρίς να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Το λέω εδώ και καιρό ότι η συνεργασία με εταίρους όπως η Τουρκία και η Βόρεια Αφρική είναι κάτι το απαραίτητο, είναι απαραίτητο η διαδικασία αυτή να γίνει πιο διεθνής, να περιλάβουμε τα Ηνωμένα Έθνη, διότι δεν πρόκειται για ένα περιφερειακό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο ε, πρόβλημα, διότι οι συνέπειες ε, είναι παγκόσμιες. και δεν μπορούμε να αποφύγουμε να εξετάσουμε τις ρίζες του προβλήματος. Αποφασίσαμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη ε, στις χώρες που υφίστανται πίεση μεταναστευτική. Συμφωνήσαμε να εφαρμόσουμε την κατάλληλη διαδικασία μεταναστευτική. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα που δεν λειτουργούν. Όλες οι χώρες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρόλο που η χώρα μου επιβεβαίωσε ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Η Τουρκία μπορεί να καταπολεμήσει τους διακινητές που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από τους μετανάστες που παράνομα μεταφέρονται στην Ευρώπη. Αλλά τους λένε ψέματα για τις δυνατότητες που θα έχουν στην Ευρώπη, προβάλλοντας ε, τα εξωτερικά σύνορα δεν θα βασιστούμε μόνο στις εξωτερικούς εταίρους. Πρέπει να τηρήσουμε τις δικές μας ε, ε, υποχρεώσεις, να γίνουν πιο ανθρώπινες οι ροές των μεταναστών, να δούμε ποιοι είναι οι πόλεμοι, τα εγκλήματα, οι γενοκτονίες, η Τουρκία είναι ένας μεγάλος γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ελευθερίας του τύπου. Ανεξάρτητα από τις λύσεις που θα υιοθετήσουμε πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Ένωση είναι μια αξία αυτή καθεαυτή που πρέπει να προστατευτεί όπως επίσης και το σύστημα Schengen. Ενάμιση λεπτό κυρία Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, τον προηγούμενο μήνα πήγα στην νότια Ανατολική Τουρκία και τα πράγματα εκεί πέρα είναι ξεκάθαρα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Τουρκία από μόνες τους δεν μπορούν να επιλύσουν την προσφυγική κρίση. Αυτό είναι σαφές για μένα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Το ότι η κατάσταση είναι εκτό ελέγχου. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ειλικρινή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία και η χρηματοδοτική βοήθεια προ την Τουρκία θα πρέπει να πάει σε αυτού που πραγματικά την έχουν ανάγκη για τρόφιμα, για προγράμματα εκπαίδευση, για κοινωνική ένταξη και ένταξη στην αγορά εργασία των προσφύγων. Η Τουρκία όμω από τη δική τη την πλευρά θα πρέπει να καταπολεμήσει τα δίκαια κινητών στο Αιγαίο Πέλαγο και θα πρέπει η ανταλλαγή προσφύγων να γίνει βάση του διεθνούς δικαίου. Είπατε κι εσείς αγαπητοί συνάδελφοι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, ή μάλλον ότι πρόκειται να σταματήσουν οι ροές μεταναστών στην Βαλκανική Οδό. Η Σλοβενία όμως από σήμερα επαναφέρει στα σύνορά της με την Κροατία το καθεστώς Σέγγεν. Πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιπε χώρες και οι χώρες του Βίσεγκρατ να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους προκειμένου να επιζήσει και να επιβιώσει ο χώρος Σέγγεν. Η Τουρκία σίγουρα είναι στρατηγικός μας εταίρος. Το μέλλον όμως τη σχέση αυτή θα έχει να κάνει με την ίδια την πρόοδο τη Τουρκία και είναι πραγματικά παράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα μέσα μαζική ενημέρωση καθώ επίση και με την αντιμετώπιση των Κούρδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Τουρκία από κοινού θα πρέπει να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά στα πλαίσια τη διεθνού κοινότητα. Κύριε Ντομπρόφσκη, η προχθεσινή Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό είναι μνημείο αποτυχίας και κινησμού. Η αναβολή λήψης μέτρων για το προσφυγικό και η παραπομπή του στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17 και 18 Μαρτίου σημαίνει ότι οι προσφυγικές ροές θα συνεχίσουν αμύωτες στην Ελλάδα με αποτέλεσμα στα τέλη Μαρτίου να φτάσουν τους 150.000 οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να χορηγήσει στην ελλάδα εδώ και τώρα κονδύλια για τους πρόσφυγες. κύριε ντομπrovskis η ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί να μετατραπεί σε ένα απέραντο προσφυγικό νταχάου. δεν πρόκειται να ανεχθεί τα ανατολίτικα παζάρια της τουρκίας που στοχεύουν στην αύξηση της πρίκας που ζητάει προκειμένου να σταματήσει τα δουλεμπορικά κυκλώματα που γεμίζουν τα νησιά του αιγαίου με πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες η ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί τι παρανομίε των σκοπιανών και των αλβανών που έχουν κλείσει τα σύνορα. ήρθε η στιγμή η ελλάδα να αποχωρήσει από τη σέγγεν να αναστείλει το δουβλίνο 3 και να επιβάλει οικονομικό εμπάργκο σε σκόπια και αλβανία ως αντίπεινα για τα κλειστά σύνορα. ευχαριστώ. Υπάρχει ένα ερώτημα για σας από τον ε, κύριο Φάνη. Κύριε Φάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να θέσω αυτό το ερώτημα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, έχω ένα ερώτημα για σας και στέκομαι στα σχόλια που κάνατε τώρα. Μιλήσατε για κινησμό και μιλήσατε και για το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες προσπάθειες εκβιασμού της Ευρώπης. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο η Τουρκία το κάνει αυτό, κάνει εκβιασμού, αλλά υπάρχει και εκβιασμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Κάμερον θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κουλτούρα αυτού του είδου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριε Μαρία, έχετε το λόγο. Κύριο Κάμερον, τοποθετήθηκα χθε αναλυτικά και εξήγησα ότι η απόφαση για τη Βρετανία που ψήφισαν όλοι οι ηγέτε στην ουσία δημιουργεί μια κατάσταση όπου επιβάλλονται πλέον αποφάσεις εις βάρος όλων των εργαζομένων με βάση την ηθαγένειά τους. έτσι ευρωπαίοι που θα δουλεύουν στη βρετανία δεν θα έχουν δικαιώματα αλλά και βρετανοί που θα δουλεύουν στη γερμανία θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα. ευχαριστώ. Ο μην με παρεξηγήσετε. Εγώ είδα να υπάρχει μια πρόοδο στην διάσκεψη κορυφής με την Τουρκία και ξέρω ότι έχουμε μια εταιρική σχέση με την Τουρκία. Μερικές φορές δεν μπορούμε να διαλέξουμε τους ε, εταίρους μας που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και κατάσχουν μέσα ενημέρωση. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να επηρεάσουμε το περιεχόμενο αυτή τη συμφωνία. Και εγώ δεν είμαι σίγουρο <clears throat> ότι η συμφωνία που έχει γίνει με την Τουρκία μα οδηγεί προ τη σωστή κατεύθυνση. ένα για ένα Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια δυνατότητα νόμιμης μετανάστευσης, αλλά δεν συνάδει με τις αρχές μας. Φιλελευθερωποίηση για τις βίζες. Μα τι σχέση έχει αυτό με τη μεταρρύθμιση. Και γιατί ανοίγουμε κεφάλαια στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όταν κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει στην Τουρκία. Για μένα το θέμα είναι πρέπει να έχουμε μια συνολική συμφωνία και πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ληφθούν και για την εσωτερική αγορά. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Υπουργέ, θέλω να υπάρξει και στην πράξη πρόοδος για το πακέτο σιδηροδρόμων στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τέλσκα. Για ένα λεπτό ο κύριος Χατζηγεωργίου. Κύριοι συνάδελφοι, εγώ σε τη συμφωνία αν αναφερόταν σε εμπορεύματα, αν αναφερόταν σε κυβότια ή φέρετρα, ειλικρινά ντρέπομαι γιατί ανθρώπινα πλάσματα αποφάσισαν για ανθρώπινα πλάσματα με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη έβγαλαν ανακοίνωση λέγοντας ότι καταστρατηγεί ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν δίνουμε αυτά τα τρία, έξι, εννιά δις και δεν ξέρω πόσα θα γίνουν να ανακηρυχθούν δύο πόλεις μέσα στη Συρία ως ασφαλείς πόλεις υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών της Αμερικής και της Ρωσίας και να ξαναχτίσουμε δύο πόλεις για αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Είναι μια συμφωνία Ρουσφέτη υπέρ της Τουρκίας. Επέστρεψα προχτές από τον Διάρμπακυρ. Είδαμε το κλείσιμο της εφημερίδας Ζαμάν. Δίωξη χιλίων ακαδημαϊκών και 200 άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στη Σουρ και απαιτούμε να υπάρξει ασφαλής τρόπος και δίωδος εξόδου αυτών των ανθρώπων. Και μέσα σε όλα αυτά η εξής χτεσινή εικόνα. Ο κύριο Νταβούτογλου να δίδει τριαντάφυλλα για την ημέρα της γυναίκας σε δημοσιογράφους γυναίκες την ώρα που στη χώρα του κλείνει και καταπατεί. Για ένα λεπτό κυρία Κέλλερ. Γιατί... Το Συμβούλιο της Δευτέρας ήταν ένα Συμβούλιο ντροπή και όνειδου. Όλα αυτά τα οποία αποφασίζουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι να παραδιάσουν το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και τις, αρχικές αρχές, τι βασικές αρχές του ανθρωπισμού. Θέλετε να κάνετε αποθήσεις, να στείλετε πίσω τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Μα η Τουρκία μπορεί να του καταστήσει στη Συρία ή το Ιράκ. Κλείνετε τα σύνορα, ώστε άνθρωποι που χρειάζονται διεθνή προστασία δεν μπορούν να την έχουν. Ακυρώνεται το δικαίωμα να ζητήσει κανείς και να έχει άσυλο. Και όλα αυτά τα κάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Και πώς μπορείτε να κοιμάστε το βράδυ με όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλερ. Για ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό, ο κύριος δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς αντιτιθέμεθα στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς λόγους. Και ο πρώτος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι η χώρα αυτή δεν ανήκει στην Ευρώπη, δεν τοποθετείται γεωγραφικά στην Ευρώπη. Μόνο το 3% της επικράτειας της Τουρκίας βρίσκεται στην Ευρώπη. Και επίσης θα έχουμε σύνορα έτσι με τη Συρία, το Ιράκ, με το Ιράν μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πραγματικά για εκβιασμό. Εκβιασμό κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία, προκειμένου να έχει περισσότερα χρήματα, προκειμένου να έχει απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων και προκειμένου να ενταχθεί τελικά κάποια μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πραγματικό εκβιασμό προκειμένου να μα βοηθήσει η Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή καταστήλει τα δικαιώματα μειονοτήτων, όπω οι Κούρδοι. Επίσης καταστήλει την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της δημοσιογραφίας και της έκφρασης και είμαι ιδιαίτερη επίκη σε αυτά τα οποία λέω και πραγματικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν Ισλαμιστικέ τάσει στη χώρα αυτή, οι οποίε συναντιούνται όλο και περισσότερο εξαιτία επίση και του κυβερνώντο AKP. Όσον αφορά το τουρκικό ΑΕΠ, αποτελεί μικρό ποσοστό το ΑΕΠ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα εγώ αυτή τη στιγμή να επιδεινώ τα, να κάνω τα πράγματα πιο δύσκολα για τους Σουηδούς, για παράδειγμα, φορολογούμενους από μια ενδεχόμενη προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, περισσότερο εκβιασμό θα δούμε από την περαιτέρω συμμετοχή της Τουρκίας στον διάλογο που έχουμε για το προσφυγικό. Ανταυτού πιστεύω ότι χρειαζόμαστε διάλογο με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση εκεί, στον διάλογο και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε 1,5 λεπτό κύριος Βιλίνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την οργή μου για την στάση των βουλευτών του, των μεγάλων κομμάτων με την συμμετοχή και των βουλευτών της αριστεράς για μια συμφωνία η οποία ζητά να παραμείνουν ανοιχτά τα τα σύνορα, τα σύνορα στην Ευρώπη και συγχρόνως να δοθούν δισεκατομμύρια στην Τουρκία και να δοθούν περισσότερες διευκολύνσεις στην Τουρκία ώστε να μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η στάση του, των αυστριακών κομμάτων της δεξιάς και των σοσιαλιστών έχει δημιουργήσει το πρόβλημα αυτό. Ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με συνισταμένες εσωτερικής πολιτικής. Το ίδιο πράγμα κάνει και η κυρία Μέρκελ, η οποία έχει θέσει όλη την Ήπειρο σε αυτή την κατάσταση. Και νοιάζεται περισσότερο για τους ανθρώπους στην Αραβία και στη Μέση Ανατολή από ότι για τους πολίτες στην ίδια της τη χώρα ως, ε, ως ε, καγκελάριος της ε, Γερμανίας δεν μπορεί με την απόφασή της να δεσμεύσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αυτή λοιπόν η συμφωνία είναι απαράδεκτη. Η Αυστρία θέλει να έχει την απόλυτη κυριαρχικότητά της για τον έλεγχο των συνόρων της και θέλει να απορρίψει οποιαδήποτε δυνατότητα να υπάρξει μέρος της Ευρώπης η Τουρκία χωρίς δημοψήφισμα. Ευχαριστώ κύριε Βιλίνσκι. Για ένα λεπτό ο κύριος Συναρινός προχθές πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη κορυφής μεταξύ ευρωπαϊκής ένωσης και τουρκίας. τα αποτελέσματα αυτής ήταν όχι απλά απογοητευτικά αλλά ένα διπλωματικό βατερλό για τους ηγέτες της ένωσης. 28 τουρκολάγνοι ηγέτες με ανάστημα νάνου κάθονταν και άκουγαν ένα στιγνό εκβιαστή ένα κοινό απατεώνα τον Ταβούντογλου, να θέτει όρους παράδοσης και υποταγής. θα αναφέρω τέσσερις από τους απαράδεκτους όρους που μεταξύ άλλων έθεσε επιπλέον χρηματοδότηση τρία δισεκατομμύρια ευρώ ευνοϊκότερο καθεστώς χορήγησης βίζας πρώτα η κένωση των ελληνικών νησιών από πρόσφυγες και μετά να ξεκινήσει η επαναπροώθηση λαθρομεταναστών άμεση επανακίνηση πέντε κεφαλαίων της ενταξιακής πορείας. κύριοι όπως έχουν γράψει οι οθωμανοί λόγοι ο τούρκος είναι πνευματικά βάρβαρος θεομπαίχτης αγύρτης και βρωμιάρης. ο τούρκος είναι σαν του σκυλί κάνει τον άγριο αλλά όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο το βάζει στα πόδια. ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να αντιμετωπίσει τον τούρκο είναι με πυγμή και αποφασιστικότητα τέτοια χαρίσματα όμως λείπουν από τους εκλεγμένου και μη πολιτικούς αφεντάδες της ευρώπης. έχετε ξεπουληθεί στον οθωμανό ερντογάν. ευχαριστώ. Κύριε Συναδρινά, δέχεστε ένα ερώτημα από τον κύριο Τσαμπάσκη. Παρακαλώ κύριε Τσαμπάσκη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν έχετε μετάφραση. Δεν μπορείτε να ονομάσετε μια χώρα η οποία να, λέτε ότι μια χώρα είναι βάρβαρη. Αυτό είναι ντροπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λέει ένας βουλευτής. Κύριε Τσαμπάσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, μήπως θεωρείτε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Ερντογάν είναι ντροπή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο και χοντρό πολιτικό σφάλμα των γραφειοκρατών στην Ευρώπη. Έχουμε προσκαλέσει εκατομμύρια μεταναστών να έρθουν στην Ευρώπη και τώρα υποτάσσονται στη δικτατορία του Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά τους θέλει να ανοίξει κεφάλαια διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι ουσιαστικά πολιτική αυτοκτονία. Είπατε κύριε συνάδελφε και νομίζω ότι η Ευρώπη κάλλιστα μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της ενάντια της Τουρκίας. Απλά αυτά είναι παιχνίδια και παζάρια τα οποία παίζονται μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Πιτικόφερ, είχατε θέσει ένα διαδικαστικό ερώτημα. Χωρίς μικρόφωνο, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο συνάδελφος που έλαβε το λόγο ονόμασε σκύλους τους Τούρκους. Αυτό είναι μια ρατσιστική διατύπωση που δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Παρακαλώ να το καταγράψετε αυτό στα πρακτικά και να αντλήσετε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Είπα ότι θα το ελέγξουμε κύριε Βιτικοφέρ Αυτή τη στιγμή είχα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσαμπάσκι και δεν παρακολούθησα τη διερμηνία. Η κυρία Γκροστέ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την Δευτέρα στις Βρυξέλλες ήταν βεβαίως η τελευταία ευκαιρία. Ακόμα μια άλλη σύνοδος, τα αποτελέσματα όπως και τα προηγούμενα είναι απογοητευτικά και ανησυχητικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Μαρτίου θα είναι κρίσιμο. Θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε μια Ευρώπη της Ένωσης, έτσι όπως επινοήθηκε πριν από 60 χρόνια και μια Ευρώπη όπου καθένας είναι για τον εαυτό του. Ο εγωισμός δεν είναι η απάντηση στην μεταναστευτική κρίση. Όπως πάντα η θέση μας απέναντι στην Τουρκία είναι τελείως αμφίσιμη. Αυτό ε, που άρχισε με την Τουρκία τη Δευτέρα είναι η χειρότερη διαπραγμάτευση που γνωρίσαμε εδώ και καιρό. Η Ευρώπη διαπραγματεύεται με την Τουρκία διρεμένη περισσότερα από ποτέ και χωρίς στρατηγική, χωρίς συνεννόηση μεταξύ όλων. Η Ευρώπη παραδίδεται στους ε, Τούρκους ε, στο λύκο. Αυτό που προτείνεται κυρία Υπουργέ είναι κάτι το απαράδεκτο. Κάθε εβδομάδα η Τουρκία έχει νέες ε, διεκδικήσεις, 12 κριτήρια, θεωρήσεις, είναι ένα μια κλιμάκωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύθηκε πριν από την 1η Ιουνίου να απαλλάξει από την υποχρέωση θεώρησης. Είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να ασκήσει την συναπόφαση στον τομέα. Το Συμβούλιο θα δώσει δώσει επιπλέον 3 δισεκατομμύρια. Δεν ήσασταν ικανοί ούτε καν να δώσετε τα 3 δισεκατομμύρια που υποσχεθήκατε τον Οκτώβριο. Και πώς θα ελέγξετε ε, την χρήση αυτών των χρημάτων. Η υποκρισία είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό και δεν θα πραγματοποιηθεί. Αυτό που θέλουμε είναι πράξεις, διότι η Ευρώπη δεν πρέπει να ρίχνει τις ευθύνες της στους άλλους. Ας σταματήσουμε αυτό το ατιμωτικό παζάρεμα και εκβιασμό για την Ευρώπη. Δέχεστε ένα από τον κυρία Γκροστέτ. Παρακαλώ, κύριε Λεμπρετόν. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτησή μου. Κυρία Γκροστέτ, συμφωνώ με τα όσα είπατε, καταγγέλλετε αυτή την συμφωνία με την Τουρκία που χαρακτηρίσατε ως ε, υποκριτικό. Θα απελευθερεθούν οι θεωρήσεις πολύ εύκολα και χωρίς να τηρούνται οι κανόνες. Υπενθυμίσατε ότι θα δοθούν 6 δισεκατομμύρια. Με τι αντάλλαγμα, με αντάλλαγμα υποσχέσεων από μια κυβέρνηση που δεν τήρει καμιά από τις ελευθερίες ε, στην χώρα της. Πώς μπορείτε να συνεχίσετε να υποστηρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιες σύνθηκες. 30 δευτερόλεπτα είναι η ερώτηση και 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Κύριε Αγκροστέτ, έχετε το λόγο και πάλι. Απλώ λέει η κυρία Αγκροστέτ, πιστεύω ότι η Ευρώπη δημιουργείται με τι διαδοχικέ κρίσει. αλλά σήμερα έχουμε μια κρίση χωρί προηγούμενο. Πιστεύω ακόμα στην ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει σε αυτή την κρίση, αλλά θα πρέπει να υπομειστεί πλήρω τι ευθύνε τη. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Μπουστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει λύση στη μεσταυτική κρίση αν δεν έχουμε συνεργασία με την Τουρκία. Πάντως, οι όροι της συζήτησης τη Δευτέρα δεν ξέρω ήταν οι σωστοί. Το να, το να καταφέρουμε να μειώσουμε τους πρόσφυγες προς την Ευρώπη ουσιαστικά μας έκανε να παραβλέψουμε πράγματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία αυτή με την Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει επιτυχία αλλά και αποτυχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης προκειμένου να λάβουν από κοινού τι ευθύνε του απέναντι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση. Βέβαια, παρόλα αυτά, θα πρέπει να επενέσουμε την Τουρκία για το ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει πάρα πολλού πρόσφυγε από τη Συρία και το Ιράκ και αυτή τη στιγμή δέχεται να υποδεχθεί ακόμα περισσότερου πρόσφυγε. Θα πρέπει να αναλυφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σταματήσουν οι παράνομοι δρόμοι μετανάστευση και να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών. Υποψήφια χώρα λοιπόν η Τουρκία αλλά η προσφυγική κρίση και οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει θα πρέπει να αποτελέσουν διαφορετικέ παράλληλε διαδικασίε. Και από αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά δείχνει μια στάση η οποία είναι πάρα πολύ δειλή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ καταδικάζω την καταστολή της εφημερίδας Ζαμάν από τις τουρκικές αρχές. Επίσης, η Τουρκία δεν θα πρέπει να λάβει καμία δράση η οποία θα θέσει εν κινδύνο την εκεχηρία στην Συρία και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στην περιοχή και επίση σε καμία περίπτωση θα πρέπει να προχωρά σε απειλέ προ κάποιου Τούρκου υπήκου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν ειρηνευτικέ συνομιλίε με τον κουρδικό πληθυσμό. Δέχεστε από τον κύριο Τόμπερ ένα ερώτημα. Κύριε Κόμπερν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μήπως θα μπορούσατε να συμφωνήσετε μαζί μου ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τελείως διαπερατά η καγκελάριος Μέρκελ ζήτησε από, σε πολλούς να έρθουν στην Ευρώπη ότι ήταν ανοιχτές στήρες της Ευρώπης και η συμφωνία με την Τουρκία για τη μετανάστευση είναι ανέκδοτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευρωπαϊκά κόσκινα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόμπον, λέει ο πρόεδρος. Άρου αγαπητέ συνάδελφε, πέρα από τις λαϊκίστικες αυτές δηλώσεις που τόσο συχνά ακούμε από αυτή την πλευρά του Κοινοβουλίου, πρέπει να σας πω ότι στην πράξη χρειαζόμαστε απεγνωσμένα ένα σύστημα το οποίο θα προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο τα σύνορα του Σέγγεν, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι υπέρ όλων μας και θα πρέπει με τους γείτονές μας να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το προσφυγικό ζήτημα. Λαϊκίστικες δηλώσεις ουδέποτε ουσιαστικά θα ευοδοθούν και δεν προσφέρουν καθόλου στη λύση. Ένα λεπτό για τον κύριο Κέρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Είναι μια κρίση αυτή. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ακόμα μια αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι ήταν το θέμα τη επανεγκατάσταση και τώρα είναι η λαθασμένη αυτή συμφωνία με την Τουρκία. Όπως είπε ο κ. Καμάλη, οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινεί μεταξύ τους. Δεν πρέπει να λέει ο ένας τον άλλο αυτό το οποίο πιστεύει. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια θαυματουργή λύση. Αν υπάρξει αποτυχία, αυτό θα επισκιάσει όλες τις άλλες λογικές λύσεις που μπορούν να γίνουν. 6 δισεκατομμύρια είναι πολλά για μια αποτυχημένη λύση. Σταματήστε να περιμένετε μια πανάκια. Στο τέλο θα καταλήξουμε με χρήση ατομική βόμβα. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε του κανόνε, να διατηρήσουμε ταχύ... τους κανόνες στα σύνορα, να έχουμε ταχύτερη επεξεργασία των προσφύγων. Όχι υπηχαίους τίτλου, αλλά είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτά που πρέπει για να λύσουμε την τωρινή κρίση. Ευχαριστώ κύριε Κύρκοφ. Δέχεστε μια ερώτηση από την κυρία Γιάκονσάρη. Ναι, κυρία Γιάκονσάρη. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστό είναι αυτό που λέτε κύριε Κύρκοφ, ότι δεν υπάρχουν απλές λύσεις και ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Μα αυτό ακριβώς δεν είναι το δια κυβευόμενος στη συμφωνία με την Τουρκία. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε το χειρότερο, να γίνεται αυτή η διακίνηση προσφύγων για να μπορέσουμε έτσι να επιτύχουμε και κάποια ενότητα δράση στα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό, περί αυτού δεν πρόκειται. Κύριε Κύρκοφ, και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το διακυβευόμενο. Όλο αυτό το σχέδιο συμφωνίας είναι κάτι που γίνεται βεβιασμένο και χωρίς τον σωστό προβληματισμό. Νομίζω πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας παρά την κρίση και να εστιάσουμε στις προτάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν όπως και ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Κίρκοπ. Ένα λεπτό κυρία Ντεσαρνές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι φυσικό να συνομιλούμε με την Τουρκία αλλά δεν είναι, είναι απρεπές να τις αναθέτουμε την φύλαξη των σύνορων, την διαχείριση του δικαιώματος ασύλου που είναι κατά της ολοκληρωμένης Ευρώπης που επιθυμούμε. Αν η Ευρώπη θέλει να υπάρξει θα πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Ε, να βεβαίως να αφήσει, να μην αφήσει την Ελλάδα μόνη της στην πρώτη γραμμή, να δεχθεί άλλους ε, και να ασχοληθεί με τα δικαιώματα ασύλου αυτών που βρίσκονται στην επικράτειά της, να θεσπίσει μηχανισμούς επανεισδοχής, να θεσπίσει γραφεία που θα τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες υποδοχής για την καταγραφή των αιτήσεων ασύλου, να τις δεχτεί, να τις αρνηθεί, να συνδέσει την οικονομική βοήθεια στην Τουρκία με το σταμάτημα των δικτύων των κυκλωμάτων διακινητών και να διαχειριστεί τις, ε, τα δικά της σύνορα με σύνοριοφύλακες και κατάλληλη ακτοφυλακή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δεσσαρνές, δέχεστε ένα ερώτημα από τον κύριο Φουντούλη. Ε, αγαπητοί, η Ελλάδα δεν έχει χερσαία σύνορα με χώρες της σέγγεν. συμφωνείτε με την ιδέα ότι η ελλάδα θα έπρεπε να βγει από τη σέγγεν ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν κίνητρα να έρχονται στην ελλάδα για να πάρουν χαρτιά και να ταξιδέψουν στην ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια τελείως αντίθετη θεώρηση με τη δική σας. Η Ελλάδα είναι μέρος του Σέγγεν. Οφείλουμε αλληλεγγύη σε κάθε στιγμή, πράγμα που δεν επιδείξαμε αρκετά τον τελευταίο χρόνο. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι η Ελλάδα, αλλά είναι και τα εξωτερικά σύνορα της δικής μας Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Ελλάδας περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριο Σουρμπάν Κρέχπο. Κυρίες και κύριοι, η πρόταση συμφωνίας με την ε, Τουρκία έχει σαν στόχο να, επιτρέ... να επανέρχονται άτομα τα οποία έχουν ζητήσει άσυλο χωρίς όμως να το έχουν καν ζητήσει. Έχουμε κάτι που είναι άδικο και ανήθικο και παραβιάζει το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο όπως είπε και ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών σε αυτό το ίδιο το ημικύκλιο. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη αρνείται τον εαυτό της. Εξωτερικεύει τον έλεγχο των συνόρων τους και κάνει υπεργολαβία στους Τούρκους το καθήκον μας για να παρέχουμε άσυλο. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει σε μια χώρα όπου μπορούν να παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα τους. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Με τη συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση νομιμοποιεί και γίνεται συνένοχος των επιθέσεων της Τουρκίας κατά του δικαιώματος ε, διαδήλωσης, κατά του τύπου, κατά των ε, μειονοτήτων και γίνεται συνένοχος και στους βομβαρδισμούς που γίνονται στο Κουρδιστάν. Με όλα αυτά γίνεστε συνένοχοι. Αν θέλετε να σταματήσετε τις μασφίες των διακινητών, ανοίξτε ασφαλείς διάβλους για να φτάσουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη. Αλλιώς τα χέρια σας θα είναι βαμμένα με αίμα. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη κορυφής κατέδειξε ότι υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύη, Υπάρχει έλλειψη κοινή ευθύνη για του ανθρώπου, του άνδρες, τι γυναίκε και τα παιδιά που φεύγουν από τον πόλεμο και του βομβαρδισμού και ζητούν καταφύγιο. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει να του δώσει στο όλο και πιο αυταρχικό καθεστώ τη Τουρκία όλο και περισσότερο εμείς απομακρυνόμαστε από τις ευρωπαϊκές αρχές και τις αρχές της, ε, ε, του ανθρωπισμού. Δυστυχώς, όλο και περισσότερο η κυβέρνηση της χώρας μου, της Αυστρίας, είναι έτοιμη να ακολουθήσει αυτόν τον επονίδιστο δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν οι εκπρόσωποι των αυστριακών κομμάτων να παραμείνουν πιστοί στην ε, θέση τους που είπαν ότι αυτή η στάση της Αυστρίας δεν είναι σωστή και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπε χθε ο ε, Επίτροπο των, Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να έχουμε <clears throat> με τύχη και με φράχτε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δείτε τι εικόνε στην ειδωμένη, δεν είναι αυτό το οποίο ε, θα πρέπει να μας ενοχλεί, θα πρέπει να μας ενοχλεί η καταστροφή της ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Ο κύριος Πάξας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί που επενούν αυτή τη στιγμή τη συμφωνία με την Τουρκία. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την ομάδα. Προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά τι έχει συμβεί, να καταλάβω τι συμβαίνει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εξαγοράσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια απελευθέρωση των θεωρήσεων Προσπαθεί να μας εξαγοράσει εν γέννη για 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει εγγενώσει η χώρα αυτή. Τι θα γίνει επίσης με τα 75 εκατομμύρια Τούρκων. Ενδεχομένως να έρθουν και να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά ενδίδουμε στον εκβιασμό της Τουρκίας. Περιμένουμε ότι η Τουρκία θα επιλύσει τα δικά μας τα προβλήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοκρατία δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά καθόλου με την υποχώρηση τη δηλή αυτή. Προφανώ πρέπει να τηρήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύσουμε κατά προτεραιότητα τα δικαιώματα των δικών μα πολιτών. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε διάφορες απαγορεύσεις που ενδεχομένω να έχουμε απαγόρευση του μπέικον, απαγόρευση των χριστιανιάτικων δέντρων, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία που επιθυμούμε για το μέλλον. Ή μήπω τελικά η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία γίνεται όλο και περισσότερο κάτι το οποίο δεν υφίσταται στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Παρόλα αυτά έχουμε ακόμα 50 ομιλητές για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να δώσουμε και μπλε κάρτε στη στιγμή που πρέπει να έχουμε και τη δικασία catch the eye και στη μία ακριβώ πρέπει να ξεκινήσουμε με τι πληροφορίε. Α περιορίσουμε λοιπόν τα αιτήματα μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε πάντω στο ερώτημα που έχετε από τον κύριο Φεράντ. Μπορείτε, αλλά σας παρακαλώ πολύ, ας μην υπερβείτε το χρόνο αγόρευσης και σας αποφύγουμε εν γέννη τη διαδικασία μπλε κάρτα. Λεκάρτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώ θέλει περισσότερα ανταλλάγματα η Τουρκία. Θέλει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, θέλει θεωρήσει. Δεν πιστεύετε αγαπητέ συνάδελφε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι πάρα πολύ αδύναμη στην συζήτηση αυτή, διαπραγμάτευση αυτή που γίνεται με την Τουρκία. Αγαπητέ συνάδελφε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει να μιλά απλώ γενικό λόγο για τα προβλήματα και να αναλάβει δράση. Έχουμε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων καταρχά και στη συνέχεια την πρόληψη των διενέξεων γύρω από την Ευρώπη. Έχουμε κάποια θετικά παραδείγματα σήμερα στον κόσμο. Το παράδειγμα τη Αυστραλία, για παράδειγμα. Δείτε πώ η Αυστραλία κατάφερε να, να λύσει το προσφυγικό πρόβλημα. Α ακολουθήσουμε τα θετικά αυτά παραδείγματα και ας μην προσπαθούμε εκ νέου να εφεύρουμε τον τροχό. Ο κύριος Υπουργέζο έχει το λόγο. Αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Επίτροπε, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το προσφυγικό, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η λύση η οποία προτείνεται είναι αναξιοπρεπής. Να ανοίγουμε τις πόρτες κατά αυτόν τον τρόπο στα αιτήματα του Ερντογάν. Ένας αναξιόπιστος ηγέτης ο οποίος τελικά έχει μετατραπεί σε πραγματικό εκβιαστή. Βλέπετε αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τι είπαν ορισμένοι Έλληνες συνάδελφοι οι οποίοι προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν όχι τον τουρκικό λαό πιστεύω αλλά την υπεροπτική και επιθετική αυτή πολιτική και στάση που ακολουθεί η τουρκική ηγεσία. Ορισμένοι όροι δεν λέω ότι θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί αλλά μπορούν να γίνουν κατανοητοί. Πραγματικό εκβιασμό έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας 20 δισεκατομμύρια ενδεχομένω να ζητηθούν. Και βλέπετε αυτό το αρχικό αίτημα πώς μειώθηκε στα επιπλέον τρία. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι θα ζητούσαν και 12 δισεκατομμύρια. Στην πράξη όμως δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζουν και έρχονται οι πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καθεστώς αυτός πώς άραγε χρησιμοποιεί τα χρήματα που του χαρίζει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά για να κρατήσει σε υπάνθρωπες συνθήκες τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην τουρκική επικράτεια. Η Amnesty International το είπε αυτό. Πραγματικό όνειδος αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω εγώ που συνήθως μιλάω κατά της μετανάστευσης. Αντί όμως να ακολουθούμε μία λογική τελικά λύση, Ουσιαστικά το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ακολουθούμε μια στάση επονίδιστη και νομίζω ότι οι ίδιοι οι ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα ντρέπονται αυτή τη στιγμή για τη στάση την οποία κρατούμε. Πραγματικά είναι όνειδο, πραγματική ντροπή αυτό το σχέδιο συμφωνία. Ο κ. Παπαδάκη έχει το λόγο τα συμπεράσματα συνολικά της συνόδου συνιστούν πρόκληση για τους λαούς επικροτώντας τη βαρβαρότητα που ζουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην ελλάδα επιβραβεύοντας το σφράγισμα συνόρων και τις απελάσεις. το άσπρο το κάνετε μαύρο τους κυνηγημένους πρόσφυγες από τη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου που εσείς η ευρωπαϊκή ένωση το νατο και οι ανταγωνιστές σας ανάψατε τους θεωρείτε παράτυπους μετανάστες. το ποιος είναι πρόσφυγας κρίνεται αυθαίρετα στο κοινικό αλυσβερίσι ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας με την ένθερμη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. το νατο που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο αιγαίο μετατρέπεται σε χωροφύλακά του η αστική τάξη της τουρκίας που συστηματικά αμφισβητεί σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα που οξύνει την επιθετικότητά της στη συρία απολαμβάνει τις ευρωνατοικές πλάτες ανταλλάγματα επιδοτήσεις και εμπορικές συμφωνίες. το συμπέρασμα αβίαστο σέγγεν δουβλίνο και όλοι οι μηχανισμοί καταστολής ενισχύονται και η ευρωπαϊκή ένωση και το νατο αποκαλύπτονται πλήρως ως αντίπαλοι των λαών και ενώσεις συμφερόντων των μονοπωλίων. γι' αυτό και η λαϊκή πάλι πρέπει να βάλει αυτούς και το εκμεταλλευτικό του σύστημα στο στόχαστρο. Κύριε ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για μένα υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία για το θέμα αυτό, πέραν όλων αυτών που έχουν αναφερθεί. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια αρχή που δεν μπορούμε να λησμονήσουμε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση μόνο με κοινό τρόπο. Και αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί στο προσκήνιο. Συγγνώμη. Δεύτερον, σε καταστάσεις όπως αυτή είναι απαραίτητο να υπάρξουν περιφερειακές συμμαχίες, όπως γίνεται σε αυτήν την περίπτωση με την Τουρκία ή με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας, πρέπει να κάνουμε κάποιες συμφωνίες, αλλά η αρχή είναι ότι αυτές οι περιφερειακές συμφωνίες είναι απαραίτητες για να λυθεί το πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή με την Τουρκία. Τρίτο, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να διατηρήσουμε τους μηχανισμούς ώστε οι βοήθειες αυτές που πηγαίνουν προς τους πρόσφυγες να φτάσουν πραγματικά στους δικαιούχους και όχι να υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει ένα τμήμα από αυτή τη βοήθεια στη μέση του δρόμου. Τέταρτον, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που συνδέεται με όλα αυτά, περισσότερο από πάντα είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία γιατί είναι και ένας παράγον ενίσχυσης της κατάστασης ασάφειας και αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε. Και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά και επίσης να ενισχύσουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων γιατί δεν είναι μονάχα το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών. Χωρίς την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων θα μείνει κουτσί η ευρωπαϊκή ενία αγορά. Γι' αυτό υποστηριζώ τον τον οδικό χάρτη της Κομισιόν ώστε η λειτουργία του Σέγγεν να αποκατασταθεί πλήρως πριν από το τέλος του 2016. Κυρία Ροντρίγκης. Πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα αυτή τη φορά να, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο μιας στρατηγικής, πολιτικής και ηθικής αστοχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς πρέπει να δημιουργήσουμε διάβλους από τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης για τους μετανάστες. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε τρόπους για να επανακτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης μέσα στα δικά μας κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την δυνατότητα προστασίας του Σέγγεν και των ευρωπαϊκών συνόρων. Δεν μιλώ για ένα. Για φράκτες και τείχους μιλούμε για πραγματικό έλεγχο των συνόρων από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για να εξασφαλίσουμε ότι οι πρόσφυγες γίνονται αντικείμενα αξιοπρεπούς υποδοχής και να οργανωθεί η εγκατάστασή τους στην Ευρώπη. Μόνο έτσι μπορούμε να επανακτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης και αυτό πρέπει να οργανωθεί ως μια μεγάλη στρατηγική επένδυση για το καλό της Ευρώπης. Μιλάμε για ένα ζωτικό συμφέρον της Ευρώπης και πιστεύω ότι αυτή η επένδυση μπορεί να δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπω σύνδεση μεταξύ των δύο θεμάτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και επίσης αντιμετώπιση των λύσεων που χρειάζονται για πιο έντονη ανάκαμψη στην Ευρώπη. Βασίζομαι λοιπόν στην Ολλανδική Προεδρία και την Κομισιόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια πιο φιλόδοξη λύση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Βαντάνελ το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο Δ. Φάρ, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πουλούμε ουσιαστικά ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στην Τουρκία. Βλέπετε την βία, τη βία καταστολή που χρησιμοποιήσει η τουρκική κυβέρνηση κατά της εφημερίδας Ζαμάν. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό. Είναι μια χώρα η οποία θέτει στη φυλακή πάρα πολλού ε, ανθρώπου αυτό που θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο παραδεινόμαστε στον εκβιασμό της Τουρκίας. Το 1632 η Βιέννη δέχθηκε επίθεση, αυτή τη στιγμή όμως δίνουμε στην Τουρκία που είχε επιτεθεί τότε πάρα πολλά ανταλλάγματα απελευθέρωση θεωρήσεων, ταξιακή πορεία, ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι η Τουρκία καταπατά την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της έκφρασης. Σταματήστε λοιπόν αυτή τη διαπραγμάτευση με τους σουλτάνους της Τουρκίας. Κύριε Βαντάλεν, μία μπλε κάρτα έχουμε για σας, θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Μπονάνο, σας παρακαλώ πολύ να είναι πραγματική ερώτηση και όχι μια παρέμβαση. Αν δεν είναι σύντομη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Αν είχατε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εσείς, αγαπητέ συνάδελφοι, στην επόμενη σύνοδο, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι θα κάνατε, τι βασική δράση θα επιλέγατε προκειμένου να αντιταχθείτε στα φαινόμενα αυτά τα οποία περιγράψετε πριν από λίγο. Αγαπητέ συνάδελφε, πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει το προσφυγικό να συνδεθεί με την ταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δύο διαφορετικά ζητήματα είναι για μένα αυτά. Δεύτερον, πάρα πολλά χρήματα προτιθέμενα να δώσουμε στην Τουρκία. Πού θα πάνε τα χρήματα αυτά, ποιο θα ελέγχει τη χρησιμοποίηση αυτών των χρημάτων, πώ θα ξέρουμε ότι τα πανώνται σωστά. Εγώ θα προτιμούσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση να πάμε εμεί στην Τουρκία, να χτίσουμε εμεί τα κέντρα υποδοχή και να μην αφήσουμε όλα αυτά τα χρήματα να πάνε στι τσέπε των Τούρκων ηγετών. Περισσότερη λιγή επίση πρέπει να δείξουμε με την Ελλάδα προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν πλήρω τα hot spots στη χώρα αυτή και θα πρέπει επίση η καταγραφή εκεί πέρα να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριε Παγκατσορταντού Ερούιθ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία βουλευτής είπε πριν από λίγο ότι η Ευρώπη πέρασε από τη μία κρίση στην άλλη. Και έχει εμπιστοσύνη, θα ξεπεράσει και αυτή την κρίση. Εγώ δεν νιώθω αυτή τη στιγμή τέτοια εμπιστοσύνη. Αν θέλουμε να υπάρξει αυτή η μασική απόθυση των προσφύγων από τη Σουρία, Συρία στην Τουρκία. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι κυβερνήσεις μας έχουν παραβιάσει την αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να προστατεύσουν τα κράτη αλλά όχι την Ευρώπη. Ο πανικός τους δείχνει ότι θα έχουμε ένα πιο αβέβαιο μέλλον όλοι μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραμένουμε αδρανείς μπροστά στα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη μας. Λένε ότι με αυτή τη συμφωνία θα λείψουν τα κίνητρα για να περάσει κανείς στο Αιγαίο. Αλλά μιλάμε για άτομα που έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν μια αίτηση ασύλου. Μετά από μήνες ψευδών υποσχέσεων, αυτή τη στιγμή του αποστερούμε και από αυτό το δικαίωμα. Σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές οι χώρες μας δεν έχουν τηρήσει τις προηγούμενες ε, συμφωνίες για επαναγκατάσταση των προσφύγων, για χρηματοδότηση, για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Και αντί να γίνει αυτή η απρεπή συμφωνία με την Τουρκία, που ούτε και αυτή θα τη τηρήσουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε εσά και στο Συμβούλιο και ακόμα περισσότερο δυστυχώς και στην Κομισιόν. Αντιδράστε λοιπόν επιτέλους. Ο κύριος Παπαδημούλης. Κύριοι του Συμβουλίου, έχετε υπερβολικές προσδοκίες στο ανατολίτικο παζάρι με το αντιδημοκρατικό καθεστώς Ερντογάν επειδή εσείς οι 28 κυβερνήσεις αποδεικνύεστε ανίκανες να εφαρμόσετε τις δικές σας αποφάσεις. Τις αποφάσεις που πήρατε το Σεπτέμβριο για μια ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό σύμφωνα με όσα πρότεινε η Κομισιόν και συμφώνησε και πίεσε να εφαρμοστούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι η χώρα μου η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν τεράστιο καταβλισμό προσφύγων με κλειστά τα βόρεια σύνορά της και με το δράμα της ιδωμένης που αποτελεί ντροπή για την ευρώπη. οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό χωρίς την ελλάδα και πολύ περισσότερο εναντίον της ελλάδας. ο ευρωπαϊκός βαλκανικός διάδρομος πρέπει να ανοίξει τώρα αμέσως για τους πρόσφυγες και όχι εν καιρό όπως μας είπατε. οι χώρες του Βίζεγκρατ που παραβιάζουν τις κοινέ ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να υποστούν κυρώσεις σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέλος της συνθήκης Σέγγεν και φυλάσσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι τιμωρία. Κουραστήκαμε εμείς οι Έλληνες να ακούμε λόγια και φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Θέλουμε επιτέλους έμπρακτη αλληλεγγύη και πράξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Βαλέρο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα περισσότερα πράγματα υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Καταγράφω αυτή τη στιγμή ότι ακούμε πάρα πολλές επικρίσεις από τους συναδέλφους. Οι πράσινοι και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι αποδοκίμασαν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Ελπίζω οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου να ακούσουν πραγματικά αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή. Ξεπουλάτε, όπω είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά στρέφεστε κατά τη ίδια τη Σύμβαση τη Γενέβη μόνο και μόνο για να προχωρήσετε σε ένα μέτρο όπου ουσιαστικά προσφέρει ένα σύρο για έναν άλλο σύρο γιατί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο το σύστημα αυτό, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, πώς θα επιλέξουμε αυτή τη στιγμή ποιος θα αποφεληθεί του συστήματος και ποιος όχι και πώς μπορούμε να κάνουμε το σύστημα αυτό να λειτουργήσει χωρίς να στρεφόμαστε κατά του διεθνούς δικαίου και τι θα γίνει με όλες τις υπόλοιπες εθνικότητες, με τους υπόλοιπους υπηκόους που υποφέρουν εξίσου με τους Ήρους. Για όλα αυτά δεν δώσατε απαντήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ κακή και ελπίζω πραγματικά ότι θα αποτύχει γιατί αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι αλληλεγγύη υπευθυνότητα. Δεν θα πρέπει να παζαρεύουμε απλώς με γείτονες χώρες. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Δεν είναι μια τρίτη χώρα στην οποία μπορούμε να στείλουμε κατά αυτόν τον τρόπο πρόσφυγες. Άνεμανς, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην ε, ιδεολογία που ακολουθείτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, <clears throat> τα προβλήματα των προσφύγων δεν έχουν καμιά σχέση με το κράτος ευμάριας και την ενιαία αγορά. Εσείς έχετε διαπραγματευτεί με τους Τούρκους και έχετε συνδέσει το προσφυγικό θέμα με ζητήματα τελείως άσχετα, όπως παραγματικά χάρη η φιλελευθερωποίηση στις βίζες, τα δισεκατομμύρια που θα δώσετε στην Τουρκία και νέα κεφάλαια στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας. 3 δισεκατομμύρια και 3 δισεκατομμύρια 6 και ο πρόεδρος της φιλελεύθερης ομάδας μίλησε για την εξωτερήκευση της διαδικασίας υπολογής των προσφύγων. Εσείς έχετε οδηγηθεί σε μια σύγχυση αρχών και δέχεστε την ε, εκβιαστική στάση της Τουρκίας. Η πολιτική σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται πια ένας εφιάλτης. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε μπροστά μας μια Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια Ευρωπαϊκή μη ένωση. Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε. Εμείς ως εκπρόσωποι των λαών πρέπει να καταλάβουμε την οργή τους και την ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γκαρντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2015 πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα φτάσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 3.700 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Μεσόγειο από το Γιβραλτάρ μέχρι το Αιγαίο Πέλαγος. Ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε όλα αυτά. Είναι μια οπισθοδρόμηση συνεχής, θα έλεγα, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές και σε σχέση με τα γεγονότα τα οποία προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν τη μεταναστευτική κρίση. Εμείς σήμερα εδώ πέρα συζητάμε μια συμφωνία που λέμε τελικά ότι δεν μας αρέσει. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις λεπτομέρειες συμφωνίες αυτές, θα τις μάθουμε μετά τις 17-18 Μαρτίου. Παρ' όλα αυτά, εκ πρώτη όψεω δεν μα αρέσει το περιεχόμενο τη συμφωνία αυτή και πραγματικά έχουμε την εντύπωση ότι υποχρεούμαστε να κινηθούμε προς συμφωνία αυτή εξαιτίας του έκτακτου χαρακτήρα της κρίσης. Μα αυτό είναι απόλυτα ο λάθος θεωρώ, γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι εντελώ διαφορετική από αυτή που ήταν στο παρελθόν και νομίζω ότι φταίμε και εμείς γι' αυτό. Ως Ιταλίδα θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα τα οποία με δυσαρεστούν όλους ιδιαιτέρως. Εδώ και κάποια μήνες μιλάμε μόνο για το Αιγαίο Πέλαγος. Πολύ ωραία. Η συμφωνία μεταξύ Frontex και ΝΑΤΟ για την επίβλεψη των διαλέψεων. Για ποιο λόγο δεν μιλάμε όμως και για την κεντρική Μεσόγειο, για όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ισία, από τη Λιβύη. Στη Λιβύη έχουμε το ISIS. Και ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διακινητέ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο τμήμα αυτό της Μεσογείου πάρα πολλοί εκ των οποίων εμπλέκονται και στην ISIS. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια βραχυπρόθεσμη κοντόφθαλμη πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε αντίθετα μια μακροπρόθεσμη πολιτική και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταλέξουμε τελικά σε μια συμφωνία η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αποτυχία. Κυρία Γκαρντίνη, έχουμε μια μπλε κάρτα για σας, θέλετε να απαντήσετε. Δηλβέιος. το λόγο παρακαλώ. Μπορείτε να θέσετε το ερώτημά σας. Που Με... ερώτησή μου. Ήθελα να σα ρωτήσω, εάν οι Έλληνε, οι οποίοι θίγονται από, αυτά, από αυτές τις απαράδεκτες παραχωρήσεις που έκανε εχθέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδράσουν δυναμικά, ποια νομίζετε ότι θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ενδεχομένως βέβαια θα μου πείτε ότι αυτή είναι μια αφελής ερώτηση, γιατί η απάντηση είναι ότι δεν θα κάνει τίποτε. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι επάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Γκαρντίνη, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Κοιτάξτε, ενδεχομένω να μην κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σα. Πάντω, επαναλαμβάνω τα όσα είπα και θεωρώ ότι πραγματικά βρίσκονται στην ουσία τη απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Πρέπει να καταφέρουμε να είμαστε μία Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βγουν από τι εθνικιστικέ του πολιτικέ. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή εμεί να δώσουμε μία απάντηση αποτελεσματική απέναντι στο φαινόμενο αυτό αν ουσιαστικά αναδιπλωνόμαστε στι εθνικέ μα θέσει. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερωτησία και κατηδίαν θα μπορούσα να σας μιλήσω περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια πολύ, πολύπλοκη κατάσταση και δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει εύκολη και οριστική απάντηση. Ναι, πράγματι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε εμείς να συζητήσουμε με την Τουρκία. Είναι γείτονά μας, είναι ένας σημαντικός γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να διαλέξουμε ποιους έχουμε σε επίπεδο γείτονος, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, μια καλή σχέση γειτονίας, να έχουμε σεβασμό αμοιβαίο και να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι μεταξύ μας. Αλλά το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία και πώς θα αντιμετωπιστεί ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και τι έχετε να πείτε για την καταστολή στην Τουρκία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης. Και τι λέτε για μια χώρα η οποία αρνείται να λύσει ειρηνικά το θέμα των Κούρδων και κάνει πόλεμο στο ίδιο της το έδαφος. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όλα αυτά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την γείτονα αυτή χώρα και προς το συμφέρον της Ελλάδος που υφίσταται μια ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε αφελείς σε αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Μπάρεκοφ έχει το λόγο. Ναι, Βεβαίως αυτή η συμφωνία με την ε, Τουρκία είναι πολύ κακή συμφωνία διότι λέμε στην Τουρκία ότι τους δεχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεχθούν ε, τους μετανάστες μας. Η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη, το Ισλάμ δεν έχει τίποτα να κάνει με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ε, και εγώ διαρωτώ με γιατί κανείς δεν είπε στον Πρωθυπουργό ότι η επίθεση κατά των δημοσιογράφων είναι επίθεση κατά της ανθρωπότητας. Είναι κάτι που το βλέπουμε σε ολοκληρωτικά κράτη. Ο Ερντογάν είναι ο δημιουργός του προβλήματος του Ισλαμικού κράτους και τώρα τον θεωρούμε σωτήρα μας, αλλά νομίζω ότι αυτό το λάθος θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Δεν υπερασπιζόμαστε τα εξωτερικά μας σύνορα ε, και θα, θα, αυτοί θα καταστρέψουν τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν ήσαν ποτέ υπέρ και νομίζω ότι αυτή η βιασύνη με την οποία η Ένωση θα αφήσει από τον Ιούνιο να μπαίνουν ε, όλοι οι Τούρκοι χωρίς θεώρηση που το επιθυμούν και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Αρντογκάν του οποίου η μεγαλομανία, η ε, κακή πίστη είναι κάτι το απαράδεκτο. Βεβαίως αυτό το σχέδιο συμφωνίας που έχουμε επιτάπητος δεν μου αρέσει καθόλου και θα προσκρίσουμε σε σημαντικές νομικές δυσκολίες αλλά επειδή δεν έχουμε κάτι καλύτερο θα υποκύψω ακόμη και αν το τίμημα μου φαίνεται υπερβολικό και αν η Τουρκία είναι μάλλον εκβιαστής και όχι εταίρος. Το κάνω διότι είμαι πεπισμένος για δύο πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι αδύναμη. Μπορεί να καταρρεύσει αν έχουμε ακόμα δύο εκατομμύρια μετανάστες με μεγάλη αταξία αν φτάσουν ε, στα ελληνικά νησιά και προσπαθούν να περάσουν από τα σειρματοπλέγματα και δεν έχουμε το δικαίωμα να μετατρέψουμε φτιάξουμε ε, την Ελλάδα ε, σε ένα μεγάλο στρατόπεδο όπου θα υπάρξουν ε, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες μετανάστες με τις χειρότερες συνθήκες. κυρία Σπινέλη, ευχαριστώ πολύ ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, κάποια λόγια που ε, ξέφρασε πρόσφατα ο πρόεδρος ε, κύριος Τούσκ. Είπε στις 3 Μαρτίου ε, ότι οι πρόσφυγες δεν πρέπει να έρθουν στην Ευρώπη. All for nothing λες και είχαν επιλογή όταν έφευγαν και χτες είπε ότι πάνε πια οι μέρες της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Αυτό είναι λάθος και το γνωρίζει ο Τούσκ. Το 91% των προσφύγων στην Ελλάδα φεύγουν από, την, από τον πόλεμο και πηγαίνουν στην Τουρκία τους ε, κατηγορούν ότι είναι παράτυποι και ότι θα τους ε, επαναπροσθήσουν. Ε, αυτά όμως καταδικάζονται από την Διεθνή Αμναστία και από άλλες πολλές οργανώσεις. Ο Ερντογάν δεν λέει τίποτα για τη σφαγή στο Κουρδιστάν και για την επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας. Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τους Κουρδούς για δικό του όφελος. Οι πρόσφυγες έχουν ε, μια τραγική μοίρα και αυτό που τους απομένει είναι και η απαξίωση. Εμείς ε, αυτό το αποκαλούμε στα αγγλικά appeasement, απλά εφησυχασμό. Η κυρία Σαρτζεντίνη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ περίεργο ότι ήσασταν ε, εδώ ε, κατά το παρελθόν και ήσασταν εδώ. Αν λοιπόν ήσασταν εδώ θα χειροκροτούσατε αυτά που είπε ο κύριος Φεχόφστατ για το πόσο επονίδιστο είναι το πρόγραμμα αυτό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, πλέον ε, θα αναζητηθούν νέες οδοί μετανάστευσης και προσφυγιάς. Υπάρχει μια νέα πολιτική, έχετε και ένα νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Ρούτα, ο οποίος κύριος Ρούτερ λέει ότι πρέπει η μετανάστευση και οι μεταναστευτικές ροές να περιστούν στο μηδέν. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, θέλετε την ασφάλεια των προσφύγων ή μήπως ε, θέλετε να τους απομακρύνετε. Και άλλη μια ερώτηση. Η Τουρκία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Συρία. Σημαίνει άρα γι' αυτό ότι ε, θα έρχονται άνθρωποι μέσα από το Αιγαίο και όχι με τα αεροπλάνα. Ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μου επιτρέψετε μία παρατήρηση. Ε, πρέπει να σας πω ότι δεν χρειάζεται να σας ε, επισημάνω ότι υπάρχουν παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Τουρκία και εγώ παραμένω ε, να είμαι αντίθετο ε, με την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, τη συζήτηση αυτή σήμερα τη βρίσκω τρομακτική. Από τότε που μιλάμε για του πρόσφυγε, άκουσα πάρα πολλέ αιτιάσει ε, για το τι δεν πάει καλά. Πολύ σωστά, λοιπόν, συζητήσαμε για την Ουγγαρία και για του φράχτε και αυτά που κάνει και η Αυστρία. Πολύ σωστά. Μερικοί επικρίνουν την ιδιαίτερα ανθρωπιστική πολιτική τη κυρία Μέρκελ και σήμερα όλοι κριτικοί πια ασκούν, παρότι κατά την άποψή μου το μοντέλο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αποτελεί μια λύση που κάτι κάνει. Μια λύση η οποία μεριμνά έτσι ώστε οι πρόσφυγες ε, να έχουν ε, μια ασφαλή δίωδο. Ε, πάντα θέλαμε να έχουμε ένα περιορισμό στην Ευρώπη και το έχουμε ήδη πει αυτό και αυτή τη στιγμή όμως επιτέλους μοιάζει να έχουμε τη δυνατότητα να στριμώξουμε τους διακινητές. Δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση απόλυτη αποτελεσματική. Αν όμως τελικά ακολουθήσουμε αυτή την προτινόμενη λύση, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια ε, τομή, ε, μια πρόοδος ε, και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Κομισιόν που δούλεψε πάνω σε αυτό. Το να καταδικάζει κανείς τα πάντα και να είναι κατά των πάντων, αυτό δεν βοηθάει. Επιτέλους αυτή η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάτι πρόσφερε. Πολύ πολλοί επικρίνουν τους εθνικούς εγωισμούς. Ένα λοιπόν επιτέλους κάτι υπάρχει μια συνεννόηση. Εντάξει, δεν είναι ακόμα ε, τελική η αριθμή και εγώ προφανώς έχω κάποια ερωτήματα σχετικά με την απελευθέρωση των θεωρήσεων, όμως υπάρχει μια ευκαιρία και γι' αυτό ε, θέλω να παρακαλέσω το Συμβούλιο και την Κομισιό να συνεχίσουν να δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση και όχι μόνο αυτούς, ε, αλλά και συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει το χρόνο τους για να προχωρήσουν λιγάκι με την Τουρκία. Συνεχίστε λοιπόν, έχουμε κάνει το πρώτο καλό βήμα, επιτέλους το πρώτο καλό βήμα. Εγώ είμαι αισιόδοξο. παρά τα προβλήματα που είναι συνδεδεμένα με την Τουρκία και θα παραμείνουν, όμως ε, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει τίποτα ή κάνοντα το ένα πρέπει να αναιρέσει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρόιλ, τρεις μπλε κάρτες για σας. Από ό,τι φαίνεται σήμερα είσαστε ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ο Φλίν Φοντζούλη Γκραπίνη. Τρεις ερωτήσεις, τρεις μπλε κάρτες. Ο κύριος Φραντζούλικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, η συμφωνία αυτή με την Τουρκία έχει κατά τη γνώμη μου κάποιες καλές πτυχές και κάποιες λιγότερο καλές. Θα καταβάλουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με ακούτε κύριε Ρόιλ. Ακούτε αυτά που σας λέω κύριε Ρόιλ. Γιατί κάνατε, εν πάση περιπτώσει και οι λαθροδιακινητές ε, και όλοι οι άλλοι θα βρουν άλλους τρόπους να φέρουν τους μετανάστες στην Ευρώπη. Δεν πιστεύετε ότι σε τελική ανάλυση ε, ίσως θα χρειαστεί ένα ειδικό ε, δικαστήριο ε, ή ένα ειδικό σώμα για να φυλάσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ειδικό σώμα για, τα, για τη φύλαξη των εξωτερικών σύνορων. Κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε, είπατε ότι μείνατε ικανοποιημένο με τι ενέργειες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μια δημοσκόπηση όμω διάβασα ότι 52% των Ευρωπαίων ε, δεν καταλαβαίνουν ε, αυτή τη στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο πιστεύετε εσεί ε, ότι είναι ο καλύτερο τρόπο για να βγούμε από την κρίση και τι συμφωνία μιλάτε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι τα πράγματα είναι τέλεια. Είπα ότι υπάρχει κάποια μικρή πρόοδο. Ε, ε, άρα δηλαδή οι πρόσφυγες ε, μπορούν να έχουν μια ασφαλή δίωδο. Τρίτον, δεν θα υπάρχει ζήτηση για διακινητές. Ε, οι άνθρωποι δεν θα είναι αναγκασμένοι να μπαίνουν στα σαπιοκάραβα και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Δεν είναι τέλεια λύση, είναι όμως μια πρόοδος. Και οι δυνατότητες που εξετάστηκαν μέχρι σήμερα, δηλαδή ε, να κλείσουν τα σύνορα, να αναγερθούν φράχτες, αυτό ήταν μια πλήρης ανοησία. Αυτό που έχουμε τώρα είναι αδιαμφισβήτητα καλύτερα. Κύριε Ρόλ, έχετε ο κύριο Φλάναγκαν. Ο κύριος Ρόιλ είπε ότι δεν είναι τέλεια η συμφωνία. Φυσικά τίποτα δεν είναι τέλειο. Και είναι δύσκολο να πετύχουμε την τελειότητα. Πάντως, το να έχουμε ε, δοσοληψίες με τον ηγέτη μιας χώρας που ε, ε μίλησε υπέρ της διακυβέρνησης ε, και της δομής της εξουσίας του Αδόλφου Χίτλερ Εντάξει, τελειότητα δεν επιδιώκουμε, αλλά τουλάχιστον κάποιες υψηλότερες προδιαγραφέ από το να έχουμε παρεδώσει με έναν τέτοιον άνθρωπο. Κοιτάξτε, προφανώ και εμένα όλα αυτά με ενοχλούν. Αλλά ξέρετε, μερικέ φορέ πρέπει κανεί να βρει κάποια λύση. Τι να κάνουμε, να συνεχίσουμε όπω κάναμε μέχρι τώρα, να του αφήνουμε να πεθαίνουν, να πνίγονται και να μην βρίσκουμε καμία λύση απλά και μόνο γιατί θέλουμε να παραμείνουμε ηθικολόγοι. Όχι κάθε άλλο. Η δουλειά μα είναι να βοηθάμε συγκεκριμένα και μερικέ φορέ είναι κανεί αναγκασμένο να καταφύγει και σε λύσει που δεν του είναι αρεστέ. Ο κύριος Φλέκενστάιν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Ρόιλ, πρέπει να σας πω ότι κάπου με αυτά που είπατε έχετε δίκιο, γιατί και εγώ για πρώτη φορά ελπίζω ο κύριος Τούσκ να παίξει το ρόλο του συντονιστή, το ρόλο του διευθυντή ορχήστρας για να παίξουν όλοι μέσα στην ορχήστρα. Αλλά το θέμα είναι τι μουσικό κομμάτι θα ανεβάσουν. Οι υπόλοιποι βέβαια έχουν δίκιο και αυτοί με την κριτική τους γιατί ξέρετε κάτι πρέπει να είμαστε και λιγάκι ρεαλιστές. Πράγματι και εγώ πιστεύω ότι κάπου μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία όμως ελπίζω ότι σύντομα θα επιλύσουμε τα ανοιχτά θέματα, θα έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος δράσης, ποιος θα πάρει πόσα χρήματα. Επίσης πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπονομεύεται η προσπάθεια προσπάθεια να υπάρχει καταγραφή των προσφύγων. Είναι σαφές ότι πρέπει να επικρίνουμε την Τουρκία για θέματα ελευθεροτυπίας και να της πούμε ότι περιμένουμε από εκείνη να ε, αποδώσει και πάλι πίσω ε, την ιδιοκτησία της εφημερίδας ε, στους ιδιοκτήτες. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες στη μοίρα τους. Ούτε και τους Τούρκους γιατί θέλουν μεγαλύτερη ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ συμφωνώ με το να ανοίξουν και άλλα κεφάλαια με την Τουρκία. Αν όμως δεν συμπεριλαμβάνονται τα ε, κεφάλαια 23 και 24, εγώ να σας πω κάτι, δεν θα σας στηρίξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόλμελ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, σκεπτόμενος αυτή τη συνάντηση κορυφής με την ε, Τουρκία, σκέπτομαι το εξής. Όταν κάποιος συμφωνεί σε επίπεδο αρχής σε κάτι δεν έχει καμία δυνατότητα να αλλάξει λεπτομέρειες. Αυτό ισχύει και γι' αυτό αυτή η υποτιθέμενη συμφωνία δεν περιέχει λεπτομέρειες. Δηλαδή τελικά δεν ξέρουμε τι ακριβώς ε, θα επιπέσει επί της κεφαλής μας. Όμως αυτή η μεγάλη κρίση απαιτεί επιτέλους να γίνουμε συγκεκριμένοι. Δεν χρειαζόμαστε τις ε, μεμονωμένες ψηφίδες του μοσαϊκού, αλλά ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει το πόσους πρόσφυγες είναι πρόθυμοι να δεχτούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το κομπικό σημείο. Όποιος αποφεύγει αυτή την ερώτηση δεν θα βρει ποτέ ικανοποιητική λύση. Η βοήθεια είναι προαιρετική, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόση βοήθεια επιθυμούν να προσφέρουν. Όλα τα άλλα είναι φαρισαϊσμός. Και φοβάμαι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι, οι κακόμοιροι που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους, τους αξίζει κάτι καλύτερο από φαρισαϊσμό. Και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτοί έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Σας παρακαλώ τερμά από κοινού να αγωνιστούμε για ένα συνολικό πακέτο. Ο κύριος Άλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά τις ε, συνολικές εξελίξεις των σχέσεων με την Τουρκία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι ως προσωρινό, αλλά στρατηγικό, αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Επίσης θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε αμοιβαίως εποφελή συνεργασία. Υπάρχει παγκοσμιοποιημένη κατάσταση και διασύνδεση. Είναι πολυδιάστατη η κρίση και για να επιβιώσουμε ε, χρειαζόμαστε στενές και φιλικές σχέσεις με τους εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Τουρκίας στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης ε, είναι απαραίτητος. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Τουρκία. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως και από αυτή την άποψη δεν είναι παραγωγικό να επικεντρώνουμε την προσοχή μας μόνο ε, στην ε, κατανομή των κονδύλιων μόνο στο οικονομικό σκέλος. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε το κοινό σχέδιο δράση με την Τουρκία το συντομότερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας ευρωπαϊκά σύνορα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια ενωπημένη θέση με την Τουρκία και από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις. Θα πρέπει να κάνουμε εξαγωγή της ασφάλειας. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε μονίμως εισαγωγή της έλλειψης ασφάλειας, της ανασφάλειας. Ο κύριος Φεραίρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Αυτό που συνέβη στη Σύνοδο Κορυφής με την Τουρκία και αυτό που θα συμβεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, μας επαναφέρουν σε μερικές από τις πιο μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Έχουμε μια ανθρωπιστική τραγωδία που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και μάλιστα εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άμεσες και έμεσες ευθύνες απέναντι σε εκατομμύρια ανθρώπου που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, την πείνα, την εξαθλίωση. Και εμεί στηριζόμενοι στην μηχανή του πολέμου του ΝΑΤΟ απαντά με εκφοβισμό, με εξευτελισμό, με ενοχοποίηση, ποινικοποίηση και απέλαση μεταναστών και προσφύγων. Ε, ενώ ε, αντί να ε, έχουμε ε, ηθικές και δοντολογικές αρχές δείχνουμε την παρακμή μας, τη ρατσιστική, αντιδημοκρατική και μυσαλόδοξη όψη μας. Νομίζω ότι αν δεν αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία, όλα αυτά μπορεί να μας έρθουν μπούμεραγκ στο εγγύς μέλλον. Γιατί οι αποφάσεις αυτές θα ξαναγκάσουν ε, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βρουν πιο επικίνδυνους ακόμη τρόπους για να διέλθουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να επαναπαυθούν. Και σίγουρα αυτές οι τραγωδίες δεν θα πρέπει να μείνουν γιατί υπάρχουν πολιτικοί ηθήνοντες για αυτά θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες. Ο κύριος Μπιουτικόφερ. Η ε, ονομαζόμενη προσφυγική κρίση κατ' ουσία είναι κρίση της ευρωπαϊκής συνοχής, ευρωπαϊκής αυτοπεποίθησης και ευρωπαϊκής ε, ανθρωπιάς, ε, ανθρωπισμού αν θέλετε. Η συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία 7 Μαρτίου δεν επέφερε καμία αλλαγή, η κρίση συνεχίζεται και στη συζήτηση ε, μας το έδειξε αυτό ο κύριος Ντομπρόψκης, ο αντιπρόεδρος, ε, ο οποίος είπε ότι ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να ε, τεθεί το θέμα επιτάπητος. Το ίδιο είπε και η εκπρόσωπος της Ολλανδικής Προεδρίας, η οποία μάλιστα ούτε καν χρησιμοποίησε τις λέξεις πρόσφυγας και άσυλο. Αυτή μίλησε μόνο για παράτυπους μετανάστες. Ξέρετε, η γλώσσα μπορεί να φέρει και ελευθερία, αλλά μπορεί και να ασκήσει και βία η κυρία ε, βλέπει ότι υπάρχουν μόνο παράτυποι μετανάστες, προφανώς επιλέγει τη δεύτερη λύση που σας είπα προηγουμένως. Η ανθρωπιά όμως αφορά όλους και αυτό το πέτυχε η κυρία Μέρκελ. Είναι μια Ευρώπη η οποία αρνείται να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις, ε, να αναλάβει την ευθύνη της. Μια Ευρώπη που χάνει τη δυνατότητα να επηρεάσει καταστάσεις. Είναι μια Ευρώπη που με τον τρόπο αυτό χάνει και την ηθική της υπόσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαλπέτς, παρακαλώ. Η κυρία Γκαλπέτς, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Ντομπρόφσκι, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, είπε ότι λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο οι ψηφοφόροι μας θα αξιολογήσουν τις συνέπειες. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουν οι ψηφοφόροι μας. Ζούμε τη μία κρίση μετά την άλλη. Οικονομική, δημογραφική, προσφυγική κλπ. 4,5 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω των 25 ετών. Και ταυτόχρονα έχουμε και την προσφυγική κρίση. Έχουμε λοιπόν πολλά παραδείγματα που μας οδηγούν να πούμε ότι ε, έχουμε κάνει βήματα αντιμετώπιση ορισμένων από αυτέ, για παράδειγμα την οικονομική κρίση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για παράδειγμα, μα ε, δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι χώρε και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ουγγαρία ε, έχει ε, επιδείξει πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα τελευταία με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ε, ενώ σε ό,τι αφορά την Διεθνή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ουγγαρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, την μεταναστευτική κρίση, νομίζω ότι η συμφωνία της Δευτέρας δεν είναι τέλεια, αλλά συμφωνώ με τον κύριο Ρόιλ δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις, μην κρινιάζουμε μόνο, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα σύνορα, πρέπει να κλείσουμε σύνορα, όπως είπε ο κ. Βέμπερ αν χρειαστεί. Υπάρχουν όμως και άλλα εκκρεμή θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων ή της διευκόλυνσης των θεωρήσεων. Γιατί δεν μιλάμε για την Ουκρανία. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα επίσης του ότι ε, για ένα σύρο που θα μπαίνει στην Ευρώπη ένας θα πρέπει να επιστρέφεται στην ε, Τουρκία. Πού υπάρχουν εγγύσεις ότι θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα κονδύλια με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Ε, θέλουμε μακροπρόθεσμες λύσεις, όχι βραχυπρόθεσμες. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε ένα καλό βήμα όμως. Ευχαριστώ. Υπάρχει μπλε κάρτα για σας κύριε Γκαλπέλτς. Ε, τη δέχεστε? Και ο Σουγέντη, αλλά να πω το εξή. Οι μπλε κάρτες ε, είναι για να θέτετε ερωτήματα. Γιατί πολλά μέλη ε, χρησιμοποιούν την μπλε κάρτα για να μιλήσουν απλώς. όχι, η μπλε κάρτα είναι για μια ερώτηση σε κάποιον που έχει ήδη λάβει το λόγο, έτσι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θέλω να ρωτήσω τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος του κ. Ορμπάν. Ο, ο, ο κ. Ορμπάν πριν τη συμμετοχή του στη Συνοκορυφή, είπε ότι δεν θα πρέπει η Ουγγαρία να γίνει Ευρώπη. Τι θα πει αυτό. Να γίνει σαν την Ευρώπη δηλαδή. Τι θα πει αυτό. Μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο του Πούτιν. Απάντηση. Ο πρόεδρος ε, σας προειδοποίησε. Ε, δεν ήξερε τι ερώτηση θα κάνετε. Ε, ίσως θα έπρεπε να ακούτε πρώτα τι λέω και μετά να κάνετε τις ερωτήσεις σας κάνατε την ερώτηση που, ε, που θα θέλατε να θέσετε στον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και επειδή δεν μπορείτε την κάνετε σε μένα. Νομίζω ότι η Σύνοδος Κορυφής Δευτέρας είναι ένα θετικό βήμα, Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προστατεύουμε τα σύνορα της Ευρώπης, τα κλείνουμε. Είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Αντί λοιπόν να κάνουμε ανεύθυνες δηλώσεις, καλό είναι να, να προστατεύουμε την Ουγγαρία προς όφελος των πολιτών της. Εγώ μίλησα για μια κατάσταση πριν το 2010 που μας έφερε στη σημερινή συγκυρία. Ευχαριστώ. Κύριε Πύρη, καταρχήν το αυτονόητο. Η Ευρωπαϊκή και η Ένωση και η Τουρκία χρειάζονται μια την άλλη για να βρουν μια κοινή λύση στο προσφυγικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε τις ροές. Ε, Απλά θα πρέπει να το μετριάσουμε έτσι ώστε ε, όσοι χρειάζονται ε, βοήθεια και προστασία να τη βρουν και οι οικονομικοί πρόσφυγε να επιστρέφονται. Η πρόσφατη συμφωνία δεν αποτελεί επαρκή απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Πώς 28 ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπέβαλαν ένα πρόγραμμα στο οποίο νόμιμε οδοί για πρόσφυγες υπάρχουν μόνο αν ε, κάποιοι άλλοι επιστρέφονται. Ε, αυτό είναι, ε, παραβιάζει το διεθνές ε, δίκαιο αλλά και την ηθική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ αδυναμή θέση γιατί διατηρεί ένα μονοδιάστατο διάλογο με την Τουρκία που βασίζεται μόνο στον αριθμό των ατόμων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά κάθε μέρα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λένε θα έρθουν αργότερα. Αυτό είναι λαθασμένη στρατηγική και ιδιαίτερα την στιγμή που η Τουρκία παραβιάζει το κράτος δικαίου και επιτίθεται στους δημοσιογράφους. 255.000 Κούρδοι πολίτες έχουν, ε, της Τουρκίας έχουν φύγει από τα έχουν καταλήψει αιστείες τους λόγω της έκρηξης βίας που ε, έχει γίνει το τελευταίο καιρό εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να κοιτάει αλλού όταν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ε, το, ε, μην ξεχνάμε ότι θα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πραγματική δίκαιη κατανομή του βάρους με τους Τούρκους πολίτες που έχουν ήδη φέρει σημαντικό βάρος τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Πιοτρόφσκι, παρά τις ε, διπλωματικές αναγγελίες στην τελευταία σύνοδο κορυφής, η σύνοδος αυτή ήταν μια φρα... αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησε την Τουρκία να, την... να... να τη βγει από πάνω και φαίνεται ότι έτσι θα τελειώσουν ε, οι μεταναστευτικέ ουρέ, όπω είπε ο κύριο Τούς και ο κύριο Γιούνκερ είπε ότι στέφθηκε με επιτυχία η Σύνοδο Κορυφή, ότι ήταν πραγματική επανάσταση αυτή που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι για τίποτα σίγουρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προσπαθεί να πείσει την Τουρκία να ε, ε, συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο παζάρι με δισεκατομμύρια και προσπαθεί έτσι να σώσει τη μεταναστευτική της πολιτική ε, προσφέροντας και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η Τουρκία πέτυχε αυτά που ήθελε, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στριμωγμένη στον τοίχο. Επίσης, είπαμε την επιτάχυνση των ανταλλαγών ένας προς ένας. Ε, τι γίνεται, τι θα γίνει με αυτές τις ε, αλλαγές, ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την συμφωνία που έγινε. Ο κύριος Βάγκλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το θέμα των προσφύγων, μεταναστών και ετούντων άσυλο είναι πια όχι μόνο ηθικό θέμα, όχι μόνο θέμα συμπόνιας, ε, για τα δεινά που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είναι ένα ζήτημα που μας φέρει ε, ενώπιον των ηθικών και των πολιτικών μας ευθυνών. Είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε καθήκον να παραμείνουμε ενωμένοι και να γίνουμε αποτελεσματικοί στην Ευρώπη. θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και φυσικά να αναγνωρίσουμε το ρόλο κλειδί που παίζει η Τουρκία στην κρίση αυτή. Φυσικά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το αυταρχικό καθεστώς του Ερδογκάν και τις συλλήψεις δημοσιογράφων ή τις πιέσεις που ασκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε και σήμερα και στο μέλλον την Τουρκία ως εταίρο μας. Και η συμφωνία αυτή δεν είναι ένα οικονομικό παζάρεμα. Αφορά τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα εταίρο που ε, λογικό είναι να επιδιώκει τα δικά της ε, συμφέροντα. Η Ευρώπη αποσαφήνισε την θέση της και τη συμπεριφορά της απέναντι ε, στην Τουρκία και στο παρελθόν. Και σίγουρα δεν είναι αυτή η κρίση η κατάλληλη στιγμή για να το κάνει τη συμφωνία αυτή έτσι ώστε η Τουρκία να αποτελέσει τον τείχο της Ευρώπης ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για 6 δισεκατομμύρια ευρώ πουλάμε τόσους ανθρώπους πόσο αξίζει ο καθένας 1000, 2000, 3000 ευρώ Ποια είναι η τιμή του κατά κεφαλή. Ε, τους καταδικάζουμε ε, να επιβιώσουν σε μια μαύρη τρύπα. Τι θα συμβεί με αυτούς. Κανείς δεν ξέρει. Εμείς πληρώνουμε και αν τους ξεχάσουμε. Α του έχουν εκεί να ζουν σε απάνθρωπες ε, συνθήκε, να επιστρέψουν στην πείνα, στον πόλεμο ή τέλο πάντων να του καπνίσει. Εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό και η Τουρκία αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Οπότε η Τουρκία θα λειτουργήσει ως ε, σύνορο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να κοιτάει προς μια άλλη κατεύθυνση ενώ οι Κούρδοι δολοφονούνται ε, εκεί στο νότο της Τουρκίας. Παραβιάζουν τις συνδεσμάσεις της Γενέβης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανθρώπους από τη Συρία, το Σουδάν και το Αφγανιστάν πρόσφυγες και να τους, να τους επιστρέφουμε στην Τουρκία. Είναι παράνομο. Παραβαίνει τις, ε, διεθνείς, κανόνες ανθρωπιστικού δικαίου και ελπίζω όσοι το υπογράψουν αυτή τη συμφωνία κάποια στιγμή να δικαστούν. Πιστεύω ότι Μόνο μια ε, ευρωπαϊκή λύση με όλους τους συμμετέχοντες θα μας ε, βγάλει από το διέξοδο. Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του προγράμματος. Ε, η συμφωνία αυτή έχει πολλές αδυναμίες, το είπε και ο Σβέμπερα, είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι για τις αρχές μας και με εκπλήσει που η συζήτηση γίνεται μόνο για τα χρήματα. Τα χρήματα που θα δώσουμε για τους πρόσφυγες στην Τουρκία είναι σημαντικά. Χρειάζονται, αν μοιραστούν σωστά. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί τμήμα απλώ του όλου σχεδίου. Ε, κλείνουμε, αν κλείσουμε τη Βαλκανική οδό, οι άλλε οδοί θα χρησιμοποιούν περισσότερο. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να μιλήσουμε λίγο και για την οικονομία. Γιατί αναφέρθηκε ο κ. Ντομπρόφσκι σε αυτήν. Η κατάσταση τη παγκόσμια οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ασφαλώ θα πρέπει να μα απασχολεί. Και να μα απασχολεί και η κατάσταση στην Κίνα. Το πιο σημαντικό όμω για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι η εσωτερική κατάσταση. Η σταθερότητα της εσωτερικής ζήτησης και επενδύσεις. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ε, τις προτεραιότητές μας ανάπτυξη και απασχόληση ε, καθώς επίσης και ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες μας, συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή έχει την πλήρη στήριξή μου στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τέλο, κάτι που δεν βρίσκεται στη μέση διάταξη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Ε, γίνονται σειράξει, οι ζωέ των ανθρώπων απειλούνται, αποτελεί μια πηγή αστάθεια πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Στην πολιτική μας μην περιμένουμε ότι θα μαλοποιηθεί ε, η κατάσταση στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος. Η ε, κυρία Γκυγιόμ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ακούσαμε για να χαρακτηρίσουμε τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Τουρκία. Οι περισσότεροι λένε είναι όρο και δεν και εμεί. Ε, άλλοι, η Τουρκία είναι τμήμα τη λύση και θα πρέπει να συμμετέχουμε. Βέβαια, θα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα τι συνέπειε αυτών τον προσανατολισμό και των καθευθυντηρίων γραμμών. Ε, καταρχήν, ποιε είναι η συνέπειε του κλεισίματο τη Βαλκανική Οδού. Κακό ο υπολογισμό των κρατών μελών. Γιατί καταρχήν ε, βάλαμε τη, σε τεχνητή βοήθεια την ε, Ελλάδα, αλλά τι θα γίνει με το Σέγγεν. Ε, ουσιαστικά εγκρίνουμε τι μονομερεί αποφάσει για τα κλεισίματα των συνόρων. Επίση, συνεργασία με την Τουρκία. Σίγουρα είναι αναπόφευκτο εταίρο ε, και η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη. Αλλά θα πρέπει να βρούμε αλλού λύσει. Και πρώτα απ' όλα να βρούμε τις λύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ όχι μόνο υποκύπτουμε στις απαιτήσει ε, της Τουρκίας, αλλά με κάποιους πληστηριασμούς αστικά και δημοπρασίες κάνουμε υπεργολαβία των ευθυνών μας ε, ε, και το έργο μας στην Τουρκία. Και τι γίνεται με την αρχή της αλληλεγγύης. Επίσης, ό,τι αφορά την επανεκατάσταση των σύρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση η ανταλλαγή ένας προς έναν. Αυτή η, ανταλλαγή είναι πραγματικά ανέντιμη. Ε, δηλαδή, ένα σύρος θα κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή του να πνιγεί, ε, προκειμένου ένας άλλος να βρει μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι αμφίβολης ε, εγκυρότητας και ε, η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Επίσης, τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι είναι έτοιμα να στηριχθούν σε κάποιες αξίες και να εθελοτυφλήσουν στην αυταρχικότητα του τουρκικού καθεστώτος, στις συλλήψεις των δημοσιογράφων, στο κλείσιμο των πανεπιστημίων και στις απειλές στο δικαστικό σύστημα. Και υπό το πρόσχημα μια κοινή λύση, η ιδέα μια αλληλέγγυα και υπεύθυνη Ευρώπη φαίνεται ότι βαδίζει προ την αποτυχία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τρεμπέζιος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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μέρκελ είχε δίκιο. Δηλαδή διαφαίνεται ευρωπαϊκή λύση, βέβαια όχι λύση εκείνη που είχε κατά νου η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τέλο σε αυτή την πολιτική του περάστε όλοι. Πολλά κράτη κατέσθησαν σαφέ ότι Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τέλος σε αυτή την πολιτική του «περάστε όλοι». Πολλά κράτη κατέστησαν σαφές ότι η Γερμανία είναι απομονωμένη με τη στάση της. Έτσι λοιπόν η κυρία Μέρκελ, η οποία μόνη της το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους άνοιξε τα σύνορα, τώρα επιπλήττει την Αυστρία, αλλά τουλάχιστον η Αυστρία βρήκε μια συμφωνία. Τα κουμπέντιασε με τις άμεσα θυγόμενες ε, χώρες και περιοχές. Τώρα λοιπόν υποτίθεται η Τουρκία θα προστατεύσει τα σύνορα. Το γεγονός λοιπόν ότι εξαρτώμεθα και δεχόμεθα εκβιασμούς από μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη δημοκρατία, ούτε με τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά ούτε και με την ελευθερία του τύπου, ε, το να ξεκινήσουμε με αυτή τη χώρα ε, ενταξιακέ διαπραγματεύσει, αυτό μα αφήνει εννοού. Έτσι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Γερμανία απλά αγνοεί τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας. Και τι το ερώτημα, εδώ διακυβεύονται μόνο γερμανικές ή μήπως και ευρωπαϊκές αξίες. Καλούμε άλλους να πράξουν αυτά τα οποία δεν θέλουμε να πράξουμε μόνοι μας. Κοιτάξτε, αν είναι έτσι τα πράγματα, με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη δεν έχει κανένα μέλλον. Επόμενος ομιλητής... Ο κύριος Αρτουή. Όταν ε, έφτασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Ίσως περίμενε να συναντήσει τις κυβερνήσεις Ευρώπης. Αλλά ε, προσγειώθηκε μέσα σε ένα μεγάλο παζάρι. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεών μας φάνηκαν ανίκανοι να αποφασίσουν και προτίμησαν το παζάρεμα. Και μετά τον εκβιασμό του David Cameron που απείλησε με το ένα πόδι μέσα, ένα πόδι έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ήταν ο εκβιασμό τη Τουρκία ε, για να βάλει ένα πόδι όμω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, ποια ήταν τα αποτελέσματα το Ευρωπαϊκό Σώμα Συνοριοφυλακής και Ακριτοφυλακής ε, και η κεντρική διαχείριση των ε, αιτήσεων άσυλου. Ακόμη τα περιμένουμε αυτά. Επίσης, ε, συνθήκες επανεισδοχής ε, σε τρίτες χώρες. Ε, δεν έχουμε ούτε καν ε, στα σπάργανα μια εξωτερική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε αξιόπιστα τη σύγκρουση στη Συρία. Τρία δισεκατομμύρια για την Τουρκία. Πώς θα δώσουμε όμως στο Λίβανο ή στην Ιορδανία ή μετά για την ανασυγκρότηση της ε, Συρίας. Ντρέπομαι για αυτή την Ευρώπη, ντρέπομαι για την εικόνα αδυναμίας και ανιγανότητας που δείχνουμε απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να ξανα κατακτήσουμε τη θέση μας στην ιστορία. Και μάλιστα η επόμενη διάσκεψη κορυφής, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι ένα ιστορικό ραντεβού από αυτή την άποψη. Κύριε Ραντζέλ, ε, σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που έχει προβλεφθεί για σας, γιατί στη μία η ώρα το μεσημέρι προβλέπεται η ψηφοφορία. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, ε, ο, καθήκοντά του ο πρόεδρος της ε, Δημοκρατίας ε, στην Πορτογαλία και ε, ανέφερε ποιε είναι οι αρχές οι οποίες ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε στο μέλλον. Είναι οι ανθρωπιστικέ αρχέ. Είναι οι αρχέ επίση που σχετίζονται με την ταυτότητα τη Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποδεχόμαστε να υποδεχθούμε ε, ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Ε, και χαίρομαι που ελήφθησαν μετά σε αυτή τη συμφωνία έτσι ώστε η Ελλάδα να καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της. Και δεύτερον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ΝΑΤΟ ε, έτσι ώστε να εγγυηθούμε των ελχών των συνόρων. Το Συμβούλιο της 17ης και 18ης όμως πρέπει κυρίως να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας μιας ε, ευρωπαϊκής ε, συνοροφυλακής και ακτοφυλακής. Είναι το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση ασφάλειας στην Ευρώπη. Στο, τελευταία δημοσ... σε μια τελευταία δημοσπρόσφατη δημοσκόπηση αναφέρεται ότι το 79% των Ευρωπαίων είναι υπέρ της δημιουργίας μιας ε, ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης για την προστασία των ακτών και των συνόρων ε, και ζητούν μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης όχι μια εθνική πολιτική ούτε μια ε, ε, επιμερισμένη πολιτική. Θέλουν μια κοινή πολιτική των 28, όχι 2, 3, 4 χωρών. Μιλάμε για πλειοψηφία 70-80% των ατόμων σε όλη την Ευρώπη που το ζητούν. Ακόμα και στις χώρες που είναι ε, ε οι πιο διστακτικές όπως οι χώρες του Βίσεγκράτ. Ε, και εκεί η πλειοψηφία είναι 55-60%. Με τέτοια υποστήριξη τη κοινή νόμη, πιστεύω ότι το επόμενο Συμβούλιο Κορυφή δεν έχει κανένα λόγο για να αποφύγει να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα ε, υπέρ των αρχών μα, ε, των ανθρωπιστικών αρχών και υπέρ τη ασφάλεια. Ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διχασμένη Ευρώπη, η αδύναμη Ευρώπη διαπραγματεύεται με την Τουρκία υπό άνισος όρους. Πρόκειται για μια συμφωνία για να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, αλλά ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Η εξωτερική κατάσταση, ε, αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι για να αποφύγουμε τις ευθύνε μας. Η συμφωνία είναι πολύ κρίσιμη, έχει πολλές αμφισημίες, υπάρχει η ιδέα του να επιστρέψουν αυτοί οι πρόσφυγες. Ε, το Συμβούλιο δεν μοιάζει να ε, προσέχει ακριβώς τι διαδραματίζεται. Ε, υπάρχει αίτηση ασύλου από τους καταβλισμούς της Τουρκίας. Αυτό μπορεί να λάβει η χώρα μόνο εφόσον όλα αυτά γίνονται κάτω από την ευθύνη της Ευρώπης. Ε, οι ευρωπαϊκοί και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να διαρματίσουν σημαντικό ρόλο. Αγαπητοί εκπρόσωποι της Ολλανδίας και της Προεδρίας του Συμβουλίου. Αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να αφορά όμως τους πρόσφυγες που έχουν έχουν ήδη φτάσει στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να επιστρέψουν στην Τουρκία οι πρόσφυγες που μετά από την κόλαση έφτασαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ε, απάνθρωπο, είναι ενάντιο σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία. Είναι σαν να λέμε ε, στα παιδιά ότι ε, ναι, μπορεί να κερδίσετε, αλλά ξεκινήστε από την αρχή. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ με μια τέτοια λύση. Ο Ζαχραντήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια για τη Σύνοδο Κορυφής. Να ξεκινήσω από το θετικό. Χαίρομαι που βλέπουμε μία προσπάθεια να διαχωρίσουμε τους Σύρους από τους λοιπούς πρόσφυγες και κυρίως να διαχωρίσουμε αυτούς που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο από τους οικονομικούς μετανάστες γίνεται επιτέλους μια προσπάθεια να γίνει κάτι για όσους βρίσκονται στην Τουρκία και να αποτρέψουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους να πάρουν το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, είναι λογικό να πρέπει να πληρώσουμε κι εμεί ένα τίμημα γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τον κόσμο στι αιστείε του, για να μην ξεκινήσουν να συνεχιστούν νέε μαζικέ ροέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, προ την Ευρώπη. Επίσης υπάρχει η απόπειρα αυτής της ανταλλαγής ένας προς ένα. Δηλαδή όσοι επιστρέφονται στην Τουρκία να αντικαθιστούνται από αυτούς που θα αποστέλλονται από, την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βέβαια, αυτά είναι όλα κάποια τεχνάσματα υπό το φύλλο της αλληλεγγύης και των κοινών λύσεων και κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Κυρία Σόμερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και έχουμε και τους ε, σχετικούς νόμους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόθυμα να τηρήσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, επί το οποίο και οι ίδιοι και τα ίδια αποφάσισαν. Αρνούνται τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν και το διεθνές δίκαιο και μόνο αυτό το αγνοούν επιπλέον. Γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση στο προσφυγικό. Και τώρα πλέον λόγω όλων αυτών εξαρτώμεθα από την προσφορά της Τουρκίας να συγκρατεί, να δέχεται πίσω τους πρόσφυγες ακόμα και να του ανταλλάσσει. Μα αυτό το πρόγραμμα είναι άραγε συμβατό με το διεθνές δίκαιο και τι εικόνα εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα εκπέμψει αν τελικά επικρατήσει αυτή η συμφωνία. Μία ε, φτωχή θα τη χαρακτήριζε εικόνα αλλά αυτή τη φτωχή εικόνα ε, την δημιούργησαν τα ίδια τα κράτη-μέλη τα οποία αρνήθηκαν να εφαρμόσουν ε, μια πολιτική αλληλέγγυα. Τώρα, για πρώτη φορά θα ονοματίσω την ε, Αυστρία, η οποία προκάλεσε ολόκληρη αλυσίδα αντιδράσεων με την άρνησή της να δεχθεί αυτούς τους ε, πρόσφυγες. Αρνείται να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως η Τουρκία ζητάει ανταλλάγματα. Ε, και εμείς το ίδιο θα κάναμε, αν ήμασταν στη θέση τους. Όμως, αγαπητοί φίλοι, τι σημαίνουν άλλα 3 δις Μπορεί να σας μοιάζουν πολλά. Αλλά αν σκεφτείτε πόσα λεφτά έχουμε δώσει για την Ελλάδα, τα 6 δις δεν είναι τίποτα σε σχέση με όσα έχουμε ήδη εκμεταμιεύσει. Και τα 6 δις δεν είναι τίποτα αν τελικά σκεφτούμε ότι θα έπρεπε εμείς να πάρουμε τους πρόσφυγες. Εντάξει, δεν είναι καλή αυτή η λύση το να πρέπει κανείς να καταβάλει χρήματα για να παραμείνουν οι πρόσφυγες εκτός Ευρώπης. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν μπορεί να γίνει αλλιώ και οι δεξιοί λαϊκιστές ε, και αυτοί ε, μέχρι τώρα αφιόνισαν τις κυβερνήσεις τους ε, και το τραγικό είναι ότι ε, σε κάποιες χώρες είναι μάλιστα τα κόμματα αυτά και στην κυβέρνηση. Οι δεξιοί, οι ακραίοι είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει την κρίση και εγώ ντρέπομαι για αυτά στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο έχει ως καθήκον η συμφωνία να κλείσει με την Τουρκία γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μόνη διέξοδος η λύση ευπατή με τις αξίες μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρί εμά δεν θα υπάρξει απελευθέρωση των θεωρήσεων, δεν θα υπάρξει ένταξη της Τουρκία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και εμείς έχουμε ευθύνε και αρμοδιότητες. Η κυρία Ζίπελ. Εμείς τι κάνουμε με τους πρόσφυγες, εκτός της Ευρώπης ε, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν ασφαλείς θέσεις ε, για τους πρόσφυγες ε, αλλά αυτά που έγιναν τη Δευτέρα ενίσχυσαν την άποψη ότι η Ευρώπη κλείνει τα σύνορά της κλείνει η Βαλκανική οδός, οι πρόσφυγες θα επιστραφούν πίσω στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται η εγκατάσταση των προσφύγων από την Τουρκία προς την Ευρώπη είναι σε απόλυτη εκκρεμότητα. Ευρωπαϊκά κράτη μας εκβιάζουν και αυτό το εκμεταλλεύεται η Τουρκία και ξέρετε γιατί. Διότι η πολιτική κρατών μελών είναι εκείνοι οι οποίοι μετακινούνται προς τα δεξιά αντί να ταχθούν ανεπιφύλακτα υπέρ της δημοκρατίας των ανθρωπίνων και υπέρ όλων εκείνων των πολιτών οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν στους πρόσφυγες. Η επόμενη συνδιάσκεψη κορφής πρέπει να προσφέρει αποτελέσματα, να είναι υπέρ μιας ανθρώπινης πολιτικής, υπέρ της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή, αυτό το καιρό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχε θετική επίχυση η είδηση για τη συμφωνία ότι κλείνει η Βαλκανική οδός γιατί η Κροατία είναι στο, στη Βαλκανική αυτή διαδρομή αλλά ας μην ξεχνούμε και την ανθρωπιστική τραγωδία. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όταν έχουμε μπροστά μας αυτό το ανθρώπινο δράμα. Επίσης ε, είπε ο κύριος Τούσκ στους ε, ε, πρόσφυγες μην πιστεύετε στους λαθροκινητές, μην έρχεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ όμως μιλούμε για ανθρώπους, για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, δεν μιλούμε για απλούς αριθμούς. Οπότε εγώ χαιρετίζω αυτή τη συμφωνία, δεν θα την έλεγα παζάρεμα, αλλά θα πρέπει στην επόμενη συνοδοκορυφή και στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία και ελπίζω τελικά να τα καταφέρουμε. Επίση, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτή τη συμφωνία μια επιταγή ελευκό, γιατί δεν πρόκειται για τέτοια. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία από τη συμφωνία για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Αν δεν κάνουμε τη διάκριση αυτή, θα δεχτούμε και όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Δηλαδή, την ε, παραβίαση της ελευθεροτυπίας, ε, τον περιορισμό των ε, ελευθεριών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά να τα θέσουμε ως όρους στην Τουρκία. Επίσης, θα πρέπει ε, τα επιπλέον 3 δισεκατομμύρια, συνολικά 6 δισεκατομμύρια δηλαδή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα τα χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την Τουρκία, για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος νόμιμος και σωστός τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα θα ήταν αρνητικά και στραβά. Επίσης θα πρέπει να ανακτήσουμε τον πλήρη έλεγχο στα εξωτερικά μας σύνορα. Συμφωνώ λοιπόν με τις αποφάσεις των κρατών μελών και επιτέλους ε, σωστή είναι αυτή η κατεύθυνση να αναζητήσουμε συγκεκριμένη λύση τώρα ως προς την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα μόνη της δεν θα πρέπει να γίνει ένα κλουβί για πρόσφυγες. Θα πρέπει να τη βοηθήσουμε να, ε, να επιλύσει αυτό το πρόβλημα που ε, ε, αντιμετώπισε λόγω της πολιτικής και γεωπολιτικής της θέσης. Ευχαριστώ δυναμία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το προσφυγικό για το οποίο ευθύνη φέρουν και ευρωπαϊκές χώρες όπως και η Τουρκία. Είναι φανερό και ολέθριο το γεγονός ότι η Ευρώπη εκβιάζεται από τις πολιτικές του κυρίου Ερτογά. Εδώ εξελίσσεται ένα φτηνό ανατολίτικο μπαζάρι χείρις της μορφής που στο βωμό των σκοπιμοτήτων θυσιάζονται τα πάντα. Και όλα αυτά προκύπτουν γιατί η Ευρώπη δυστυχώς δεν λειτουργεί στη βάση των αρχών και αξιών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε αλλά στη βάση συμφερόντων. Η κοινοτική αλληλεγγύη προπολού έχει πάει περίπατο και λειτουργεί μόνο το εθνικό συμφέρον. Ορθώνονται φράχτες και εξακολουθούν να χάνονται εκατοντάδες αθώες ψυχές στη θάλασσα αντί να λειτουργήσουν η από αντιμετώπιση του προβλήματος ως οικογένεια για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσει η πολιτική ενοποίηση. η ένωση κινδυνεύει με διάλυση και αυτό έχει επιτρέψει στους ευρωσκεπτικιστές που είναι εντός των τυχών να νιώθουν δικαιωμένοι. οφείλουμε να αποφασίσουμε άμεσα ότι θα γίνονται δεχτοί όσοι πρόσφυγες περνάνε από χερσαίες νόμιμες οδούς έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το απάνθρωπο φαινόμενο της διακίνησης μέσω θαλάσσης με τα θλιβερά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το προσφυγικό δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι και διεθνές πρόβλημα. Και χρειάζεται βεβαίως ευρωπαϊκή λύση, αλλά και διεθνής λύση με βάση αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Την κρίση την καταλάβαμε με χρονική στέρηση. Μας βρήκε απροετοίμαστοι. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε περισσότερη ευρώπη καλύτερη ευρώπη εμβάθυνση και διεύθυνση των δημοκρατικών μας θεσμών πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση. η συμφωνία με την τουρκία είναι σημαντική. δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή. η συμφωνία με την τουρκία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός ανατολίτικου παζαριού. με την τουρκία χρειάζεται μια εταιρική σχέση σε όλους τους τομείς και όχι μια σχέση εξάρτησης από την τουρκία. Τη λύση πρέπει να τη δώσουμε εμείς. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το δίκαιο όμω τη θαλάσση δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα. Και το δίκαιο τη θαλάσση είναι αυτό που επικύρωσαν όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 1982 από τι αποφάσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μόνο η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει το δίκαιο τη θάλασσα. Χρειάζεται επίση να επανέλθουμε στου κανόνε του Σέγγεν τι θα γίνει με τις χώρες του βίζεγκραντ. δεν ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο αρνούνται να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο. χρειάζεται ενίσχυση και έκτακτη ανάγκη εντός της ευρωπαϊκής ένωσης μια πολύ θετική απόφαση πολιτική αλληλεγγύη στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και κυρίως του νότου και την ελλάδα. αλλά και στα δυτικά βαλκάνια δεν τιμά την ευρωπαϊκή ένωση η κατάσταση στην ιδωμένη. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι περιμένουμε τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου στις 17 και 18 μαρτίου. ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως πολύ σωστά είπε η κυρία μέρκελ και ο κύριος juncker. σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Η κυρία Πέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μία εβδομάδα Ακούγαμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ, να προειδοποιεί τους ε, μετανάστες να μην έρθουν στην Ευρώπη. Ε, πραγματικά γύριζαν τα έντερά μου και τώρα καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο αυτών των απειλών. Η ενημπορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει προσφυγική κρίση καταλήγει σε μια συμφωνία που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αντιμετωπίζει του ανθρώπου, τα ανθρώπινα όντα ω εμπορεύματα και χρησιμεύει ε, την Τουρκία ω ένα τεράστιο τείχο προστατευτικό με αντάλλαγμα δισεκατομμύρια ευρώ. Είδαμε φρικτές, φρικαλές εικόνες, παιδιά να πεθαίνουν στις παραλίες, να τα ξεβράζουν τα νερά, γυναίκες να υφίστανται κρυγόνα. Ε, ένα πραγματικό ανθρώπινο δράμα, μια ανθρώπινη τραγωδία. Και ποια είναι η λύση που προτείνουν η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, να τους επιστρέψουμε στην Τουρκία. Τι ντροπή, τι κρίμα. Πραγματικά έχουμε ακόμη καιρό, γιατί έχουμε δείξει πολλέ φορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την βούλησή μα να τροποποιήσουμε αυτή τη λύση. Επιτέλου, σκεφτείτε του ανθρώπου. Σκεφτείτε να επαναφέρετε στην Ευρώπη την ελάχιστη αξιοπρέπεια που τη έχει απομείνει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, Κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης ε, διερωτήθηκα ανθυπομοιδιώντας ότι αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα γινόταν με τους ε, μετανάστες. Θα προσπαθούσαν οι μεμονωμένες χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μόνες τους. Μήπως τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα περιζόντουσαν μόνο στο να ομιλούν αλλά και να διαθέσουν τα εξειδείς. Νομίζω η απάντηση θα ήταν πολύ δυσάρεστη αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν πράγματι προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα όπου καλούμεθα να υποστηρίξουμε κάποιους ε, που έρχονται από άλλες περιοχές. Αναφέρομαι στον κανόνα ένας προς έναν. Ε, έγινε λόγος για αυτόν τον κανόνα και, με πάση περιπτώσει, κάτι είναι και αυτό. Αυτή η λύση ένας προς ένα, πρόσφυγες προφανώς, δεν σημαίνει ότι τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί. Σίγουρα αυτή η λύση δεν είναι ασφαλής, είναι και λίγο επικίνδυνη, αλλά παρόλα αυτά είναι κάποια λύση. Είμαι λοιπόν στις 17 Μαρτίου, παρεμπιπτόνως παρένθεση εδώ, στις 17 Μαρτίου εμεί στην Ιρλανδία έχουμε αργία, είναι εθνική εορτή, κλείνει παρένθεση. Στις 17 λοιπόν Μαρτίου ελπίζω όλοι να εμπνευστούν από τους Ιρλανδούς ήρωες και να βρουν μια καλή λύση. Και πάω τώρα στην αναγκαιότητα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Γιατί δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση, αν τα σύνορά μας ε, είναι κλειστά ε, είτε για περίπτωση πολέμου είτε για οτιδήποτε άλλο. Και τίθεται και το ερώτημα των ποσοστώσεων. Εφόσον τα κράτη-μέλη λένε ότι αυτούς μπορούμε να δεχτούμε και όχι παραπάνω, ε, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με πρακτικό τρόπο, να πούμε, ξέρετε, θέλουμε να βοηθήσουμε. Αυτό τουλάχιστον είναι μια σαφής κατεύθυνση. Και πάλι κλείνω, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πού θα βρισκόμασταν λόγω της κρίσης και εν ώψη της κρίσης. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεστε το χρόνο που έχει προβλεφθεί για τον καθένα από εσά. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ. Η απάντηση που περιμένουμε από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων 17 και 18 Μαρτίου στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι να μα πούν ότι από την Τουρκία εξαρτάται το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει εκείνοι να λάβουν τι ευθύνε του. Και είναι κραυγαλές οι ευθύνε αυτές. Κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί ότι η προσφυγική ροή ε, θα επιληθεί ω διαμαγεία με την επαναφορά των προσφύγων στην, ε, ή την επιστροφή του στην Τουρκία. Και το έδειξε αυτό η σύνοδο κορυφή που αφιερώθηκε στο θέμα αυτό. Το επόμενο ε, Συμβούλιο Κορυφής θα πρέπει να εξακριβώσει και σε τι βαθμό βρίσκεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει να ξεσφίξουμε τον κλειό των πολιτικών λιτότητας για να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δανειστεί εκεί που χρειάζεται για να περιθάλψει, να υποδεχθεί με αξιοπρέπεια τους πρόσφυγες και να επιτρέψει και στις χώρες που το έχουν ανάγκη να στηρίξουν το λαό τους μετά από χρόνια λιτότητας και αυτό να το κάνουν υπό συγκεκριμένε ε, προϋποθέσεις και με κατάλληλους όρους. Γι' αυτό το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής θα έχει και οικονομικό χαρακτήρα αλλά θα αποτελεί και έκκληση προς την αλληλεγγύη. Κάτι που προϋποθέτει μια ικανότητα πιθανότητα δανεισμού για να χρηματοδοτηθεί αυτή η αλληλεγγύη. Ο κύριος Χριστοφόρου. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους λαούς οφείλει να μιλήσει ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές και χωρίς ακαταλαβίστικες θεωρίες και χωρίς αυθυσιμίες τόσο για το προσφυγικό όσο και για την Τουρκία. Πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι το προσφυγικό δεν είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό μόνο θέμα δεν είναι μόνο ζήτημα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα διεθνές ζήτημα που οφείλουν και οι υπόλοιπε χώρες διεθνώς να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια για επίλυσή του. Για όσου εργολάβους της καταστροφολογίας και του ευρωσκεπτικισμού θέλουν και θεωρούν ότι με το προσφυγό μπορεί να ενταφιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι πεπισμένος ότι και για αυτό το ζήτημα η Ευρώπη μπορεί να βρει λύσει. Για την Τουρκία, τι έκανε σε όλη αυτή τη διαδρομή για το προσφυγικό η Τουρκία. Να θυμίσω ότι η Τουρκία ήταν μέρο του προβλήματο γιατί με τη στάση και τη συμπεριφορά και την πολιτική τη στην περιοχή δημιούργησε το προσφύγιο. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη συμφωνία για να περιορίσει τι ροέ προ την Ελλάδα όχι μόνο δεν τη σεβάστηκε αλλά αύξησε τι ροέ. Και να θυμίσω τώρα ότι μια χώρα που είναι υπό ένταξη και μάλιστα θέλει να επιταχύνει τι διαδικασίε ένταξη συμπεριφέρεται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ομό κοινικό εκβιαστή βάζοντας μπροστά το ανθρωπιστικό ζήτημα και χρησιμοποιώντας το ζόρι για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα και να πάρει ανταλλάγματα. Πρέπει να θυμίσω και πάλι ότι σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί η Τουρκία σήμερα να ζητά το άνοιγμα των κεφαλαίων για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία όταν όλες οι χώρες γνωρίζουν τις αρχές, τις αξίες αλλά και τη διαδικασία που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει το Συμβούλιο να μην ξαναδεχθεί να τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων θέμα ανοίγματο του κεφαλαίου τη Τουρκία εάν δεν υλοποιήσει τι συμφωνίε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωτόκολλο τη Άγκυρα και αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προ την Τουρκία και οφείλει να ουσιαστεί μέχρι τέλου. Η συνάντηση κορυφή τη Δευτέρα κατέδειξε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και νομίζω ότι στις 17-18 Μαρτίου ε, θα ληφθούν οι αποφάσεις για το διατάφτα. Βεβαίως και πρέπει να βοηθήσουμε την Τουρκία, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Σήμερα πλέον δεν υπάρχει πολιτικό θάρρος και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε κράτη τα οποία με απόλυτο εγωισμό επιθυμούν να επιβάλλουν τα δικά τους τα συμφέροντα χωρίς να σκέπτονται καν την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αδύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αλλά ξέρετε με τον τρόπο αυτό ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε κοινή λύση. Η λύση είναι μία, δηλαδή να επιμεριστεί το βάρος με δίκαιο τρόπο και στα 28 κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας να προσπαθεί μόνος του να κάνει ότι του καπνίσει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Κέλλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, η Σύνοδος Κορυφής ε, της Δευτέρας ε, διάλεξε την καλύτερη λύση μεταξύ των σχετικά κακών ε, προτάσεων. Ε, θέλει να ανακτήσει τον έλεγχο και να δείξει στους λαθρο, ε, ε, τι συμβαίνει. Επίσης, ε, πολλές φορές οι λαθροδιακινητές συνεργάζονται με τους τρομοκράτες. Αφού προσπαθήσουμε να ανεχιετήσουμε, αλλά δεν αρκούν αυτά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους της Συρίας. Και αυτό ήταν πολύ καλοδεχούμενο το μήνυμα που μας ε, υπενηχθήκατε σήμερα και δεν το δηλώσετε ρητά κυρία Υπουργέ. Επίσης, ε, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και προστασία τους. Αυτό εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να μην παραμείνει στα λόγια, αλλά να περάσει και στα έργα. Ε, οπότε χρειαζόμαστε συνεργασία και χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορέσουμε από κοινού να διαφυλάξουμε και τα βορειοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είχαμε το φιλανδικό παράδειγμα και η Ρωσία ίσως αποπειραθεί να αποσταθεροποιήσει από, απρόβλεπτη, από απρόβλεπτο σημείο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η προκάτοχός σας, κυρία Υπουργέ, είχε υποσχεθεί ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα το είχε ολοκληρώσει και το έκανε για τα δεδομένα. Επίσης, ελπίζουμε να διεκπαιρεωθεί αυτό το θέμα στην Ολλανδική Προεδρία και όλα τα πρακτικά μέτρα και τα μέτρα εφαρμογής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν μέχρι το καλοκαίρι αν το Συμβούλιο δεν λάβει μια απόφαση. Και μάλιστα και εμείς ε, έχουμε κολλήσει και δεν μπορούμε να λάβουμε την κατεπίγουσα αυτή απόφαση, γιατί μερικά, μερικές πολιτικές ομάδες καθυστερούν σε ό,τι αφορά την οριστικοποίηση του πακέτου. Ε, επισπεύστε παρακαλώ τα πράγματα. Κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Τούσκ είπε ότι η παράτυπη μετανάστευση, η λαθρομετανάστευση θα τελειώσει. Η συμφωνία με την Τουρκία όμως δεν θα περιορίσει τελικά τις μεταναστευτικές ροές. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του Συμβουλίου στις 17 και τις 18, αλλά μεταξύ, πολλοί υποφέρουν. Πολλοί πρόσφυγες λιώνουν μπροστά σε κλειστέ πόρτε. Η πολιτική που ακολουθούμε δεν είναι παραγωγική. Το σύστημα ένας εναντί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Ποιες είναι οι εγγυήσεις που μας δίδονται ότι η Τουρκία θα μειώσει τις μεταναστευτικές πιέσεις. Όταν στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υφίσταται μια παράλληλη οικονομία δικτύων διακινητών. Επιτέλους, έχουμε κάποιες καλύτερα μαντάτα από το προσφυγικό μέτωπο και από το οικονομικό. Γιατί είχαμε την αίσθηση της ανήμπορης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και μερικές φορές αυτό έπαιξε το παιχνίδι των λαϊκιστικών τάσεων. Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης έγινε θύμα κακών αποφάσεων γιατί αναγκαστικά αρχικά είχαμε τα προβλήματα στα ανατολικά σύνορα, μετά αδιαφορήσαμε για τα αρνητικά μηνύματα από, από τη Μεσόγειο με τη Μάλτα και τη Λαπεντούζα και μετά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο λαθρεμπόριο ανθρώπινων όντων αν προηγουμένω για τον 21ο αιώνα. Επίσης είχαμε ε, σύρους σε καταβλισμούς προσφύγων στο, στην Τουρκία, Λίβανο και Ορδανία. Επιτέλους θέλουμε κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και απάντηση ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσφυγική κρίση. Ε, δύσκολη θα είναι η συνεργασία με την Τουρκία, το είπαμε, αλλά είναι απαραίτητη, γι' αυτό θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί επίσης η βοήθεια προς την Ελλάδα, να συγκεκριμενοποιηθεί και να λύσουμε τα προβλήματα στη Συρία, αυτή είναι η πηγή των προβλημάτων. Ο Τούσκ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, είπε ότι τελειώνουν οι μέρες της ε, λαθρομετανάστευσης στην Ευρώπη. Μακάρι να έχει δίκιο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται σε κρίση. Το ίδιο και όλη η Ευρώπη. Εδώ και 3,5 ώρες συζητούμε τη συνοκορυφή της Δευτέρας όπου κανείς μας δεν ήταν παρόν, ούτε καν ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ούτε ο Προεδρεύων. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κρίνουμε τι πραγματικά έγινε στην συνοκορυφή γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Ίσως καλύτερα να διαβάζουμε το, το πολίτικο, την εφημερίδα αυτή. Βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες από ό,τι ακούμε εμείς εδώ στην ενημέρωση που μας γίνεται. Θα έπρεπε τουλάχιστον ο κ. Γιούνκερ να είναι εδώ σήμερα. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στη συνοκορυφή. Όλοι λένε ότι βρισκόμαστε ενώπιον τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αλήθεια, πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα. Κυρία Βαλενθιάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι λυπηρή η απουσία του Πρόεδρου Τούσκ και του Πρόεδρου Γιούνκερ σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Λυπηρή. Πολλοί από εμά, μάλιστα, Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβαίνει τις αρχές της ε, και τις ευθύνες της. Η Προκαταρκτική Συμφωνία για την οποία ενημερωθήκαμε έμεσα, όχι μέσω της, ε, των πληροφοριών μας στο Συμβούλιο, ε, είναι αμφισβητούμενης νομιμότητας, αποτελεσματικότητας και ηθικής. Πέστε στον πρόεδρο Τούσκ ότι είναι απαράδεκτο σε αυτό το κείμενο να μην αναφέρεται ούτε μία αφορά η, ε, η, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς είναι να τους ξέφυγε αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αποκλειστικά σήμερα είναι το Συμβούλιο, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να ακούσουν τις φωνές αυτών που πραγματικά σκέφτονται τους υπόλοιπους. Υπάρχει μια διαφορετική Ευρώπη. Ευρώπη διαφορετική από αυτήν που εσείς κατασκευάζετε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Ο κύριο Σοχίνιο. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχε ω επίκεντρο τις ε, μεταναστευτικέ ροέ και τι προτεραιότητε για την απασχόληση ε, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, είναι σημαντικό να μην κάνουμε λάθο στη διάγνωση. Και η διάγνωση είναι σαφέστατη. Δεν ήταν ε, οι μεταναστευτικέ ροέ που προκάλεσαν την ευρωπαϊκή κρίση. Ήταν η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανεμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέτρεψε ένα πρόβλημα διαχειρίσιμο με αλληλεγγύη και συνεργασία σε, ένα... σε μια σοβαρότητα κρίση ταυτότητας ε, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει στις χώρες τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Αυτές ε, οι συστάσεις, ιδιαίτερα για τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι ενέργειες ε, μερικές φορές αλόκοτε και αεροπρόσωλες, ε, γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους ασύμμετρους κραδασμούς. Γιατί από τη μια μα ζητά να επενδύσουμε στην παιδεία, στην επαγγελματική κατάρτιση έρευνα, στην αναβάθμιση αλυσίδα αξιών, στην απασχόληση και να καταπολεμήσουμε τι μακροοικονομικέ ισορροπίε. Και από τι άλλε μα ζητούν να περικόψουμε τυφλά τι βασικέ και κεντρικέ λειτουργίε του κράτου. Θέλουμε ένα, μια νέα όθηση στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Όραμα και ηγεσία. Ε, θέλουμε να σταθούν επιτέλου για μια φορά στο ύψο των προκλήσεων οι ηγέτε μα. Ο κύριο Σαντ. Ελπίζουμε ότι η συμφωνία αυτή θα γίνει, η προκαταρχή συμφωνία θα γίνει μια πραγματική τελική οριστική συμφωνία. Δεν βλέπω καλύτερη λύση. Θα πρέπει όμω να αναγνωρίζουμε τι πραγματικότητε. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, διαφορετικά συμφέροντα ασύμετρα και αντιβαίνοντα πολλέ φορέ. Και στη Συρία και στο προσφυγικό. Ε, επικρατεί μια κάποια ασάφεια, η οποία είναι ε, επικίνδυνη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλει να ελέγξει τις ροές ε, των προσφύγων και θα δώσει χρήματα γι' αυτό. Η Τουρκία από την άλλη μεριά θέλει να προχωρήσει η αίτησή της για ένταξη. Όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια πλειοψηφία εναντίον τη εισόδου. Εγώ είμαι στη μειοψηφία βέβαια. Απ' την άλλη μεριά η Ευρώπη κατακρίνει την Τουρκία για την αυταρχικότητά τη και τον τρόπο που αντιμετωπίζει του Κούρδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαιρεμένη. Η Τουρκία είναι ενωμένη. Η καλύτερη λύση θα ήταν να πούμε τα πράγματα με το όνομά του βέβαια και να βρούμε ένα τρόπο να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίτσουλα, μετά από έξι χρόνια πόλεμο στη Συρία δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το δράμα. Ε, έχουμε τώρα επιτέλους συγκεκριμένε προτάσεις γιατί έχουμε ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο. Μερικά είναι πολύ θετικά. Κυρίως θα πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση της ανθρώπινης οδύνης και της ανθρώπινης απελπισίας. Δεν θα πρέπει όμως να κάνουμε χειραγώγηση της ανθρωπιστικής καταστροφής για ιδιαίτερα κρατικά συμφέροντα. Θα πρέπει να μην εθελοτυφλούμε σε ό,τι αφορά την καταστρατήγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Επίσης, ε, η διατύπωση που υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο. Επίσημα έχει κλείσει η Βαλκανική οδός, υποτίθεται. Αλλά εξακολουθούν να μένουν μπλοκαρισμένοι, εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα σύνορα Ελλάδας-Μακεδονίας. Και τα σύνορα αυτά υφίστανται τεράστιες πιέσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ε, και τα, τις χώρες που είναι εκτός ε, της ζώνης ε, Σέγγι και παρόλα αυτά ορθώνουν σειρματοπλέγματα με ξηράφια στη, στα σύνορα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Νίνα Τζιλ. Άλλη μια σύνοδος κορυφής και πάλι δεν είμαστε κοντά στο να λύσουμε το προσφυγικό. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αντί να κοιτάμε τα προβλήματα μόνο των συνοριακών κρατών όπως η Ελλάδα, μεταφέρουμε το πρόβλημα στην Τουρκία και τι τίμημα πληρώνουμε. Όχι σε ευρώ, αλλά εξαιτία του ότι παραβιάζουμε τις αρχές μας. Κλείνουμε τα μάτια στην καταπίεση της, ε, του τύπου και στην παραβίαση των ελευθερών έκφρασης στην Τουρκία. Και ξεχνάμε ότι ο τουρκικός στρατός τιμωρεί συλλογικά τον πληθυσμό στην Ανατολική Τουρκία. Ε, χρειάζεται να ανακοχή ανάμεσα στο ΠΚΚ και τον τουρκικό στρατό αμέσως. Να, το να προσφέρουμε επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους θα πλήξει την αξιοπιστία μας σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αξιοπιστία επέτρεψε στη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μεγάλα βήματα στο, στο κράτος δικαίου στη γειτονιά μας. Ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι στην αντιμετώπιση της προσφυγικής τραγωδίας αυθονούν μέχρι τώρα τα ωραία λόγια που διαψεύδονται όμως από τις πράξεις. Είναι φανερό ότι μια ικανοποιητική λύση πρέπει να περιλαμβάνει και μια συνεργάσιμη Τουρκία. Σε αντίθεση όμως με την Ελλάδα που τηρεί τις δεσμεύσεις της, η Τουρκία δεν εφάρμοσε την υπάρχουσα συμφωνία και προβάλλει διαρκώς και νέες απαιτήσεις σε ένα ανατολίτικο παζάρι διαπραγματεύσεων μόνο που το παζάρι αυτό αφορά ψυχές και ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς πρέπει λοιπόν να απαντήσει η Ευρώπη αν θέλει να παραμείνει ενωμένη και σύμφωνη με τις εμελιώδεις αξίες της πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλάβει τις δικές της ευθύνες απέναντι στους πρόσφυγες και τις περιοχές που δοκιμάζονται δυσανάλογα όπως είναι τα ελληνικά νησιά πρέπει τέλος να επιμείνει ότι η συνεργασία της τουρκίας στο προσφυγικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ένταξης και όχι προς θεού το κλειδί που θα της ανοίξει διάπλατα την πόρτα. θέλω σήμερα να θυμηθούμε τη φράση του Ζων πολ Σάρτ. εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μάτια μας για να βλέπουμε τότε θα τα χρειαστούμε για να κλάψουμε. Η κυρία Πόστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μέρκελ εχθές ε, είπε ότι ήταν μια πολύ καλή ημέρα γιατί υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις με τον κύριο Ερντογάν. Ίσως ε, αυτό ε, να μην ίσχυε καταλέξει. Περισσότερο ήταν μια καλή μέρα για τους ε, Τούρκους ε, διαπραγματευτές. Ήταν μια καλή μέρα για τους διακινητές. Ένας προς έναν είπαν θα τους ανταλλάσσουν. Θα έρχονται δέκα και θα πηγαίνουν δέκα Σύριοι από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Κάπως έτσι. Δεν θα είναι βέβαια ίδιοι άνθρωποι. Αυτό είναι κατ' ουσίαν σκλαβεμπόριο, εμπόριο σκλαβιάς. Και από ό,τι φαίνεται η κυρία Μέρκελ αλλά ούτε και ο κύριος Ρούιτε θα μπορέσουν να περάσουν αυτή την πρόταση. Ο κύριος Όρμπαν ήδη απείλησε ότι θα καταθέσει βέτο. Το χειρότερο βέβαια είναι ε, ότι μπορεί να υπάρξει και καμία απολύτως λύση. Εχθές δεν ήταν καλή ημέρα. Στη δική μου την Ευρώπη δράκανης με σοφία, με υπευθυνότητα και όχι όπως ο κύριος Ο κύριος Ανδρουλάκης στην αίθουσα του κοινοβουλίου όπω και στο συμβούλιο υπάρχουν εκπρόσωποι λαών που φαίνεται ότι ξέχασαν την ιστορία του και το γεγονό ότι ήταν πρωταγωνιστέ τεράστιων προσφυγικών ροών για δεκαετίε. εάν επίση δεν θυμούνται πώ δημιούργηκε το κοινό ευρωπαϊκό όραμα και το μόνο που του ενδιαφέρει είναι τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να τα ξεχάσουν και αυτά όσο δεν εφαρμόζουν τι κοινέ αποφάσει για τη μετεγκατάσταση. επίση κάποιοι άλλοι δεν βλέπουν ότι η συμφωνία με την τουρκία είναι ανεφάρμοστη παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και προκαλεί όταν αποκρύπτει τον πραγματικό ρόλο του κύριου ερντογάν τόσο στην αστάθεια της συρίας όσο και στην καταβαράθρωση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ίδια την τουρκία. όσο αυτό το τραγικό έργο συνεχίζεται το πρώτο θύμα θα είναι οι πρόσφυγες και το δεύτερο ο ηθικός νομικός και πολιτικός πολιτισμός της ευρώπης. ως έλληνας το μόνο παρήγορο που μπορώ να σημειώσω είναι ότι ένας λαός που ζει σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία με πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας αποδεικνύει σε συντριπτικό ποσοστό ότι η αλληλεγγύη δεν είναι la και δεν είναι μόνο χρήσιμη όταν τη δέχεσαι αλλά πάνω απ' όλα είναι λυτρωτική όταν την προσφέρεις. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεστε το χρόνο που προβλέπετε για σας. Ε, Ζωηντρόβα παρακαλώ. Πίτροπε, ε, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που ακούω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περι, αναμένει φέτος μία μικρή μόνο αύξηση στον αριθμό των προσφύγων. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα για να φέρουν αυτή την ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ε, δεν είναι η μόνη λύση ούτε το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να δράσουμε στη Μέση Ανατολή, χρειάζεται να προστατέψουμε τα εξωτερικά μας σύνορα Και στην κατανομή των 3 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη... Ε, και στη χρήση τους ε, θα πρέπει να έχουμε έλεγχο του, του θα είναι οι παραλήπτες. Το σύστημα του ένας εναντίον ενός είναι ένας τρόπος να σταματήσουμε την παραμεταναστεύση. Γιάννα Γκόμες. Ε, η Τουρκία θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της λύσης, αλλά <laughs> κυρίως είναι τμήμα του προβλήματος. Ε, όχι μόνο γιατί διατηρεί τα κυκλώματα ε, διακινητών, αλλά γιατί δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στο Ιράκ, Συρία και στην Ανατολική Ασία. Ε, το Συμβούλιο τα ξέχασε όλα αυτά ε, και υπέκυψε σε αυτό τον ε, εκβιασμό του Ερντοάν νομίζοντας ότι μπορεί να εξάγει τις ε, δικές μας ε, υποχρεώσεις, δικές υποχρεώσεις στην Τουρκία, διευκολύνοντας την Τουρκία με τις ε, θεωρήσεις και κλείνοντας τα μάτια στις παραβιάσεις των κριτηρίων της Κοπενχάγης και του καταπίεσης του δικού του λαού πλευράς του κ. Ερντοάν, επίσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των Τούρκων Κούρδων, όπως επίσης και των Κούρδων στη Συρία, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται πολύ θαραλέα εναντίον του Ισλαμικού στρατού. Το Συμβούλιο με, την, με τις πολιτικές επιστροφής τους και με το σύστημα ένα προς ένα εναντίον ενός είναι κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπρόθεση. Και τώρα το Κοινοβούλιο πώ τολμούν να μιλούν για τα Το Συμβούλιο και, το... και η Κομισιόν πώ μπορούν να μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, όταν. Ε, ε, η μεταχείριση που ε, δίδουμε προς τους πρόσφυγες είναι πραγματικά απάνθρωπη. Ευχαριστώ. Κυρία, Κυρία Ευχαριστώ. Από την πρώτη μέρα της παρούσας ε, μεταναστευτικής κρίσης λέω ότι το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε στην πηγή του, στη Συρία, στο Ιράκ και να μεριμνήσουμε για τους πρόσφυγες σε συμφωνία με τους διεθνείς εταίρους μας από την περιοχή. Η παρούσα συμφωνία με την Τουρκία θα ήταν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αν επρόκειτο για αξιόπιστο εταίρο. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις υπηρεσίες της Τουρκίας ε, που περιέθαλψε τεράστιο αριθμό σύρων προσφύγων. Αλλά είναι πλέον σαφές ότι εδώ και καιρό η Άγκυρα χρησιμοποιεί ε, και ε, εκμεταλλεύεται αυτή την κρίση για να κάνει πολιτικούς εκβιασμούς και να υλοποιήσει τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Τα προβλήματα που βιώνει η Ευρώπη εξαιτία μεταναστευτική κρίση δεν είναι αμεληταία και θα γίνουν όλο και οξύτερα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από του Ρώσου και του Αμερικάνου να, λύσουν, ή να έχουν κίνητρα ή να δείξουν ενθουσιασμό για να επιλύσουν τα προβλήματα όπως εμεί. Ε, θεωρώ ότι ήρθε ο καιρό να δείξουν οι ευρωπαϊκέ χώρε ότι με συντονισμό μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ε, επίλυση τη ε, κρίση στην Μέση Ανατολή. Ο κύριο Ε, θεωρείται η συμφωνία αυτή ως αρχή της επίλυσης του προβλήματος. Καλύτερα βέβαια συμφωνία παρά αναρχία. Η αναρχία της οποίας γίναμε μάρτυρες του τελευταίους μήνες για να μην πω και χρόνια. Γνωρίζουμε ε, τι συνέβαινε στη Βαλκανική Οδό. Είδαμε τις συμπεριφορές σε αυτή τη Βαλκανική Οδό. Είδαμε ότι μερικές χώρες που δεν έκανε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα η Μακεδονία και η Σερβία, έκαναν πολύ περισσότερα από ό,τι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε πως κάποιες χώρες ε, έβαλαν σειρματοπλέγματα ε, και φράχτες. Και θα πρέπει επιτέλους να επηρεάσουμε αυτή την κατάσταση και πιστεύω ότι αυτά τα σύρματοπλέγματα θα αρθούν αν κλείσει επιτέλους η Βαλκανική οδό. Γιατί ήταν ντροπή αυτό που ε, συνέβη τους τελευταίους μήνες. Επίσης, τα σύνορα Κροατίας-Σλοβενίας, ε, θα πρέπει να, να αρθούν αυτά τα σύρματοπλέγματα. Είναι δραματική κατάσταση και στα ε, ελληνομακεδονικά σύνορα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και την Ελλάδα, να βοηθήσουμε και τη Μακεδονία, λέει ο μιλήτης η κυρία Σένερα Ροντρίγκε. Η κυρία Σένερα Ροντρίγκε. Σένερα Ροντρίγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Γεωργίας, όταν θα μιλήσετε για την απασχόληση, θυμηθείτε και την κρίση του ευρωπαϊκού γεωργικού κλάδου. Μάλιστα, η κρίση αυτή τη στιγμή έχει πλήξει ε, κυρίως ε, το τομέα των απορροκυπευτικών, του χειρίου κρέατος και το γαλακτοκομικό τομέα. Η ανικανότητα του επιτρέπου Χόγκαν ε, να, να ε, προτείνει λύσεις στην γαλακτοκομική κρίση στην Ευρώπη δείχνει κατάφορα την αποτυχία των πολιτικών σας. Σας θέρμο παρακαλώ στο επόμενο Συμβούλιο επιστρέψτε στην πραγματικότητα, προσγειωθείτε και ανοίξτε τους δρόμους στη ρύθμιση της παραγωγής στο γαλακτοκομικό τομέα. Κάτι που σημαίνει ότι θα σταματήσει επιτέλους η καταστροφή των θέσεων απασχόλησης γιατί δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνο για δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση, αλλά να αποφύγουμε την καταστροφή των ε, υφισταμένων θέσεων απασχόληση. Λάβετε υπόψη την κατάσταση του γεωργικού ε, κλάδου. Αφήστε επιτέλους, ε, σταματήστε αυτή την αφέμαξη και σώστε το γεωργικό τομέα. Ο κ. Μαραγκάλ, η Τουρκία σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα το οποίο μας ενώνει εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, Ευρώπη δεν μπορεί να είναι το άθροισμα των εθνικών συμφερόντων. Ποιο εκπροσωπεί την Ευρώπη εδώ, Το Συμβούλιο σίγουρα όχι. Το σημερινό Συμβούλιο είναι διακυβερνητικό έχει ξεχάσει τις ευρωπαϊκές αρχές. ένα αστυνομικό κράτος, η Τουρκία, ε, παίρνει χρήματα από εμά ε, για να μπορέσουμε εμείς ε, να παραβιάσουμε τις δικές μας αρχές. και τιμωρούμε την Ελλάδα, την καταδικάζουμε να γίνει μια φυλακή, γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους βαλκανικούς τείχους που σηκώσαμε. Την Ευρώπη την εκπροσωπεί το κοινοβούλιο μας. Εδώ έχουμε ένα κράτος μέλος, 21, το που ονομάζεται Ευρώπη. Θα χρησιμοποιήσουμε το βέτο μας. Θα αποφύγουμε την αυτοκτονία της Ευρώπης. Θα αποφύγουμε να επιστρέψουμε στην Ευρώπη της δεκαετία του 1930. Οι αποφάσει λαμβάνονται αλλού, το ξέρουμε. Αλλά εμείς θα τις ανακτήσουμε μαζί με τους ε, πολίτες μας γιατί η Ευρώπη θα γίνει φιλόξενη όπως ήταν. Ε, όπως αυτή που θέλετε να διαλύσετε. Ευχαριστώ. Ο λόγο στον Επίτροπο Χάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ ζωντανή συζήτηση, κυρίως όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Και εγώ θα συμφωνήσω με εκείνους που είπαν ότι πράγματι χρειαζόμαστε κάτι. Χρειαζόμαστε πολιτική λύση στη Συρία, χρειαζόμαστε ε, μια ε, παγκόσμια λύση για τις μεταναστευτικές ροές, αλλά επίσης και μια διαρκή λύση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων μας. Πρέπει όμω να είμαστε και πραγματιστές. Χρειαζόμαστε και μια βραχυπρόθεσμη λύση που σημαίνει ότι οφείλουμε να βρούμε μια κάποια συμφωνία με την Τουρκία. Ε, νομίζω ότι Δευτέρα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας και ήταν και μία ημέρα που κατέδειξε ότι ε, η λύση μπορεί να είναι μόνο ευρωπαϊκή περιλαμβάνοντας όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η λύση λοιπόν ε, πρέπει να την υποβάλουν και να την εφαρμόσουν όλοι το να προσπαθεί κανείς μόνος του αυτό δεν βοηθάει, αυτό πρέπει να είναι σαφές και νομίζω αυτό φάνηκε και τη Δευτέρα. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε κάποια θεμελιώδη θέματα που ετέθησαν τόσο όσον αφορά το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των θεωρήσεων όσο και το ενδεχόμενο της επιτάχυνσης ε, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Μπορώ λοιπόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας διαβεβαιώσω ότι κάτι τέτοιο ποτέ δεν θα γίνει εις βάρος της στήρησης των προδιαγραφών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας της ε, δικαιοσύνης. Ε, θα κριθεί ποιος μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όποιος θέλει να μπει στην Ένωση πρέπει να δέχεται τους δικούς μας τους ε, κανόνες. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι κάνουμε, ψωνίζουμε σαν να είμαστε σε σούπερ μάρκετ και λέμε «Α, θέλετε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδική τιμή για σας». Δεν πάει έτσι. Πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Κατά τα άλλα, η απελευθέρωση των θεωρήσεων που δεν το θίγουν πάρα πολύ, αυτή είναι και μέρος ε, της ε, συμφωνίας επανεισδοχής που σημαίνει ότι η Τουρκία θα δέχεται μετανάστες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί άσυλο. Άρα δηλαδή εδώ επιτύχαμε πρόοδο προς όφελος της Ευρώπης. Τώρα όσον αφορά στα 3 ή στα 6 δις ευρώ. Κοιτάξτε, πραγματικά κουράστηκα. Κουράστηκα ε, να λένε οι Τούρκοι ότι δεν του στείλαμε ούτε ένα σέντ. Ούτε σέντ, μα ούτε ένα σέντ δεν του στείλουμε γιατί εμεί τα χειριζόμαστε και τα διαχειριζόμαστε τα λεφτά. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν λένε αλήθεια, όχι μόνο του στείλαμε αλλά και τα στείλαμε μετρητής. Εγώ προσωπικά πήγα στην ε, Δυτική Ανατολία, στο Ταζιαντέπε και σε κάποιες άλλες πόλεις και πρέπει να σας πω ότι στην τουρκική κυβέρνηση και στους διεθνείς οργανισμούς ε, υποκλίνομαι για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται οι πρόσφυγες σε καταβλισμούς όπου έχουν στη διάθεσή τους τα πάντα. Σούπερ μάρκετ, σχολεία, γυμνάσια Μιλάμε για 3.800 σκηνές, 80.000 κατοίκους αυτών των σκηνών, οι οποίοι όμως ε, ζουν εντάξει και πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα 40 δις ευρώ, εμείς διασφαλίσαμε για 6 μήνες 300.000 πρόσφυγες να μπορούν να έχουν σωστή περίταλψη. Με 55 εκατομμύρια ευρώ μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε 300.000 νέοι και παιδιά να μπορούν να επισκεφτούν το σχολείο ολόκληρο το χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι με σχετικά μερικά λίγα κονδύλια μπορέσαμε να διασφαλίσουμε οι άνθρωποι επιτόπου να έχουν ασφαλείς εστίες. Και θέλω επίσης να σας πω ότι συζήτησα με πάρα πολλούς πρόσφυγες στην Ανατολική Ανατολία και αυτοί θέλουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στη Συρία. Δεν θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Πρώτον να αναζητήσουμε πολιτική λύση αλλά και δεύτερον να διασφαλίσουμε εκεί όπου βρίσκονται προς το παρόν να βιώνουν με αξιοπρεπείς συνθήκες ε, και κυρίως οι νέοι και ε, τα παιδιά να έχουν μια προοπτική, να εκπαιδεύονται, να επισκέπτονται τα σχολεία. Στην επίσκεψή μου λοιπόν είδα επιτόπου ότι πρέπει και να ασχοληθούμε με την πρόθεση ε, οικονομικών δραστηριοτήτων για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και να μπορούν οι πρόσφυγε να εργαστούν. Κοιτάξτε κυρίε και κύριοι, η Δευτέρα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Είναι απόλυτα σαφέ ότι ο κύριο Τούσκ έχει το καθήκον να φέρει εις πέρα στις διαπραγματεύσεις και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει υπό το πνεύμα της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και τελικά και της ομόφωνης εφαρμογής εκ των υστέρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας παρακαλώ να παραμείνετε στη θέση σας και παρακαλώ και να παραμείνετε ήρεμοι. Το λόγο έχει η εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Όπως είπα νωρίτερα σήμερα το πρωί, χρειάζεται περισσότερη δουλειά με την Τουρκία. Και για αυτό το λόγο ο πρόεδρος Τούσκ ε, θα επεξεργαστεί τις ε, προτάσεις ε, και θα συζητήσει τις λεπτομέρειες με την Τουρκία μέχρι το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Συνεπώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις με λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Αλλά αναμφίβολα οι ηγέτες μας ανέφεραν ρητά στη δήλωσή τους ότι η τελική συμφωνία θα σεβαστεί το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Και συμφωνώ με τον κύριο Βέμπερ. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την Τουρκία και όχι σε εξάρτηση από την Τουρκία. Α είμαστε σαφεί. Στόχο δεν είναι να, σταματήσουμε του πρόσφυγε από τον έρχονται. Θέλουμε να περάσουμε από την παράτυπη μετανάστευση σε μια ελεγχόμενη μετανάστευση. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα και δεν ξεπουλάμε τις αρχές μας. Επιταχύνουμε, αλλά δεν συμβιβαζόμαστε σε ό,τι αφορά την ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ε, η αιρεσιμότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Το ίδιο ισχύει και για τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων ένταξης. Οπότε η διεύρυνση και η απελευθέρωση των θεωρήσεων έχουν ε, προϋποθέσεις. Δεν χαμηλώνουμε τον πύχη. Ό,τι συμφωνήσουμε με την Τουρκία οπωσδήποτε θα σέβεται τον το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Η δήλωση της 7 Η Μαρτίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το λέει ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να βραχικυκλώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να προγραμμίσω το εξής. Ε, η, α, η πρέπει να διατηρήσουμε την ηθική μας. Ασφαλώς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την τελειότητα. Και η Συμφωνία Επανεισδοχής ε, και μέσω της Συμφωνία επανεισδοχη Ελλάδα Τουρκία και μέσω της συμφωνία επανεισδοχη Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκία, η Τουρκία θα πρέπει να δεχθεί όλους τους επιστρεφόμενου μετανάστες που πέρασαν από το έδαφό τη. Αν επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες που ξεκίνησαν ήδη γιατί πάνω από 300 μετανάστες ήδη επεστράφησαν από την Ελλάδα στην Τουρκία, τότε ε, θα θεωρήσουμε ότι τηρεί τις διεθνείς υποσχέσεις ε, όπως η αρχή της μη επαναπρόθεσης και αυτή τη στιγμή πάνω, από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες ε, χαίρουν προστασία στην ίδια την Τουρκία. Τέλος. Αυτοί που αναφέρονται στη Σύμβαση της Γενέβης καταλα... Ε, ε, έχουν δίκιο να ανησυχούν. Αλλά όπως σας είπα δεν θα υποχωρήσουμε έναντι των, εθνικών μας, των ε, ηθικών μας νομικών μας υποχρεώσεων. δεν θα κάνουμε παρεδόσε. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η σημερινή κατάσταση στην οποία κάποιοι άνθρωποι μέσα σε βάρκες κάνουν επικίνδυνο ταξίδι δεν συμβιβάζει ζέτε με το δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η σημερινή κατάσταση δεν ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα δίκτυα παράνομων διακινητών. Αυτή είναι η, εθνική μας, ε, ε, ηθική μας υποχρέωση. Και ο κ. Καμάλ έχει δίκιο. Η πραγματική μας εχθροί δεν είναι οι πρόσφυγες. Ε, οι διακινητές είναι οι πραγματικοί μας εχθροί. Πρέπει να τελειώσω, διότι γίνεται, είναι πολύ θόρυβος μέσα στην αίθουσα. Να πω δύο λόγια για τη Ζαμάν, για την εφημερίδα η οποία τέθησε αναγκαστική διαχείριση. Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας ξεκάθαρα ε, στον Τούρκο Πρωθυπουργό. Και η κυρία Μέρκελ και ο δικός μου πρωθυπουργό συναντήθηκαν την Κυριακή με τον ε, κύριο Νταβούτογλου ε, και το ανέφεραν και τη Δευτέρα το ίδιο. Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν είναι διαπραγματεύσιμα αγαθά. Οπότε η Τουρκία θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση. Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια, δεν πρόκειται να φλήσουμε. Τώρα, για να απαντήσω στην κυρία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου θυμήσατε τις ε, δηλώσεις μου πριν από αρκετά χρόνια. Εξακολουθώ να τις στηρίζω. Ε, νομίζω ότι ήταν οραματικές, βλέποντας τις από, τη σημερινή συγκυρία. Θα ε, ζητώ ευρωπαϊκές λύσεις και θα συνεχίσω να ζητώ ευρωπαϊκές λύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Πριν από την ψηφοφορία θα έχουμε μία ανακοίνωση του Προέδρου κυρίου Σούλτς.